Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Συνεχίζουμε τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακόπησε στις 10 Οκτωβρίου. Τα πρακτικά, τα κείμενα έχουν εγκριθεί τη συνεδρία 9 και 10 Οκτωβρίου. Έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά, υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε τα πρακτικά θεωρούνται συγκεκριμένα. Κάποιες ανακοινώσεις να ενημερώσω την Ολομέλεια ότι δεν μου ήρθε κανένα αίτημα να ψηφίσουμε τα διορθωτικά σύμφωνα με το 241 παράγραφος 4 του κανονισμού που ανακοινώθηκε στις 9 Οκτωβρίου. Τέτοιες διορθώσεις θεωρούνται ως εγκεκριμένες όσον αφορά την κοινή θέση για την παράταση του Περιφερειακού Ταμείου της Ευρωπαϊκή Ενώσεω σε ανταπόκριση στην κρίση στη Συρία που διαβάστηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπή, στην Επιτροπή Προκελεσμών και ανακοινώθηκε στις 9 Οκτωβρίου στην έναξη της Συνόδου υπήρξαν ενστάσεις μέχρι τις, πρέπει να δοθούν οι ενστάσεις μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα δεν υπήρξαν μάλλον ενστάσεις Οπότε αυτή τη θέση την κοινή την έχουμε διαβιβάσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ομάδες S&D, ID και οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές μου ανακοίνωσαν κάποιες αποφάσεις για αλλαγές που αφορούν ε, τα μέλη των αντιπροσωπιών. Αυτά συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά και θα τεθούν σε ισχύ την ημερομηνία της παρούσης ανακοινώσεως δυνάμει 240 δεύτερη παράγραφος του κανονισμού στις 16 Οκτωβρίου του 2019 διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ε, να συνεχιστεί η εξέταση των εκκρεμών θεμάτων του Κοινοβουλίου. Κατάλογος των διαδικασιών δημοσιευτεί στο παράτημα στα πρακτικά ε, της ε, σημερινής συνεδρίασης. Η διάσκεψη των Προέδρων συνεδρίαση 16 Οκτωβρίου του 2019 μετά από τις συζητήσεις των Επιτροπών Λίμπε και Κοντ ενέκρινε την κοινή συμφωνία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου όσον αφορά το διορισμό της Λάουρα Κοντρούτσα και σαν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Θα υπογραφεί η, συμφων... Ε, εντολή για τον διορισμό της κυρίας Κεβεσή του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τον διορισμό της και τα διορθωτικά για τα κείμενα του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το 241 παράγραφος 4 του κανονισμού αυτές οι διορθώσεις θεωρούνται συγκεκριμένες εκτός αν μέσα σε 24 ώρες από την ανακοίνωση μια πολιτική ομάδα ή αριθμός των βουλευτών που είναι στο ελάχιστο όριο δεν ζητήσουν να ψηφιστούν. Τα διορθωτικά είναι στην σελίδα της Ολομέδειας και, και θα δημοσιευτούν στα πρακτικά αυτής της συνεδριάσεως. Θα ήθελα να ενημερώσω την Ολομέλεια Τετάρτη Σύμφωνα με το άρθρο 79 του κανονισμού του Κοινοβουλίου, μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τέσσερι πράξει συγκεκριμένε από τέσσερι διαδικασίε νομοθετική τη τακτική θα εφετηθούν. Ενημερώσω ότι την Πέμπτη θα υπογράψω μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου τρει πράξει που ανακρίθησαν στα πλαίσια τη διαδικασία τη νομοθετική τη κανονική, σύμφωνα με το άρθρο 79 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Οι τίτλοι αυτών των πράξεων θα δημοσιευτούν στα πρακτικά αυτή τη συνεδριάσεω μετά, μετά από τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων τη Ευρωπαϊκή Ενώση Κυβερνήσεω του Ηνωμένου Βασιλείου και την έξι πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα τη τροποποιημένη συμφωνία απόσυρση, τη χθεσινή ημέρα, το Συμβούλιο το σχέδιο απόφαση τροποποίηση για τη σύναψη τη συμφωνία και διβάστηκε στο Κοινοβούλιο αυτή η συμφωνία. Ε, σήμερα το απόγευμα ε, θα συζητηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα η διάσκεψη των Προέδρων θα συνεδριάσει σήμερα στις 6 το απόγευμα για να συζητήσει τα επόμενα στάδια διαδικαστικά όπως και διαβίβαση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές της αρμόδιες ε, του κειμένου. Τώρα πάμε στις αλλαγές ε, της ημερήσιας διάταξης. Τελικό σχέδιο ημερήσια διάταξη ανακρίθηκε 16 Οκτωβρίου σύμφωνα με το άρθρο 157 των Προέδρων και έχει διανεμηθεί. Να δούμε τι μπορεί να γίνει τη Δευτέρα η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ζήτησε να προσθεθεί μια δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ποινικοποίηση τη σεξουαλική εκπαίδευση στην Πολωνία. Σαν τελευταίο σημείο του απογεύματο πριν σπερεβάσει ενό λεπτού. Θα πρέπει να καταλήξουμε τελικά σε ένα ψήφισμα που θα ψηφιστεί στην πρώτη σύνοδο του Νοεμβρίου. Δίνω το λόγο στον κύριο Ρόμπερτ Μπιεντρόν για να παρουσιάσει αυτό το αίτημα της ομάδας S&D. Έχετε το λόγο. Απουσιάζει. Κύριε Μπιεντρό. Δεν είναι εδώ. Ε, ε Πρόεδρος Ιράτσε, θέλετε να μιλήσετε εσείς. Η ε, κυρία Καρθία, για να στηρίξω την πρόταση της πολιτικής μου ομάδας. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου να είναι σε θέση να συζητά για την ανάγκη να εγγυηθούμε θεμελιώδη δικαιώματα και ό,τι έχει να κάνει με το σεβασμό στην εκπαίδευση και ε, προκειμένου τη σεξουαλική αγωγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση κανονική στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Ποιο είναι κατά, παρακαλώ. Κάποιο θέλει να μιλήσει. Ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι έχω αντίρρηση. Ο, ο βουλευτής Μπιεντρών απουσιάζει. Γιατί ντρέπεται να εμφανιστεί. Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, στην Πολωνία δεν υπάρχει κανένα θέμα απαγόρευσης της σεξουαλικής αγωγής. Απλώς γίνεται λόγος για ένα πρόγραμμα της κοινωνίας που λέει σταματήστε την παιδεραστία. Καλώς, άρα είστε αντίθετος. Λοιπόν, ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία. Βάλτε τις κάρτες σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. Έχουμε με δήλωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ποινικοποίηση τη σεξουαλική αγωγή στην Πολωνία στο τελευταίο σημείο του απογευματινή συνεδριάσεω πριν από τι παρεμβάσει των ενό λεπτού, τη Δευτέρα, δηλαδή σήμερα. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί μέσω ψηφίσματο που ψηφιστεί στην πρώτη σύνοδο του Νοεμβρίου. Πάντα τη Δευτέρα η ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε να προσθεθεί μια δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι καταιγίδε στην Ευρώπη, κυρίω τι μεγάλε οχοπτώσει στην Ισπανία και την ε, θύελα στι Αζόρε, στην Πορτογαλία, τον κυκλώνα στι Αζόρε. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Ιζαμπέλ Μπενζουμέα για να παρουσιάσει το αίτημα του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ομάδας μου, ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε ε, μια νέα απειλή στην Ισπανία, στην Καταλωνία, στη Βαλένθια και στις Βαλεαρίδες ε, νήσους. Στις 12 και στις 15 Σεπτεμβρίου του 19 είχαμε θεομηνίες φοβερές στη Μούρφια, την Αλμερία και το Αλικάντε και στις Αζόρες είδαμε στην Πορτογαλία αντίστοιχα κρέα φαινόμενα. Ο τυφώνας Λορένσο θέλουμε να γίνει συζήτηση για τις συνέπειες αυτών και για να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης έτσι ώστε να καλυφθούν οι πλημμυροπαθείς και όσοι επλήγησαν. Είχαμε και έξι νεκρούς στη Μούρθια από ε, τις φοβερές αυτές ε, καταιγίδες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να παρέμβει κατά. Λαμπέρ. Δεν καταχαστώ του χρόνου σας. Δεν ξέρω αν κανείς θα αντιταχθεί σε αυτό το αίτημα. Εδώ έχουμε ένα αίτημα για να συζητήσουμε δύο συγκεκριμένα στοιχεία που σχετίζουν την αλλαγή του κλίματο. Θεωρώ ότι ήδη έχουμε μια συζήτηση που προβλέπεται στην ημερήσια διάταξη την αλλαγή του κλίματο. Και θα έλεγα θα μπορούσαμε ήδη να προβλέψουμε μία ή δύο ώρε σε κάθε σύνοδο για να συζητήσουμε τι πιο πρόσφατε εκδηλώσει τη αλλαγή του κλίματο. Ε, δεν θα αντίταχθω σε αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να πω να καλέσουμε τους φίλους του ΕΛΚ ίσως να υποστηρίξουν ε, τα μέτρα που ε, καταπολεμούν τα λαγή του κλίματο πιο ένθερμα παραζητούν ε, αυτού του είδου τη συζήτηση όπω αυτή που ζητούν εδώ, σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Πρόεδρο, όμω υπευλήθη το αίτημα, λοιπόν, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προστίθεται λοιπόν η δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι θύρε στην καταιγίδα και τι μεγάλε βροχοπτώσει στην Ισπανία και του κυκλώνε τη Αζόρε, τελευταίο σημείο τη Δευτέρα. Πάντα τη Δευτέρα η ομάδα Γκουε ζήτησε να προσθεθεί μια δήλωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταστολή από το ευρά τη κυβερνήση Χιλή τη κινητοποίηση τη δημόσια κατά τη λιτότητα και το ρόλο του στρατού στην Χιλή. Σαν το σημείο του απόγευματο. Οπότε θα πρέπει να παραταθεί η συνεδρίαση συνεπώ μέχρι τι 10 ώρα το βράδυ. Το λόγο ο κύριο Μποτέγκα για να παρουσιάσει το αίτημα τη Γκου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι πολλοί από εμά με σοκ είδαμε την καταστολή ε, των ε, διαδηλωτών ε, στη Χιλή. Ε, κατάπαυση, ε, απαγόρευση κυκλοφορίας ε, και επιβολή στρατιωτικού νόμου είδαμε στο Σαντιάγο και το Βαλπαραΐζο γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται γιατί αυξήθηκε το ειστήριο του μετρό αυτό μας θυμίζει τις πιο σκοτεινές εποχές της ιστορίας της χώρας και θα ζητούσαμε παρακαλούμε να μας κάνει δήλωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταστολή των λαϊκών διαδηλώσεων από πλευράς της κυβέρνησης της Χιλής και τι ρόλο παίζουν και οι ένοπλες δυνάμεις ως τρίτο θέμα ε, σήμερα το απόγευμα και παράταση συνεδρίασης μέχρι τις 10 το βράδυ. Ευχαριστώ. Ε, κανείς θέλει να μιλήσει κατά. Όχι, λοιπόν. Ψηφίζουμε λοιπόν το αίτημα αυτό. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, η ημερήσια διάταξη παραμένει αμετάβλητη. Κατόπιν των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν μετά τα αιτήματα των πολιτικών ομάδων, προτείνω να παραταθεί η σημερινή σύνοδο ω τι 23.11 το βράδυ. Άρα οι τροποποιήσει αυτέ εγκρίνονται. Την Τρίτη, οι Πράσινοι και η Γκουε ζήτησαν δήλωση Συμβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση στην Καταλωνία μετά την καταδίκη των ηγετών τη καταλανική πολιτική ε, κοινότητα και τη κοινωνία των πολιτών. Και να προσθεθεί ω τέταρτο θέμα το απόγευμα. Δίνω το λόγο στον κύριο Λάμπερτ για να υποβάλει το αίτημα των Πρασίνων. Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχει μπλοκαριστεί εξέταση του καθεστώτος της Καταλωνίας, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα πλέον ε, μετά τη διένεξη Ισπανικών αρχών και Καταλανικών. Με τα δικαστήρια δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν αποφάσεις των Ισπανικών δικαστηρίων, αλλά δεν επιφέρουν πολιτική λύση στο ζήτημα. Επίσης μπορεί να λυθεί με βία το ζήτημα αυτό σε καμία περίπτωση. Οπωσδήποτε όχι. Δεν μπορεί να καταστέλλονται οι διαδηλωτέ. Ε, γι' αυτόν ακριβώ το λόγο και επειδή θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τέτοια λύση σε προβλήματα πολιτικού χαρακτήρα παρά μόνο με πολιτικά μέσα και πρέπει εμείς να δώσουμε το παράδειγμα, Γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε με ε, νυφαλιότητα και με επιχειρήματα την κατάσταση ενός ε, κράτους μέλους, την πολιτική κατάσταση και ενός σημαντικού κράτους μέλους. Οπότε προφανώς θέλω να υποστηρίξω το αίτημα αυτό και ε, έρχομαι και εγώ ίδιος από ένα μικρό έτσι κι κράτος μέλος, δεν μιλάμε μόνο για τα μεγάλα. Πρέπει όμως να γίνει μια νυφάλια συζήτηση που στόχο να έχει να συνεισφέρει σε μια πολιτική επίλυση του θέματος για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή υπέρ η παρέμβαση αυτή και τώρα κατά ο κύριος Μορένο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε αντίθετοι με τη συζήτηση αυτή, διότι δεν έχει κανένα νόημα να φέρουμε ένα εσωτερικό θέμα κράτους μέλους στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένα κράτος μέλους όπου λειτουργεί θαυμάσια και άριστα η δημοκρατία. Είναι μια σύγχρονη δημοκρατία, ανοιχτή, εδρεωμένη και διαφανής η Ισπανία. Η Ισπανία είναι κοινωνικό κράτος δικαίου με ε, απόλυτη και αυστηρή διάκριση των εξουσιών. Και ουδή, επαναλαμβάνω, ουδή δεν είναι υπεράνω του νόμου. Όλοι οι Ισπανοί άνδρε και γυναίκε ξέρουμε ότι αν παραβαίνουμε τον νόμο θα υποστούμε τι συνέπειε. Όλοι οι πολίτε, άνδρε και γυναίκε και ιδιαίτερα οι πολιτικοί, θα πρέπει να σεβόμαστε ε, και να εφαρμόζουμε τι δικαστικέ αποφάσει. Αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί ούτε εδώ ούτε σε κανένα άλλο ε, δημοκρατικό κράτο του, του κόσμου. Και τώρα θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι στην Καταλωνία και να μην κάνουμε εδώ μια συζήτηση στήρα και επιζήμια για την συμβίωση στην Καταλωνία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μονσεράτ. δικά. Ζήτησα ε, το λόγο. Από το ΕΛΚ ψηφίζουμε και εμείς ψηφίζουμε κατά. Ναι, μπορώ να μιλήσω. Όχι. Ναι, αλλά εμεί είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, το ΕΛΚ. Με συγχωρείτε, αλλά γνωρίζετε τον ιστορικό κανονισμό. Ένα και ένα. Θα ψηφίσουμε τώρα για το αίτημα διανάταση τη χειρό. Ποιο είναι υπέρ τη πρόταση των Πρασίνων και τη Γκουε. Σηκώστε το χέρι, παρακαλώ. Κατά. Ποιο απέχει. Απορρίπτεται και παραμένει όσο έχει ημερή σε διάταξη. Ε, Με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Κανένα τσεκ δεν θα κάνουμε τώρα. Καλό τους κλητήρες να ζητήσουν από τους ε, θεατές μας, από τους παριστάμενους να καθίσουν στις θέσεις τους. Αυτό λέω. Δεν με ακούτε. Ζητώ από τους κλητήρες να υποχρώσουν το κοινό να καθίσει. Παρακαλώ. Πρόεδρε, το βλέπω και το λέω. Αυτό λέω. Ευχαριστώ. Η ομάδα Γκουε ζήτησε οι δηλώσει του Συμβουλίου και Κοιτάξτε, μπορώ και να ε, οργανώσω ψηφοφορία, αλλά ήταν τελείω δυσανάλογο το αποτέλεσμα. Φαινόταν. Ήταν ξεκάθαρο. Με συγχωρείτε. Μιλήστε στο μικρόφωνο επιτέλους. Πρόεδρε, Βάσει των κανόνων σας, το σώμα αυτό ψήφισε κατά του να επιτρέψουμε για μια τόσο μικρή διαφορά να ε, συζητήσουμε τις αποτρόπες πράξεις τη Ισπανία στην Καταλωνία. Ο κόσμος αξίζει να γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι βουλευτές εδώ που ψήφισαν κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, πρόεδρος, με συγχωρείτε εσείς τι πιστεύετε, τι ψήφισαν δηλαδή οι συνάδελφοι. Ψήφισαν για την να γίνει συζήτηση, ψήφισαν κατά τη συζήτηση. Σα ζητάω να ελέγξετε. Ωραία λοιπόν, να κάνουμε επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για πρόταση των ομάδων των ε, Πρασίνων και της Γκουε για τη συζήτηση της Καταλωνίας. Πέρας. Ερεσπίντα. Απορρίπτεται. Είχατε αμφιβολίες, συνάδελφε. Δεν υπήρχαν αμφιβολίε. Η ομάδα Γκουε ζήτησε δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την κατάσταση των μεταναστών στη Βοσνία και συγκεκριμένα στο Μπιχάκ, Μπιατς, να προσθεθεί στην απογευματινή συζήτηση ως έκτο σημείο μετά τη δήλωση του Συμβουλίου για την κατάσταση ε, του, της αποκάλυψης φορολογικών πληροφοριών για τα εισοδήματα ορισμένων εταιριών και θηγατρικών στην δημόσια υποβολή εκθέσεων αναχώρα θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να παραταθεί η σύνοδο ω τι 10. Δίνω το λόγο στην κυρία Έρνστ για να υποβάλει το αίτημα τη ΚΟΕ. Παρακαλώ, κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, περί τίνο πρόκειται. Είναι η ανθρωπιστική καταστροφή εκεί, στον καταβρισμό Μούτσακ, κοντά στον Μπίχατ, στη Βόρεια Βοσνία. Ο Δήμαρχος Μάτεα ε, ζήτησε επανειλημμένα από την κυβέρνησή του να τον υποστηρίξουν ε, οικονομικά και είπε το Σαββατοκύριακο ότι τελειώνουν τα τρόφιμα και ε, το νερό και τα φάρμακα. Τι σημαίνει από σήμερα δηλαδή, από σήμερα δεν έχουν καθόλου ανεφοδιασμό. Είναι 2.000 με 2.500 άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς ζουν σε μια χωματερή. Το Πίχατς έχει αποταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση φωνή βόντο σε την ε, Ερήμο. Εδώ και ένα χρόνο είναι γνωστή η δύσκολη κατάσταση σε αυτό το καταβλισμό. Τον έχουμε συζητήσει και εδώ και η ε, Επίτροπος ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει και η ύπατη αρμοστία έχει κρούσει τον κόδωνα κινδύνου λόγω της τρεις κατάστασης. Γι' αυτό, επειδή πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς ζητάμε δήλωση Κομισιόν και Συμβουλίου. Ευχαριστούμε. Ποιος θέλει το λόγο για να μιλήσει κατά. Παρακαλώ. Πρόεδρε, χαίρομαι που η Γκούε το θέτει αυτό το θέμα, διότι η κατάσταση πράγματι είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Πολύ οξία. Θέλουμε αυτό το θέμα να συζητηθεί όπως πρέπει σε αυτή την Ολομέλεια και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα ήταν αποτελεσματικό το να διεξαχθεί μια συζήτηση μαζί με ψήφισμα και εντός δύο εβδομάδων στη Μήνυο Ολομέλεια του Νοεμβρίου στην πρώτη σύνοδο να διεξεχθεί. Του Νοεμβρίου αυτή είναι η πρότασή μου, ούτω ώστε να γίνει διεξοδικότερη ανάλυση και ελπίζουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην συζήτηση. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Στρίχ. Και τώρα να ψηφίσουμε για το αίτημα που υποβλήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται τώρα. Εψήφισαν άπαντέ. πέρας. Απορρίπτεται. Η ημερήσια διάταξη παραμένει απαράλλαχτη. Οι πράσινοι ζήτησαν η συζήτηση τη Τετάρτη για τι δηλώσει του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άνοιξη προ χώρε για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία να ολοκληρωθεί με ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί επίση την Πέμπτη. Ποιο θέλει να υποστηρίξει το αίτημα από του Πρασίνου, κύριε Λάμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απόφαση που ελήφθη από το Συμβούλιο την Παρασκευή, την Πέμπτη το βράδυ, να μην ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει ένταξη με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, θεωρούμε ότι είναι ένα μήνυμα εξαιρετικά, εξαιρετικά ανησυχητικό. Είναι σαφέ για μα ότι αυτέ οι χώρε θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στείλαμε ένα αρνητικό μήνυμα για να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις που εξυπακούεται ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις χρειάζονται κάποιο χρόνο. Κεφαλαιόδου σημασία στο κοινοβούλιο μας να τοποθετηθεί σαφέστατα από αυτού. Βέβαια μια συζήτηση θα το επιτρέψει αυτό να γίνει, αλλά ένα ψήφισμα θα εξέφραζε ακόμα πιο ισχυρότερα τη θέση μας ε, έναντι των συμπερασμάτων που υιοθέτησε το Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, επιμένουμε επί του γεγονότος ότι αυτό το Κοινοβούλιο θα πρέπει να θετήσει αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Λάμπερτς. Ποιος θέλει να υποστηρίξει, να πάρει το λόγο κατά. Ψηφίζουμε το αίτημα, διανάταση της χειρός. Ποιος συμφωνεί, παρακαλώ υψώστε τα χέρια σας. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η πρόταση. Η συζήτηση για τι δηλώσει του Συμβουλίου για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία θα ολοκληρωθεί με την ψήφιση ψηφίσματο. Την Πέμπτη θα ψηφιστεί. Για την Τετάρτη ζήτησε Γκουε η ε, συζήτηση ε, με το Συμβουλίο και την Ευρωπαϊκή Τροπή για την ε, πολιτική δήλωση του ΟΗΕ για την υψηλό επίπεδου κάλυψη και την οικουμενική υγεία, την παγκόσμια υγεία, να ολοκληρωθεί με ψήφισμα. Δίνω το λόγο στον κύριο Φερέιρα για να υποστηρίξει το αίτημα. Παρακαλώ, κύριε Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακριβώ η ομάδα GUE NGL προτείνει η συζήτηση που θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ για την καθολική υγειονομική κάλυψη και για την ε, πολιτική δήλωση του ΙΕ ε, υψηλού επίπεδου για το θέμα αυτό να συνοδευτεί από ψήφισμα που θα ψηφιστεί στην επόμενη σύνοδο, την 1η του Νοεμβρίου. Ωραία. Υπάρχει κάποιο κατά, όχι. Άρα διανάτωση τη χειρός ψηφίζουμε ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η ημερήσια διάταξη παραμένει ως έχει. Για την Τετάρτη πάλι η ομάδα ΕΝΤΗ ζήτησε δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δίωξη των χριστιανών στην Αλγερία να προσθεθεί πριν από τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την έναρξη διπλωματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία ως θέμα. Δίνω το λόγο στον κύριο Ζερόμ Ριβιέρ για να υποβάλει το αίτημα, να υποστηρίξει το αίτημα εκ μέρου τη ομάδα ID. Ευχαριστώ, Προεδρέ, συνάδελφοι κλείνουν εκκλησίες, ε, σκυλεύονται ε, νεκροταφεία παντού στην ε, Βόρεια Αφρική, διώκονται οι χριστιανοί και η κατάσταση μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ειδικά στην Αλγερία θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποιος που θα ήθελε το λόγο κατά... Η πρόταση ψηφίζεται τώρα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται αυτό. Ψήφισαν άπαντες πέρας. Quindi l'ordine del giorno rimane invariato. Παραμένει ως έχει μερίσια διάταξη. Για την Πέμπτη, η ομάδα ΕΛΚ ζήτησε συζήτηση για την Ουγγάντα, ιδίω η πρόταση νομοσχεδίου που προβλέπει θανατική ποινή για τι ομοσεξουαλικέ ε, ε, ε, σχέσει να ακυρωθεί από την ημερήσια διάταξη. Δίνω το λόγο στον κύριο Γκάλερ για να υποβάλει το έτοιμο εκ μέρου του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Yes, colleagues. Συνάδελφοι, επίγον είναι κάτι που είναι επίγον, γιατί επίκειται κάτι αρνητικό να γίνει στα κατεπήγοντα εγγράφει και αυτό το θέμα, αλλά εμείς το διασταυρώσαμε με τους δικούς μας εκεί στην Καμπάλα και ακούσαμε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αυτή τη στιγμή ούτε της κυβέρνησης ούτε της Βουλής της Ουγγαντά να επαναφέρει αυτή τη σκληρή και ε, ε, φρικτή ε, νομοθεσία που ίσχυε στο παρελθόν και εγκαταλείφθηκε μετά από διεθνείς διαμαρτυρίες. Θεωρούμε λοιπόν ότι το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι κατεπήγον. Γνωρίζω τους συναδέλφους της χώρας αυτής εδώ και πολλά χρόνια και φοβούμε ότι εάν συζητούμε θέματα που δεν είναι επίκαιρα εκεί ε, και ε, υποκρινόμαστε ότι είναι, θα επιτύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό. Ας επαγρυπνούμε να δούμε τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κατεπήγον, δεν σχεδιάζουν καμία σχετική νομοθεσία, δεν υπάρχει θέμα. Ευχαριστώ. Ποιο θέλει να πει το αντίθετο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίω κατανοώ τη λογική που ακολουθεί το ΕΛΚ. Εκείνη εξάλλου πρότεινα το θέμα αυτό στο κατεπήγοντα και συμφωνούμε πράγματι ότι ε, δεν είναι πλέον είμαστε κατά της απόσυρσης αλλά η αλλαγή του τίτλου διόρθωση του τίτλου και να πούμε την κατάσταση των, ΛΟΑΔ, των ΛΟΑΤΚΙ στην ΟΓΚΑΝΤΑ, γιατί είναι αυτό αρκετό για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε στα κατεπήγοντα. Ευχαριστώ, κύριε Πύρη. Ψηφίζουμε λοιπόν το αίτημα. Δυνατά σα τη χειρό. Ποιο είναι υπέρ. Υπέρ τη προτάσεώ σα. Κατά. αποχές. Θα γίνει μια επαλήθευση ηλεκτρονική. Ξεκινάει. Πέρας. Απορρίπτεται. Αμεκτάβλητη. Υπάρχει έτοιμα, της κυρίας Πύρη να αλλάξουμε τον τίτλο. Αν μπορείτε καλύτερα να εξηγήσετε. Κυρία Πύρη παρακαλώ. Ο τίτλος, ο νέος τίτλος θα ήταν «Η κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ στην Ουγκάντα». Δυνατά ισχυρός, Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για την πέμπτη η ομάδα Renew Europe ζήτησε πληροφορία για τις δύο ενστάσεις δυνάμει το άρθρο 112 του κανονισμού να αναβληθούν, ε, να μετατεθούν στην Τετάρτη. Ε, κύριε Τόρβαλτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με τον άρθρο 112 θα ήθελα ε, όπως, από, για, το, για το Β να πάει τετάρτη ψηφοφορία. Και χρειάζεται και δική πλειοψηφία για να περάσει. Αν γίνει αυτή η μετάθεση από πέμπτη τετάρτη. Θέλει να παρέμβει κανείς αντίθετα από αυτή την πρόταση. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Λίζε, το συζητήσαμε με ε, εκείνους που υπόβαλαν το, το αίτημα. Ε, προτείνω μια συμβαστική λύση ε, και τα δύο είναι περίπλοκα τα θέματα και χαιρόμαστε για κάθε ώρα που θα έχουμε παραπάνω να το συζητήσουμε με υπηρογνώμονες. Αλλά επειδή πρόκειται για τις μέλισσες και χρειαζόμαστε ενισχυμένη πλειοψηφία να το βάλουμε την Τετάρτη. Αλλά όχι για το χρώμιο. Για το χρώμιο δεν χρειάζεται ε, ε, ειδική πλειοψηφία ενισχυμένη. Αυτό μπορεί να μείνει την Πέμπτη. Για τις μέλισσες να πάει την Τετάρτη. Ε, Κύριε Τόρβαλτς, συμφωνείτε εσείς. Πού είσαστε. Τόρβαλτς. Κύριε Τόρβαλτς. <laughs> Τόρβαλτς. Κύριε Τόρβαλτς, συγγνώμη, συμφωνείτε ή όχι. Ναι, συμφωνείτε. Συμφωνούμε, λέει και ο Στόρβαλτς. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση Λίζε. Ποιος συμφωνεί, διανατάσσεως της χειρός παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα μία από τις δύο ψηφοφορίες θα μετατεθεί για Τετάρτη. Πέμπτη, η ομάδα ECR και μια ομάδα βουλευτών που είναι τουλάχιστον στο κατώτατο όριο που φτάσουν σαν το πρωί της Πέμπτης από το σημείο να βάλουμε προφορική ερώτηση όσον αφορά τη λειτουργία της εταιρική αγοράς. Δίνω το λόγο στον κύριο Ζλοτόφσκι για να παρουσιάσει το αίτημα της ομάδας ECR. Έχετε το λόγο κύριε Ζλοτόφσκι. E, e- Ευχαριστώ πρόεδρε το Ευρωκοινοβούλιο ήδη από την περασμένη φοιτεία έχει εγκρίνει ένα πακέτο για την κινητικότητα, ε, τροποποιώντας την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι τριμερείς διάλογοι για το θέμα αυτό και σχετικές διαπραγματεύσεις χωρίς όμως... να λάβουμε υπόψη τις νέες νομοθετικές διατάξεις και πώς θα επηρεάσουν την εσωτερική αγορά αυτές, ή τις θέσεις εργασίας, ή τις τιμές, διότι η εφαρμογή ενό τέτοιου νομοθετικού πακέτου φυσικά θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει και να μελετήσει προσεκτικά, παρουσιάζοντά μα τα αποτελέσματα και τα πορίσματα, του τι θα γίνει αν εφαρμοστεί αυτό το πακέτο. Θα ήθελα να μάλιστα να οργανωθεί ονομαστική ψηφοφορία Παρακαλώ, εσείς έχετε να πείτε κατά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση για το πακέτο της κινητικότητας ήταν πραγματικά αμφιλεγόμενη και έχει διαρκέσει χρόνια. Ακόμη το θέμα είναι αμφιλεγόμενο και διχάζει ε, Επιτροπή και Συμβούλιο. Όμως, στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Τραν, είχε γίνει δύση ψηφοφορία και είχε αποφασίσει να σταματήσουν οι διαπραγματεύσει. Να αποσυρθούν προκειμένου να, γίνεται μεταξύ μια μελέτη αντικτύπου. Ήταν σαφέ αυτό στι ε, συζητήσει των τριμερών διαλόγων. Ε, και οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ λοιπόν το έχουν υποστηρίξει αυτό στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων και οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει συζήτηση σήμερα και δεν νομίζω ότι θα αρκέσει να το δει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του τριμμένου διαλόγου. Ευχαριστώ, αλλά διανάτε ισχυρό να ψηφίσετε για την πρόταση του κυρίου Σλοτόφη, παρακαλώ, υπέρ. Κατά, παρακαλώ. Αποχέ. Απορρίπτεται, θα έλεγα. κάνουμε μια επαλήθευση όμω. Αυτό λέω, αυτό λέω. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. απορρίπτεται, οπότε η μερίσια διάταξη παραμένει αμετάβλητη. Ονομαστική ψηφοφορία. Υπάρχει διαδικαστικό. Ε, συνάδελφε Πάντσα, έχετε το λόγο. Ε, στις 12 Οκτωβρίου δυνάμει το άρθρο 158 για τη συζήτηση της Τετάρτης το πρωί. Στις 12 Οκτωβρίου η Εύριν Καλάφ δολοφονήθηκε ε, όταν ταξίδευε ήταν στο δρόμο. Η Εύριν Καλάφ ήταν η γενική γραμματέας του κόμματο Συριακού ήταν μαχήτρια για την δικαιώματα της, ε, των γυναικών και ήθελε επίσης να προωθήσει και πρόγραμμα ίνευσης. Δεν, υπήξες, δεν ανεκαλύφθη ποιο ήταν υπεύθυνο για την εκτέλεση, αλλά υπάρχουν υποψίε για, τον, για την Αράρα Τσατζίβα, μια ομάδα επαναστατών Ισλαμιστών που βγήκαν από την ε, Αλνούζρα που ανήκουν τώρα στον Εθνικό Συριακό Στρατό που γεννήθηκε υπό την αιγίδα της Άγκυρας. Τι πρόταση κάνω σε εσά, Πρόεδρε, γνωρίζοντα ότι έχουν εκπνεύσει πλέον προθεσμία, επειδή είναι σημαντική αυτή η πράξη από πλευρά πολιτική, ε, να, να είναι υποψήφια για το 2019 βρήν Καλάφ και το βραβείο Ζαχάροφ. και αν έχει κλείσει για φέτος για το 2020, θα είναι σημαντική πράξη για το Κοινοβούλιο, μια πράξη ε, έναντι πολύ ανεκτική τάση που έχουμε δείξει έναντι της Τουρκίας και μια αναγνώριση εκείνων που θυσίασε τη ζωή του για τη δικαιώματα των ανθρώπων. Είναι μια διευθυντική κίνηση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Θα ελέγξουμε, θα κάνουμε τα δέοντα για τα τιμά σας. Λοιπόν, έχουμε καθορίσει λοιπόν τα διάφορα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τη δήλωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι συνέπειε χρεοκοπία του ομίλου Τόμας Κουκ. Um, Παρακαλώ, πηγαίνετε στους διαδρόμους για τις συζητήσεις σας, διότι πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση, αφού εγκρίθηκε πλέον η μερίσια διάταξη. Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ε, ήθελα να πω ότι ακολουθεί η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Τόμας Κουκ. Θα ήθελα να σας πω πριν από τη συζήτηση το εξής. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την μπλε κάρτα σας, υπάρχει νέα διαδικασία ηλεκτρονική, αλλά ισχύουν και οι δύο ε, διαδικασίες. Αν θέλετε να κάνετε ερώτηση σε κάποιο μιλητή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπλε κάρτα κανονικά ή με τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία, όπου και θα χρειαστείτε την ε, κάρτα ψηφοφορία σα. Επίση, την κάρτα ψηφοφορία μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να ζητήσετε το λόγο στο Catch the Αμέσω μετά ε, την ομιλία τη Επιτρόπου θα ανοίξει το σύστημα. Παρόλο που υπάρχει μια σχετική οχλαγωγία, θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, κυρία Τάισεν. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί σοβαρά με την πρόσφατη δήλωση χρεοκοπίας της Thomas Cook. Ήταν σημαντική η οικονομική δραστηριότητα του ομίλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβάλλει στο 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ εμέσως και απευθείας και απασχολεί πάνω από 25 εκατομμύρια ανθρώπους, 11% της συνολικής απασχόλησης τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Για ορισμένε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα, ο τουρισμός είναι η κύρια πηγή εισοδήματο. Ο τουρισμός είναι επίσης ε, πλήρως συσχετισμένος με άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Ένα ευρώ προστιθέμενη αξία στον τουρισμό σημαίνει 56 σεντ λεπτά ε, προστιθέμενη αξία σε όλου του υπόλοιπου. Στον τομέα αυτό δεν ενεργοποιούνται μόνο μεγάλοι ομιλοί, αλλά μεταξύ των 2,2 εκατομμυρίων επιχειρήσεων που ενεργοποιούνται στον τουρισμό, 19% είναι μικρομεσαίε. Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών κάνει τον τομέα του τουρισμού όχι μόνο περίπλοκο, αλλά τον συνδέει απευθείας και με άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η ατυχής ε, χρεοκοπία της Thomas Cook το δείχνει αυτό ανάγλυφα. Δείχνει για άλλη μια φορά ότι ο τουρισμός και όλες οι σχετικές δραστηριότητε απαιτούν μια ενιαία προσέγγιση μέσα από, που να διέπει όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Είμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη για να ε, υπολογίσουμε τον αντίκτυπο ως προς τις επιχειρήσεις, τις θέσης και τους ταξιδιώτες, τους τουρίστες που επλήγησαν ανάλογα με την κάθε περιοχή. Καθώς και να ε, ανταλλάξουμε πληροφορίες πληροφορίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να ε, καλύψουμε τι δυσκολίε. Ε, υπάρχουν διαφορετικά μέσα σε διαφορετικού πολιτικού τομεί, τα οποία θα κινητοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Πρώτον, μπορούμε να βοηθήσουμε τι αρνητικέ επιπτώσει στον κόσμο που επληγεί με την απώλεια τη θέση εργασία του. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, το EGF, είναι μια σαφή εκδήλωση τη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη παρέχει ε, αρρωγή σε αυτούς που έχασαν τη δουλειά τους και θα τους βοηθήσει να βρουν νέα δουλειά ε, με δημόσια ε, στήριξη. Το ταμείο αυτό βεβαίω ε, εκταμιεύει ποσά προ τα κράτη-μέλη βάσει ορισμένων ε, προποθέσεων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαθέσιμη να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη που πρέπει. Επίση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να βοηθήσει για την επανεκπαίδευση, την επανακατάρτιση και την αναζήτηση εργασία του ανθρώπου αυτού. Μετά, τα εργαλεία τη πολιτική συνοχή μπορεί να βοηθήσουν τι περιοχέ. Ευρω... Επίση, το Ταμείο ε, Ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Περιφοριών μπορεί να βοηθήσει τις περιοχές που δημιουργίζουν προβλήματα ε, για την απαλλαγή από τον άνθρακα, τις ε, φυσικές καταστροφές, ε, περιοχές που πρέπει να διαφοροποιήσουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες, να μην εξαρτώνται πλήρως από τον τουρισμό, να απαλλαγούν από τη βιομηχανία και το καθεξής. Η βοήθεια του Ταμείου αυτού προκύπτει από τις διαχειριστικές αρχές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσα από επιχειρησιακά προγράμματα. Τρίτον, οι ευρωπαϊκοί κανόνε κρατική βοήθεια με ευελιξία για να υποστηριχθούν επιχειρήσει που έχουν πρόβλημα ρευστότητα ε, σε άμεσο χρονικό ορίζοντα και υπό συγκεκριμένε προποθέσει. Ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέψουν ε, προγράμματα για να υποστηρίξουν μικρομεσαίες που έχουν οικονομική δυσχέρεια. Και ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να κοινοποιηθεί βεβαίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαίρως για να εγκριθεί. Τέταρτο, για το θέμα των ταξιδιωτών και των δικαιωμάτων τους. Η οδηγία για τα ταξίδια πακέτα υποχρεώνει τους tour operator, τους υπεύθυνους διοργάνωσης ταξιδιών, να ε, φροντίσουν τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών στην ε, χώρα αφετηρίας τους, σημεία αφετηρίας τους και την αποζημίωσή τους. Κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Αυτό είναι δωρεάν ε, υπηρεσία προς τους ταξιδιώτες. Ο επαναπατρισμός παγκοσμίω για όλους τους τουρίστες που ταξίδεψαν με την Thomas Cook. Η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή αξιολογεί το πώ τα κράτη-μέλη μεταφέρουν την οδηγία για τα ταξίδια σε πακέτο και επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ε, για την αφαιρεγκαιότητα και της όλης πράξης για τη χροκοπία. Ε, Βεβαίω, ελπίζουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί πλήρω το πακέτο τον Ιανουάριο του 2021. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, να θυμίσω και την προτινόμενη αναθεώρηση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών, του κανονισμού 261-2004 και με αυτή την αναθεώρηση σκοπεύουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την συνεπή εφαρμογή των κανόνων για τα δικαιώματα των επιβατών που θα πρέπει να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη και βεβαίω ε, να γίνονται στα πλαίσια των οικονομικών δραστηριοτήτων των αερομεταφορέων. Βεβαίω εδώ ακόμα σε θεσμικό επίπεδο δεν έχουμε συγκεκριμένου ε, κανόνε για περιπτώσει χρεοκοπία αεροπορικών εταιριών. Όμως η προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών και με ανακοίνωση το 2013 ε, καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ήπια μέτρα. Υπάρχουν κάποια λοιπόν εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τον αντικτυπώ αντίκτυπο σε περίπτωση αφαιρεγκαιότητα για του επιβάτε, όπω μια δέσμευση τη εταιρεία να προβλέψει ειδικέ τιμέ για του επιβάτε, κάτι που χρειάστηκε και ενεργοποιήθηκε εδώ σε πολλέ περιπτώσει. Επιπλέον, οι εθνικέ αρχέ σε πολλέ περιπτώσει δραστηριοποιήθηκαν για να διασφαλίσουν την, ε, τον επαναπατρισμό των ε, επιβατών που ξέμειναν. Εδώ λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε τα δικαιώματα αυτών των επιβατών μέσω των διαδικασιών χρονοποίησης και μελλοντικά. Υπό το φως των πρόσφατων εμπειριών μας και των μηχανισμών που διαθέτουμε, κοιτάζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη τι επιλογές υπάρχουν για να δοθεί μια εξακολούθηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των επιβατών σε περίπτωση χρεοκοπίας αεροπορικής εταιρείας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κυρία Επίτροπε, και τώρα έχουν το λόγο οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Ρώσα Εσταράς Φερραγούτ, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα και με δική μας πρωτοβουλία γράψαμε στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα για να προβληματιστεί το Κοινοβούλιο για την πτώχευση της ε, Τόμας Κουκ έχει 178 έτη ιστορίας, πέρασε δύο πολέμους, αλλά δεν άντεξε ε, τις αβεβαιότητες του Brexit, την ψηφιοποίηση και το μέλλον του νέου κόσμου του 21ου αιώνα. Οφείλουμε να προβληματιστούμε γιατί ε, ε, είχε πάνω από 200 ε, ξενοδοχεία, 500 πρακτορία, 22.000 εργαζομένους. Ε, οι Βαλεαρίδες μαζί με τα Κανάρια νησιά, την Ανδαλουσία και την Καταλωνία πλήττονται ιδιαίτερα όχι μόνο γιατί χάνουν θέσεις απασχόλησης αλλά γιατί έχουν ξεμείνει πάρα πολλοί τουρίστες ε, στα νησιά αυτά και στις άλλες περιφέρειες. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι η χρεοκοπία αυτή έχει φέρει προβλήματα και στο γενή τομέα και στις μεταφορές, όχι μόνο στα ξενοδοχεία, στις υπηρεσίες και σε όλη την οικονομία. Γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσουν το θέμα αυτό και να προβληματιστούν σε βάθος και σοβαρά για τον τουρισμό. Ζητάει ο κλάδος στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική για να βοηθήσει ε, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ψηφιοποίησης που αλλάζουν όλα αυτά ραγδαία με ταχύτητα φωτός. Χρειάζεται στρατηγική ο τουρισμός. Ε, είναι πάνω από 4% ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προετοιμάσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία για να απορροφά τους κραδασμούς ε, τέτοιων πτωχεύσεων που έχουν πολλές επιπτώσεις. Επίσης υπάρχουν και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Σε αυτή την κρίση χρειαζόταν περισσότερη πρόληψη αλλά και περισσότερος συντονισμός. Τα κράτη-μέλη στη διαχείρισή τους έχουν φωτεινές και σκοτεινές πλευρές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας πούμε στη δική μου αυτόνομη περιφέρεια, στις Βαλεαρίδες ε, νήσους, είδαμε κάποιες ε, πρέπει, Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με κάποιους φορείς και ε, πώς ε, ασχολείται ο καθένας όταν υπάρχουν τέτοιες χρεοκοπίες. Ε, ε, θα πρέπει να κινητοποιηθεί και το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα ξέρει αυτά η κυρία Τάισον. Υπάρχουν τρομερές συνέπειες, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί στον τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ κυρία Εσταράς. Και τώρα η κυρία Κρίσταλ Σχάλντε Μόζε από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες για δύο λεπτά παρακαλώ. Øh, Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τους εργαζόμενους της Τόμας Κουκ και τους επιβάτες που υπέστησαν τις αρνητικές συνέπειες της ε, κατάρρευσης της Τόμας Κουκ. Για δεκαετίες η Τόμας Κουκ ήταν μια τεράστια επιχείρηση και μετέφεραν πάρα πολλού ταξιδιώτε σε όλο τον κόσμο. Αλλά η εταιρεία δεν υφίσταται πια. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν έχουμε θεσπίσει του απαιτούμενου κανόνε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα χρεοκοπιών για να προστατεύσουμε του καταναλωτέ και του εργαζόμενου. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλέ εταιρείε, ταξιδιωτικέ εταιρείε, αεροπορικέ εταιρείε που καταραίουν. 32 αεροπορικέ εταιρείε έχουν καταρρεύσει. Και αυτό τα τελευταία χρόνια. Η νομοθεσία μας δεν είναι αρκετά καλή ακόμα. Είναι πολύ καλή, έχουμε πόρους που μπορούν να βοηθήσουν, είναι καλύτερα το τίποτα. Συμφωνώ, αλλά εμείς οι σοσιαλιστές θα θέλαμε να δούμε πιο αυστηρή νομοθεσία στον τομέα αυτών. Ε, πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τι αεροπορικέ εταιρείε και τι ταξιδιωτικέ εταιρείε, ταξιδιωτικά γραφεία στην Ευρώπη. Πρέπει να αισθάνεται κανεί ασφαλή και άνετο όταν ταξιδεύει στην Ευρώπη και όταν κανεί εργάζεται στι εταιρείε. Αυτό δεν ίσχυσε για πολλού που εργαζόταν για την Thomas κουκ και που, τους άλλους που χρησιμοποίησαν την εταιρεία για τα ταξίδια τους. Πρέπει να κάνουν περισσότερα. Τα δικαιώματα των επιβατών πρέπει να βελτιωθούν. Το ανέφερε αυτό η Επίτροπος. Είναι ντροπή, κρίμα που δεν σημειώσαμε μεγαλύτερη πρόοδο από αυτή που έχουν πετύχει. Το συζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε πρόταση, θα πρέπει να συμφωνήσει και το Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο. Πρέπει να δούμε κατά πόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να βοηθήσουμε πιο σημαντικά όταν έχουμε χροκοπίες μεγάλων εταιριών που επηρεάζουν πάρα πολλούς ανθρώπους. Χρειαζόμαστε περισσότερη δράση από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, ούτως ώστε οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι να αισθάνονται καλύτερα όταν, όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαλδεμόση. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μπαουθά Ντίαθ από την ομάδα Renew Europe. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η σημερινή συζήτηση δεν αφορά την πτώχευση της Τόμας Κουκ, αλλά πώς αυτή η χρεοκοπία επηρέασε χιλιάδες ανθρώπους και κάποιες περιφέρειες που έχουν ονοματεπώνυμο στην Ισπανία είναι οι Βαλαιαρίδες νήσι, είναι οι Κανάριες νήσι. Μετά από αυτή την αμέλεια μια εταιρεία που ήξερε πολύ καλά ώρες πριν κλείσει ότι θα πτώχευε. Εγώ θα ήθελα να γίνω σήμερα η φωνή όλων αυτών των χιλιάδων τουριστών που εναπόθεσαν ε, αυτές τις προσδοκίες και τις ελπίδες τους όλης της χρονιάς να πάνε διακοπές και να γυρίσουν σπίτι τους. Θέλω να γίνει η φωνή όλων αυτών των καταναλωτών που δεν ξέρουν σήμερα αν θα τους αποζημιώσουν. Θέλω να είμαι η φωνή όλων εκείνων των εργαζομένων που νυχτιάτικα δύο η ώρα το πρωί ε, είδα να χάνονται οι θέσει εργασία του. Και επίση του γνωρίζω πολλού από εκείνου. Είναι εξαιρετικοί επαγγελματίε. Σήμερα εξακολουθούν να εργάζονται απλήρωτη, ακριβώς ε, επειδή δεν γνωρίζουν τι πρόκειται να γίνει και τι λέει η εργατική νομοθεσία και πώς τελικά θα αποφανθεί η δικαιοσύνη και τι θα τους ξημερώσει. Επίσης θέλω να είμαι η φωνή όλων των ξεναγών, όλων των οδηγών που δεν ξέρουν του χρόνου τι θα γίνει στην επόμενη σεζόν. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Κομισιόν και ε, μην μας λέτε λόγια. Έργα χρειάζονται και εξ ονόματος των Θιουδαδάνος και του Renew Europe, της φιλελεύθερης ομάδας, θέλω να πω σε όλους ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουμε στη μοίρα τους. Θα το πάμε μέχρι τέλους δεν μπορούν να επιτρέπονται τέτοια φαινόμενα. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα. Ω πολίτε από τις Βαλεαρίδε νήσους, όπου είχα την τιμή, τη χαρά ε, να ε, είμαι και περιφερειάρχης, ξέρω πολύ καλά από πρώτο χέρι τι σημαίνει αυτό και πώς υπάρχουν ενεργητικές ε, δημόσιες πολιτικές υπέρ του τουρισμού. Τώρα είναι η ώρα, κύριοι και κυρίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα χέρια μας είναι το μέλλον και από εμά εξαρτάται. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να περάσει. Ευχαριστώ, κύριε Μπαουθά Αντίαθ. Και τώρα, εξ των Πρασίνων και της ε, Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας, η κυρία Ρόουιτς, παρακαλώ. Χιλιάδε ταξιδιώτε δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν και 21.000 ε, άνθρωποι του προσωπικού έχασαν τη δουλειά τους. Και μια πλούσια ελίτ ε, τη γλίτωσε από την κατάρρευση όμως ε, της Thomas Cook. Για κάποιους διαχειριστές των hedge funds και κερδοσκόπους αυτή ήταν ακόμα μια ευκαιρία επιχειρηματική. Δύο εταιρείε μάζεψαν πάνω από 200 εκατομμύρια λίρες όταν κατέρευσε η Thomas Cook. Αυτοί οι καπιταλιστές σαν όρνια πλούτησαν επενδύοντας σε οικονομικά προϊόντα που τελικά πληρώνουν όταν χρεοκοπεί ε, μια εταιρεία. Κάτι που συνέβη με την Thomas Cook. Πέρα από αυτή την ε, παράξενη απόχρωση, την αρνητική απόχρωση του καπιταλισμού, πρέπει να δούμε πώς ο Thomas Cook κατέληξε σε αυτόν τον προορισμό, σε αυτή τη μοίρα. Η εταιρεία ε, απαρέθεση, αβεβαιότητα για το Brexit και κύματα καύσωνας, καύσωνος σαν παράγοντες που συνέτειναν στην κατάρρευση. Τα δύο μεγαλύτερα θέματα των καιρών μας, η αλλαγή του κλίματος και οι ενωτικές συνέπειες αυτού και το Brexit έπαιξαν ρόλο. Οι φθηνές πτήσεις τροφοδοτούν τελικά την αύξηση θερμοκρασία στον πλανήτη. Αυτό με τη σειρά του ε, καθιστά τους δημοφιλείς προορισμούς στην ε, Ευρώπη ε, αφόρητους στην εποχή εχμής της τουριστικής. Η αντιμετώπιση αλλαγής του κλίματος συνεπάγεται νέες μορφές ταξιδίων και διαφορετικά είδη διακοπών, χερσαίας διαδρομές και πιο σταθερές, σταθερούς τόπους διαμονής. Και θα πρέπει τελικά ε, να υπάρξει σωστή μετάβαση για να αντικατασταθούν οι απολεστήσεις θέσεις προς ένα πιο ασφαλές ε, μέλλον. Ε, κυρία Ρόουετ, λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας αυτή και την παρέμβαση. δέχεστε μπλε κάρτα? Ο κύριος Λόγκορθ νομίζω έχει ζητήσει. Ε, ναι, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Για μισό λεπτό, παρακαλώ. Oh, Ευχαριστώ. Ποια ε, απόδειξη έχετε ότι οι εταιρείε οι αεροπορικέ χαμηλού κόστου επηρεάζουν το κλίμα. Δεύτερον, γιατί θέλετε να στερήσετε από τον κόσμο που είναι, δεν έχει πολλά λεφτά τη δυνατότητα να έχει φθηνέ διακοπέ με τι εταιρείε πτήσεων, τι αεροπορικέ εταιρείε low cost. οι αεροπορικέ εταιρείε χαμηλού κόστου δεν προσμετρούν επαρκώς τις συνέπειε των αερομεταφορών στο κλίμα. Οπότε οι εταιρείε low cost ενθαρρύνουν ιδιαίτερα περισσότερες πτήσεις από αυτές που μπορούμε να αντέξουμε λόγω της κλιματολογικής αλλαγής. Εγώ δεν προτείνω να μην έχουμε διακοπές. Προτείνω να υπάρχουν αρκετά μεταφορικά μέσα που είναι φθηνά και να μην αυξήσουμε τόσο θερμοκρασίες που τελικά να τηγανιστεί ο πλανήτης από την αύξηση θερμοκρασίας. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κατάλογο των παρεμβάσεων. Ακούμε τον εκπρόσωπο, τον κύριο Μάρκους Μπουχάιτε. Έχετε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Για ποιο λόγο επτόχευσε η Τόμας Κουκ, που ήταν μια εταιρεία 178 ετών Μπορεί να μην ξέρουμε ακόμα τις λεπτομέρειες, αλλά τις συνέπειες τις ξέρουμε. Μιλούμε για 22.000 εργαζόμενους και μόνο για την Ελλάδα είναι 250 με 500 εκατομμύρια ευρώ οι απώλειες. Τι είναι αυτό. Είναι το αποτέλεσμα αυτό που ακούσαμε. Ε, κυνήγι μαγισσών, δημιουργία εντυπώσεων, Έχουμε το νέο ε, χρυσό μόσχος και την προστασία του κλίματος. Και πρώτο θύμα είναι ο τουρισμός. Ακολουθούν και άλλοι κλάδοι. Και ιδιαίτερα σκέφτομαι τη Βαβαρία, την πατρίδα μου και την αυτοκινητοβιομηχανία ε, που εδρεύει εκεί. Ε, αυτό είναι το πνεύμα των καιρών τώρα, η κλιματική αλλαγή. Απαιτώ αυτό το κυνήγι μαγισσών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ε, βρει μιμητές, αλλά να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Θα πρέπει να αποτρέψουμε ε, τέτοια προβλήματα, τουλάχιστον νομοθετικά εμπόδια να μην βάζουμε στους tour operators, όπως το Ευρωπαϊκό Πράσινο Deal, ας πούμε, και να αναγνωρίσουμε ότι όταν πεθαίνουν τα ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά πρακτορία δεν βοηθάει το κλίμα ιδιαίτερα, απλώς βοηθάει άλλους ανταγωνιστές που θα καλύψουν το κενό. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω κυρίες και κύριοι να δούμε ότι περνάει δυσκολίες ο τουρισμός και να του παρασταθούμε όχι όπως εδώ οι πράσινοι και να υποστηρίξετε παρακαλώ το δικό μας ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μπουχάιτ. Και τώρα για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Ζλωτόφσκι, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η χρεοκοπία της Thomas Κουκ είναι μια δυσάρεστη είδηση. Είναι χιλιάδες οι τουρίστες που επλήγησαν, αλλά είναι αρνητικά τα νέα και για όλο τον κλάδο του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εκτιμηθεί ότι τουλάχιστον το ξενοδοχικό κλάδο, είναι πολλά τα ξενοδοχεία στην Ισπανία και την Ελλάδα που συνεργάζονταν με την εταιρεία και θα πληγούν άσχημα. Όλοι θα υποστούν τις συνέπειες, εμέσως ή απευθείας. Η δική μου χώρα, η Πολωνία, επίσης με, εκατο, με εκατοντάδες ε, χιλιάδες άτομα που ε, έμειναν μπλοκαρισμένοι, έχει επίσης αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν μπορεί να μας πει αν πρόκειται για μια μεμονωμένη περίπτωση ή είναι η αρχή μιας κρίσης στον κλάδο του τουρισμού. Μήπως είναι, να παραγωγηθούμε ότι είναι μεμονωμένη περίπτωση, απομονωμένη διότι είχε κακή διαχείριση στα οικονομικά του ο, ο Όμιλος Τόμας Κούκ είναι μια κρίση του τουρισμού που θα έχει ευρύτερε συνέπειε και προεκτάσει. Πώς το βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δική της τη Σκοπιά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζωτόφσκι. Και τώρα εξ ονόματος της Ανατικής Αριστεράς το λόγο έχει η κυρία Έλενα Κουντούρα. Παρακαλώ για 1,5 λεπτό. ο κλάδος των μεταφορών και του τουρισμού είναι ισχυρός αναπτυξιακός πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας. αντιπροσωπεύει το δέκα του ευρωπαϊκού αεπ και έχει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλών παραγωγικών κλάδων. η σημασία του είναι ζωτική για περιφέρειες και νησιωτικές περιοχές που δεν έχουν άλλους αναπτυξιακούς πόρους. δεν υπάρχει ενιαίος μηχανισμός στήριξης των τοπικών κοινωνιών και των θέσεων εργασίας και κανένας μηχανισμός ενίσχυσης της εικόνας του ευρωπαϊκού τουρισμού που δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με αρνητικές επιπτώσεις για όλους. η ευρώπη είναι ένας ενιαίος κορυφαίος τουριστικός προορισμός και ο τουρισμός αποτελεί το τέταρτο μεγαλύτερο κλάδο εισαγωγών με 27 δις ευρώ πλεόνασμα. ποιος θα τον στηρίξει αν όχι η ίδια η ευρωπαϊκή ένωση; δεν διαθέτουμε τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά κρίσεις που πλήττουν οριζόντια την τουριστική δραστηριότητα στην ευρώπη. έχουμε μόνο μία οδηγία για τον επαναπατρισμό των τουριστών που είχαν αγοράσει ταξιδιωτικά πακέτα και μεμονωμένες κινήσεις κρατών μελών με κριτήριο το εθνικό συμφέρον και χωρίς συντονισμό. θέλω να είμαι σαφής η κατάρρευση του thomas Κουκ δεν αποτελεί τη μοναδική πρόκληση για τη βιωσιμότητα του τουρισμού. είμαστε αντιμέτωποι με την κλιματική κρίση και τα εντυνόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα και επίσης το κρίσιμο θέμα της ασφάλειας τα ζητήματα που κυριαρχεί ανάγκη για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το προσφυγικό. ζητάμε επομένως την ενίσχυση της νομοθεσίας για την προστασία των ταξιδιωτών απέναντι σε έκτακτα γεγονότα όπου ο ίδιος ο τουρίστας δεν φέρει καμία ευθύνη και επιβάλλεται να καταρτήσουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεως στον τουρισμό για τους εργαζόμενους τις τοπικές κοινωνίες και την εικόνα της ευρώπης ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό. Ε, ε, Κυρία Κοντουρά, ε, μιλήσατε δύο λεπτά, ενώ είχατε ένα λεπτό. Οπότε κόβετε μισό λεπτό από άλλο συνάδελφό σα. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο σα. Ο κύριο Κολακούσιτ από του Μία Γεγραμμένου. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε. Εγώ ε, ήμουν δικαστής στην Κροατία ε, την περασμένη οκταετία με ζημίες δισεκατομμυρίων ευρώ ε, που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ε, στον τουρισμό στην Κροατία. Βέβαια, ο Τόμας Κροκούκη μπορεί να είναι τεράστιο πρόβλημα. Αλλά τώρα προσπαθεί κάθε κράτος μέλος να ε, καλύψει την κατάσταση ε, με εθνικά μέσα, ενώ η εταιρεία αυτή είναι πολυεθνική και τα προβλήματα τεράστια όταν χρεοκοπεί μια τέτοια εταιρεία. Εμείς στην Κροατία έχουμε ένα όμιλο που λέγεται Αγκροκό και δραστηριοποιείται σε πολλά κράτη και ε, ανησυχούμε με την κατάσταση ε, γιατί είναι πολύ σκοτεινά τα πράγματα. Και ε, στην περίπτωση Thomas Cook ε, ξέρουμε ότι εργάζονται πάρα πολλοί χιλιάδες άνθρωποι και είναι πάρα πολλοί τουρίστες, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση τι δουλειά έχει να ασχολείται με ε, χρεοκοπίες. Μάλλον όταν είναι πολυεθνικές πρέπει να ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα κράτη-μέλη από μόνα τους. Ευχαριστώ. Και τώρα ε, οι υπόλοιποι ομιλητές. Η κυρία Μοντέρο Ντάγκια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, ευχαριστώ για όλη σας την παρουσίαση, για όλο αυτό το θέμα που πραγματικά για μας είναι κρίσιμο στο Ευρωκοινοβούλιο. Αρκετές φορές η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού στο σώμα αυτό έχει καταγγείλει τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος αυτός. Έχει καταγγείλει την ανάγκη να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας για ένα τουρισμό ο οποίος θα είναι εξυγχρονισμένο. Θα λάβει υπόψη του την ψηφιοποίηση, όπω είπατε. Θα λάβει υπόψη τι κλιματικέ αλλαγέ και τι νέε προκλήσει που έχει να αντιμετωπίσει και που έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα για τόσα πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη συνολικά είναι ένας τουριστικός προορισμός. Σε σχέση με την πτώχευση, με την χρεοκοπία της τόμας Κουκ, ε, για τον Βρετανικό αυτό όμιλο, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι ε, αντίκτυπο είχε και τι κραδασμού προκάλεσε σε αυτόν τον, κλάδο. Είναι πολλά τα άτομα, του πολλοί ταξιδιώτε που παρέμειναν μπλοκαρισμένοι σε πολλά κράτη, μεταξύ άλλων Ισπανία, Πορτογαλία, στη Μαδέρα, ε, στο Αλγκάρβε. Και πραγματικά θα πρέπει να μπορούμε να δούμε και ποσοτικά τι αντίκτυπο είχαμε και αυτή η πτώχευση τι προκάλεσε. Πρέπει να ξαναδούμε πώ θα υποστηρίξουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, πώ θα υποστηρίξουμε του καταναλωτέ και πώ θα ε, αποκαταστήσουμε τα δικαιώματα των επιβατών. Ε, Επιβάτε που δημιούργησαν, αντιμετώπισαν πραγματικά δύσκολε συνθήκε λόγω τη πτώχευση και πώ θα προστατεύσουμε αυτόν τον τόσο σημαντικό κλάδο. Πραγματικά η απουσία τη εταιρεία αυτή θέτει να αμφιβόλο πολλέ ευρωπαϊκές περιοχέ ω προορισμούς και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μοντέιρο Ντεγκιάρ. Επόμενος ο κύριος Ντάνιελσον. Ευχαριστώ πρόεδρε θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την ε, λύπη μου και τη θλίψη μου για την ε, ε, πτώχευση της Τόμας του Χουκ. Τουλάχιστον 22.000 έμειναν χωρίς δουλειά, αλλά και 3.000 30.000 παρέμειναν μπλοκαρισμένοι στους προορισμούς τους. θα πρέπει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά Όργανα να λάβουν μια θέση που να έχει κάποιο αποτέλεσμα ω προ τα δικαιώματα των επιβατών. Το ζητάει το Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω, χάρη σε πολλού εργαζόμενου που ε, εργάστηκαν εργάστηκαν μισθεί κατάφεραν να βρουν μια λύση για πολλούς από αυτούς τους ταξιδιώτες. Ταυτόχρονα δεν ξέρουμε ακριβώς τι ανταμοιβή ε, θα πάρουν μακροπρόθεσμα οι άνθρωποι αυτοί που μείναν χωρίς δουλειά, τι ε, σύνταξη. Πρέπει λοιπόν για το μέλλον τους κάτι να κάνουμε, να φροντίσουμε να υπάρξει διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αμέσω το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και κανένα εργαζόμενο της Thomas Cook να παραμείνει ε, ε από την πτώχευση της Thomas Cook. Ευχαριστούμε κύριε Ντάνιελσον. Και τώρα κυρία Χαραντζόβα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ και Πρόεδρε. Η κατάρρευση τη Τόμας Κούκ επηρεάζει όλη την Ευρώπη. Πάνω από μισό εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτε είχαν μείνει ξέμειναν σε διάφορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπει κανεί πόσο σημαντική είναι η προστασία κατά τη αφαιρεγκαιότητα και καλύψει και αποζημιώσει σε περίπτωση που οι, οργανω... εταιρείε που οργανώνουν ε, τα ταξίδια χρεοκοπήσουν. Η Νέκερμαν, όπω είναι το όνομα στο Μασκούκ στη χώρα μου, κατάφερε ε, να ε, πιστέψουν ε, να καλύψει τελικά τις, ε, χωρίς να πάρει από ε, το Ταμείο Εγγυήσεων χρήματα να αποζημιώσει τους επιβάτες και θα δώσει τελικά διακοπές στους πελάτες που ήδη έχουν πληρώσει τα ταξίδια τους. Αυτό πρέπει να ειδωθεί σαν ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς μια κατάσταση χρεοκοπίας χωρίς να είναι επιβλαβής η κατάσταση για τους πολίτες και να λεχιστοποιηθούν οι απώλειες τους. Όπως ήδη ακούσαμε σήμερα, αυτό πόρο απέχει από άλλες χώρες, από τις συμβαίνει άλλες χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, τελικά η οδηγία ε, πρέπει να θεσπίσει, να εφαρμοστούν ε, τα μέτρα της οδηγίας και να υπάρχουν ταμεία που καλύπτουν τις ανάγκες. Θα πρέπει να καλύπτονται οι πολίτες που επηρεάζονται από τη χρεοκοπή στο Μασκού και των θηγατρικών στο Μασκού. Και η κατάσταση αποδεικνύει ότι η οδηγία ε, για τα ταξιδιωτικά πακέτα λειτουργεί σε αυτές τις περιστάσεις, αλλά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Σε δύο χρόνια η οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Ελπίζω να μπορέσουμε να μάθουμε από αυτά που συνέβησαν τώρα και να δούμε πού χρειάζεται να επιφέρουμε ακόμα βελτιώσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Χαράσοβα και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Χάιντερ. Έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η οδηγία του 2015 δεν μπορεί να βοηθήσει δυστυχώς στη συγκεκριμένη περίοδο ούτε να απέτρεψε τη χρεοκοπία της Thomas Cook. Το πρόβλημα είναι ότι δεν επαρκεί η ασφαλιστική κάλυψη. Φέρετε, θυμάστε το 2000 ε, που είχε χρεοκοπήσει μια άλλη εταιρεία, δεν ε, βγάλαμε τα διδάγματα που έπρεπε. Ειδικά αυτές οι μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να έχουν μια ρεαλιστική ασφαλιστική κάλυψη. Γι' αυτό προτείνω αξιολόγηση ε, της εφαρμογής της οδηγίας αυτή για τα ταξιδιωτικά πακέτα στα κράτη-μέλη. Σε περίπτωση που χρειάζονται βελτιώσεις, να ε, τις κάνουμε για να επανέλθει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ε, στον κλάδο αυτό του τουρισμού. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βανόβερτφελτ. Αλλά α, υπήρχε η γαλάζια κάρτα του κυρίου Στεχόψκη για σας. Ε, τη δέχεστε κύριε Χάιντερ. Κύριε Στοχόφσκι, εσείς θα μιλήσετε στο ΚΑΤΣΙΑΙ όμως. Ε, είστε γεγραμμένος ως ομιλητής. Δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο με γαλάζια κάρτα. Να τα πείτε στην παρέμβασή σας αυτά. can really... Μπορεί κάποιος πραγματικά να το δει αυτό για την ολομέλειά μας, να το εξετάσει. Χρειάζεται να υπάρξει κάποια δράση και αντίδραση. Στον εσωτερικό κανονισμό προβλέπεται ότι μπορούμε να ζητήσουμε να μας απαντήσει ένα συνάδελφος. κάποιο μιλάει για κάποια πρόταση και θέλει να αλλάξει κάτι, μπορούμε να ρωτήσουμε πώς θέλει να το αλλάξει. Στο μέλλον θα είναι καλύτερο αν το σέβεστε αυτό. Μπορώ να μπω πέντε φορέ στον κατάλογο τη ομάδα μου. Αλλά αυτό αφορά τη δυνατότητα να μπορούμε να θέτουμε ερωτήσεις στους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε, λέει η Πρόεδρος, έχετε απόλυτο δίκιο ότι έχουμε καθήκον αυτή η ολομέλεια να γίνει υπόδειγμα των συζητήσεών μας. Χρειάζεται συζήτηση. Αλλά τώρα αυτή είναι μια νέα ιδέα. Θα τη διαβιβάσω στον Πρόεδρο, στους συναδέλφους στο Προεδρείο και να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας και για την έμπνευση μας την ιδέα σας. Συνεχίζουμε λοιπόν. Και πάμε στον Γιώχαν Βαν Οβερτβέλτ. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η πτώχευση της Τόμας Κουκ έχει συγκλονίσει όλη την Ευρώπη. Τώρα βρέθηκε κάποιος που θα αναλάβει την εταιρεία αυτή και θα κάνει μια καινούργια, λέει, καινοτόμα αρχή. Ε, θέλω ε, όμως να το δούμε από ένα άλλο πρίσμα αυτό το θέμα. Στην Ευρώπη έχουμε ένα πρόβλημα παραγωγικότητας. Ε, υπολείπεται η παραγωγικότητά μας και έχει φτάσει περίπου στο μηδέν. Αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην οικονομική ανάπτυξη και στα δημόσια οικονομικά. Δείχνουν επίσης ε, οι συνθήκες ότι τα χαμηλά επιτόκια ε, βοηθούν ε, στην ύπαρξη προβλημάτων γιατί δανείζονται οι εταιρείε φθηνά και συνεχίζουν να βυθίζονται στο δανεισμό και τελικά χρεοκοπούν. Ε, μήπως να το δούμε και από αυτό το πρίσμα της ε, οικονομικής αυτής δραστηριότητας. Ευχαριστώ κύριε Βανόβερτφελτ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κώστας Παπαδάκης παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ah, σχεδόν ένα μήνα μετά την κήρυξη χρεοκοπίας της thomas cook οι μεγάλοι γερμανικοί γαλλικοί βρετανικοί όμιλοι με εφόδια επιδοτήσεις προνόμια φοροαπαλλαγές διαγωνίζονται με όχημα τις θυγατρικές του χρεοκοπημένου ομίλου για το ποιος θα καρποθεί το πελατολόγιο τα περιουσιακά στοιχεία ως και τις χρονοθυρίδες της thomas cook στα βρετανικά αεροδρόμια όμως την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι τόσο της thomas cook όσο και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών στην ελλάδα με μισθούς ψίχουλα και εξαντλητικά ωράρια χωρίς ρεπό έβγαλαν τη σεζόν και σήμερα συνεχίζουν να βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα χωρίς καμιά ουσιαστική στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση και την ευρωπαϊκή ένωση επιβεβαιώνεται ότι ο δρόμος ανάπτυξης που υπηρετεί τα κέρδη των ομίλων είναι πολλαπλά επιζήμιος για τους εργαζόμενους τους αυταπασχολούμενους το λαό που και στις διακοπές του ακόμα πληρώνει το μάρμαρο. απαιτούμε τώρα να διασφαλιστούν άμεσα και χωρίς προϋποθέσεις τα πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που υφίστανται τις συνέπειες με πλήρεις αποζημιώσεις σε όσους επλήγησαν. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Άριας Ετσεβερία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. 22.000 άμεσες θέσεις εργασίας, εκατοντάδες χιλιάδες έμεσες και τόσοι καταναλωτές. Το Μάιο ήταν ε, ένα 680 ε, ε, ε, δις ζημίες μόνο για το πρώτο εξάμεινο του οικονομικού έτους. Το ΕΛΚ ζήτησε να συζητηθεί αυτό το θέμα για να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να μην έχει ξεκάθαρη φωνή για τον τουρισμό. Πράγμα που εδώ και καιρό το ζητάμε και το διατρανώνουμε. Θέλουμε ξεχωριστή συζήτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κλάδο. 4% του δικού μα ΑΕΠ και 5% των άμεσων θέσεων εργασία. Η περίπτωση Τόμας Κούκ επίση. δείχνει πόσο μεγάλη είναι ανάγκη ε, ενίσχυσης των καταναλωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Ε, δεν προστατεύονται εκείνοι που έχουν αγοράσει μόνο αεροπορικά εισιτήρια και όχι πακέτα. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Το είδε σε πρώτη ανάγνωση αυτό το Κοινοβούλιο ε, για την αναθεώρηση του κανονισμού 261 του 2004 για τα δικαιώματα των επιβατών των αερομεταφορών. Τέσσερα χρόνια τον μπλοκάρει το Συμβούλιο. Ορισμένα κράτη-μέλη, η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Δεν σας παρακολουθούν οι διερμηνείς. Μιλήστε λίγο πιο αργά. Ε, μα έχω πάρα πολλές προφορίες και πάρα πολύ λίγο χρόνο. Τι να κάνω κι εγώ. Έλεγα λοιπόν, ε, ναι, έχετε δίκιο. Τέσσερα χρόνια τον μπλοκάρει το Συμβούλιο και κάποια κράτη-μέλη έχουν χρησιμοποιήσει διάφορα επιχειρήματα ως πρόφαση για να μην προχωρήσουν. Ε, ε, φτάνουν πια οι προφάσεις. Έχει έρθει η ώρα για δράση. Α το δούμε μια ευκαιρία να γίνει μια ευρεία συζήτηση που να ασχολείται με την προστασία των καταναλωτών και έτσι να ε, έχουμε πιο γρήγορη διεκπαιρέωση των πτωχεύσεων για τις αποζημιώσεις. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα πάρει σοβαρά υπόψη γιατί είναι αδύναμη απέναντι σε τέτοιε περιπτώσει οι καταναλωτέ και οι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει απέναντι σε χρεοκοπίε που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί ή τουλάχιστον να είχαν μετριαστεί. Ναι, εντάξει, έχετε πολλέ πληροφορίε να δώσετε, λέει η Πρόεδρο, αλλά ε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε καλύτερα, να πείτε λιγότερα την άλλη φορά και λίγο πιο αργά. Εντάξει, ε, σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μαλτονάδο Λόπεθ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητούμε και στις 23 του μηνός μάθαμε ότι πτώχευσε η Τόμας Κουκ είναι βρετανική εταιρεία, πολύ σημαντική στον τουριστικό κλάδο, που είναι θεμελιώδης για μια χώρα όπως η Ισπανία, η χώρα μου. Είναι πάρα πολλοί τουρίστες που επλήγησαν και πάρα πολλοί ξενοδόχοι. Ε, θα ήθελα όμως να σταθώ στους καταναλωτές. Θα πρέπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίζουμε το δικαίωμα στους πολίτες να καλύπτονται με εγγυήσει όταν αγοράζουν πακέτα διακοπών από tour operators. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τα ξέρει αυτά και το Συμβούλιο, να διδαχθούμε από αυτή την πτώχευση για να μην επαναληφθούν στο μέλλον τέτοια φαινόμενα. Και θα πρέπει επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα εξασφαλίσει να έχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να δίνουμε λύσει στου καταναλωτέ που πλήττονται ε, είναι η οδηγία του 2015 που ε, ισχύει ήδη. Ε, οι καταναλωτές είναι σημαντικό κινητήριο ε, και ελαττήριο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Σάσκουν Μπιλπάου Παραντίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η κρίση της Thomas Cook είναι νέα ευκαιρία για μας για να δείξουμε στους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα στους Βρετανούς ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στιβαρή η νομοθεσία μας και πλήρης για την προστασία των επιβατών και των τουριστών. Θα πρέπει να αποζημιώσουμε τις 600.000 ε, ενεχομένους και να δούμε ε, τι γίνεται με τα Κανάρια νησιά και τις Βαλεαρίδες που ε, είχαν εκατοντάδες χιλιάδες κρατήσεις που τώρα είναι στον αέρα. Επίσης υπάρχει το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και θα πρέπει να καλυφθούν οι απολυμένοι εργαζόμενοι και να καλυφθούν και εκείνοι που θέλουν να εργαστούν και στην ψηφιοποίηση και στις προσωπικές προσφορές. Έχουμε ευκαιρία τώρα να είναι ελκυστικό ο τουρισμό μα. Θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μα. Γιατί αυτό το χρονικό ενό προαναγγελθέντο θανάτου ήταν ε, γνωστό. Ε, γιατί ε, λέγαμε ψέματα στον ασθενή για την κατάστασή του. Ελπίζω επιτέλους να δείξει αυτό σε όσους είναι υπέρ του Brexit τι σημαίνει να είσαι μέλος Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σα τονίσω ότι πολλοί ομιλητέ ε, μιλούν πάρα πολύ γρήγορα και δεν σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Το ξέρω ότι υπάρχει ένα κουμπί, πολύ συχνά το λέω αυτό στους Ισπανούς, δεν ξέρω, μήπως εσείς Ισπανοί ε, μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα και βάζετε πάρα πολλές προφορίες σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Ε, λοιπόν, σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Ε, μιλάτε λίγο πιο αργά, γιατί έτσι το μήνυμά σας θα μεταφέρετε καλύτερα. Η κυρία Ζουλή Λεσόντο, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πτώχευση του ε, Διεθνού Ομίλου Τόμας Κουκ στι 23 Σεπτεμβρίου δημιούργησε ένα τσουνάμι στον τουριστικό κλάδο. Στη Γαλλία, ε, οι 180.000 ε, εργαζόμενοι δεν ξέρουν τι θα απογίνουν. Όλο ο κόσμο ε, ξέρει πόσο σημαντική ήταν η βαρύτητα τη εταιρεία αυτή για τον τουριστικό κλάδο και ξέρουμε ότι αυτό θα έχει προεκτάσει και με όσα συμβαίνουν με τον Brexit. Αυτό όμω που δεν λέει κανεί είναι ότι η πτώχευση τη Thomas Cook ήταν κάτι που το ήθελαν ε, οι κερδοσκόποι, οι ασφαλιστικέ εταιρείε και τα ε, και τα fans που ήθελαν να ε, ε, προχεύσει γιατί δεν υπήρχε ασφάλεια, για να πάρουν την ασφάλεια ε, της εταιρείας αυτής. Όμως βάσει ενός καθηγητή οικονομίας υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο και παραθέτω. Μια εταιρεία μπορεί να πτωχεύσει γιατί απλώς ένας κάτοχος των ε, ψευδοσουάπ μπορεί να ε, πάει στη δικαιοσύνη και να οδηγήσει σε ένα βάγιο τη διάσωσή της. Είναι λοιπόν ένα διεθνές σκάνδαλο η Thomas Cook και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το χρηματοοικονομικό κόσμο που αρχίζει να τα χάνει τελείω και να ε, αγωνιστούμε κατά τη κερδοσκοπία. Αυτή η τελευταία φορά είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν μπορούμε να θυσιάζουμε του εργαζομένου ε, στα όρνεα τη ε, χρηματοοικονομική κερδοσκοπία. Θα πρέπει επιτέλου κάτι να γίνει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. καλησπέρα σας. Ε, θέλω να χαιρετήσω και τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών που παρακολουθούν ενδεχομένω αυτή τη συζήτηση. Το λόγο έχει ο κύριο Σόντζα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χρεοκόπησε ε, το Μαρκούκ και ο τουριστικός κλάδος ε, έχει πλέον να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτή, για αυτή τη χρεοκοπία αλλά θα πρέπει κανείς να δει ότι εκτός από το κόστος, μάλλον εκτός από το συμφέρον των μετόχων, το πρόβλημα είναι και το κέρδο, τα, πώς επλήγησαν οι καταναλωτές. Η κατάσταση της εταιρείας επιδεινωνόταν διαρκώς. Ήταν λοιπόν τελείως ε, ε ο τρόπος που παρουσιαζόταν ε, το πράγμα αυτό δημόσια μέχρι να πτωχεύσει η εταιρεία. Θα πρέπει λοιπόν να πω ότι έρχομαι από μια περιοχή της Πολωνίας που στηρίζεται πάρα πολύ στον τουρισμό. Το ΑΕΠ μας θα πληγεί. Θα πρέπει να βρούμε άλλες τουριστικές πρόσφορες, εναλλακτικές που πραγματικά να είναι πιο ε, ρεαλιστικές και βασισμένες ε, σε κάτι το ε, πραγματευτικό. Είναι θλιβερή η ιστορία της Thomas Cook, αλλά θα πρέπει στο Ευρωκοινοβούλιο να ε, κάνουμε μια εξάντε ανάλυση για τέτοιες ανάλογες επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε και τώρα η κυρία Μπούλ έχει το λόγο, Μην εγγεγραμμένη. Thank Ο κύριος Μπούλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εργάζονται μόνο και μόνο για να έχουν ένα κεραμίδι από το κεφάλι του και να έχουν μια ε, σχετική ασφάλεια για τα παιδιά του. Οι αιτήσει διακοπέ είναι κάτι για το οποίο κάνουν οικονομίε όλο τον χρόνο οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό λοιπόν αισθάνομαι τρομερή συμπόνια για του ανθρώπου αυτού που καταστράφηκαν οι διακοπέ του από την κατάρρευση τη Thomas Cook. Ήταν μια τεράστια επιχείρηση με 22.000 εργαζομένου και 19 εκατομμύρια ε, πελάτε. Όμω χρεοκόπησε διότι δεν ε, συγχρονιζόταν και είχε πολύ πολύ κακή διαχείριση των οικονομικών τη. Δεν ήταν ε, κακό το, καλό το Διοικητικό Συμβούλιο και ο τρόπο που οι διευθυντέ αμείβονταν με υπέρογκα μπόνου. Είναι εκατοντάδε χιλιάδε, 178.000 οι ε, τουρίστε που μπλοκαρίστηκαν σε όλο τον κόσμο, ξέμειναν στι χώρε που ήταν και αυτό θα κοστίσει μόνο στο Βρετανικό κράτο εκατομμύρια βρετανικέ λίρε. Αλλά γιατί το συζητάμε αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν είναι και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση μια περίπτωση που χώνει τη μύτη τη σε αυτή τη την ιστορία. Διότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ανακατευτεί, δεν μπορεί να πει στο Βρετανό φορολογούμενο να λάβει να πληρώσει τα σπασμένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσω θέλει να βάλει και λίγο χρήμα πίσω από αυτά που κάθεται και υπόσχεται. Διότι κάτι θα πρέπει να γίνει για να αποζημιωθούν όλοι αυτοί. Σα ευχαριστούμε. Κύριε Μπούλ και τώρα ο Λούτκεν. Ε, madame la Commissaire, Κύριε Επίτροπε. Εδώ μιλάμε για ένα μύθο, τον Τόμα Κουκ. Επιστώσαμε ότι είχε συνέπειε σε πολλέ χώρε όσον αφορά την απασχόληση κυρίω και στη χώρα μου το Βέλγιο. 500 άτομα περίπου επλήγησαν. Είχε συνέπειε και του ταξιδιώτε και για του εργαζομένου. Θα πρέπει εντάχει να κινηθούμε μέσω μακροπρόθεσμα εμπρότη, όπω υπογραμμίσατε, κυρία Επίτροπε. Είναι σημαντικό όλα τα μέσα, τα οικονομικά να χρησιμοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο και γρήγορα όσον αφορά τη διαχείριση των συνεπειών της χρεοκοπίας, ε, κυρίως ή ε, στο μέσο των διευθυντικών ταμείων, το κοινωνικό ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής, την παγκοσμιοποίηση ίσως μας συμμετάσχουν, αλλά γρήγορα. Διότι οι οικογένειες περιμένουν ε, απάντηση για το μέλλον τους και τι εργασίε του. Και οι κοινωνικοί εταίροι είναι σημαντικό και εκπρόσωποι των εργαζομένων που επλήγησαν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα στου εθνικού κανόνε, κυρίω αφορά τη διαχείριση των συνεπειών αυτή τη χρεοκοπία, αλλά και γενικότερα και στον τομέα του τουρισμού να συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι μόνιμα και διαθρωμένα για τη θέσπιση νέων κανόνων για την μετώπιση αυτού του είδους ε, γεγονότων στο μέλλον. Και πάνω απ' όλα στο τέλος, να πω, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι πεπισμένο ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή αρμοδιότητα πολύ μεγαλύτερη στον τουρισμό. Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Έχει αντίκτυπο για πολλά κράτη-μέλη, για πολλού ανθρώπου, πολλέ οικογένειε, την απασχόληση για την ανάπτυξη και την χρήση ε, των διαφόρων προορισμών. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να κινηθεί η Ευρώπη με ιδίου πόρου στον τομέα του τουρισμού για να αντιμετωπιστούν τέτοια γεγονότα στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η χρεοκοπία της Thomas Cook είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τον τουρισμό σε όλη την Ευρώπη. Ακριβώς για το λόγο αυτό χαίρομαι που το Κοινοβούλιο συζητάει αυτό το ψήφισμα, το οποίο δεν αντανακλά μόνο την ανησυχία όλων αυτών των πληγέντων, αλλά καλεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει με τρόπο συντονισμένο και ταχύ σε μελλοντικέ τέτοιε περιπτώσεις, όπως έκανε η κυβέρνηση της περιφέρειάς μου, συντονισμένα, όχι όπως είπε η κυρία Σταράς με την Ισπανική κυβέρνηση στις Βαλεαρίδες. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι ε, οι εργαζόμενοι επλήγησαν πάρα πολύ, οι εργαζόμενοι του κλάδου. Μια τέτοια πτώχευση σημαίνει ε, ότι οι εργαζόμενοι είναι ε, οι πιο ευάλωτοι. Έχουν τα χέρια τους δεμένα. Ένας εργαζόμενος εξαρτάται απολύτως από το μισθό του και αν ή αν χρεοκοπήσει η εταιρεία του ή αν του ε, τερματίσουν τη σύμβαση προώρα, είναι δραματικές οι συνέπειες. Δεν τα βγάζουν πέρα μέχρι το τέλος του μήνα το κείμενο του ψηφίσματος θα πρέπει να καταλαβαίνει πόσο ευάλωτοι είναι οι εργαζόμενοι για να ε, ενισχυθεί η συμμετοχή τους στη διαδικασία τέτοιων πτωχευτικών ε, καταστάσεων. Μόνο με συνεργασία και συντονισμό θα έχουμε πιο ε, πολύ δικαιοσύνη για τους εργαζομένους και καλύτερη οικονομική ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ η Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ρίκε από την ομάδα Ρινιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η πτώχευση της Thomas Cook προκύπτει από την κακοδιαχείριση από την κακή εξάπλωση και ε, άνοδο τη εταιρεία, αλλά κυρίω ότι δεν εξυγχρονίστηκε η εταιρεία χρησιμοποιώντα τη ψηφιοποίηση για τι υπηρεσίε τη. Και οι πελάτε αλλάζουν τι συνηθίε του. Ε, δεν θέλουν να αγοράζουν απευθεία υπηρεσίε, ε, μάλλον αγοράζουν απευθεία τι ξενοδοχειακέ υπηρεσίε και ό,τι χρειάζονται για τα τουριστικά του ταξίδια και δεν περνάνε πλέον από κάποιο μεσάζοντα. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη. 300 εκατομμύρια ζητούσε ε, η εταιρεία για να σωθεί, 10 δι έμεσε απώλειες. Δυστυχώς δεν μπορούσε να λάβει μέτρα για να σωθεί και να προφυλαχθεί. Όμω ο τομέα αυτό που είναι εγγεγραμμένο και στη συνθήκη, το 10% του ΕΕ τη Ένωση, που είναι σημαντικό πυλώνα για πολλέ ευάλωτε και ευπαθεί περιοχέ, περιφερειακέ και εξόχω απόκεντρε, είναι σημαντικό να υποστηριχθεί από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να είναι πάντοτε ο ουραγό των κοινοβουλευτικών μα εργασιών. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Τέναντ, μη εγγεγραμμένος. Παρακαλώ να παραμείνετε στο ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ιδρύθηκε το 1841. Είναι ο πιο παλιό το γραφείο στον κόσμο το Κουκ. Και ήταν μεγάλη επιτυχία βρετανική κατά παρελθόν, Όπω και άλλε επιχειρήσει τελικά κατέρευσε. Διότι χρησιμοποίησαν για τι κρατήσει του οι άνθρωποι το διαδίκτυο. Αυτό που ήταν φρικτό ήταν ότι οι γενικοί διευθυντέ πήραν 47 εκατομμύρια λίρες σε μπόνους αμοιβέ τα τελευταία 10 χρόνια και τελικά κατηγόρησαν την αβεβαιότητα ε, του Brexit για την κατάρρευση. Προπαγάνδα κατά του Brexit. Τα ΜΜΕ που είναι υπέρ του Remain το πρόθεσαν αυτό. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Οικονομικά ε, αναλφάβητοι προσπιστές του Remain, του εργατικού κόμματο, είπαν ότι έπρεπε να σώσει η Βρετανική κυβέρνηση τον Τόμα Κουκ. Και δεν κατάλαβαν ότι ακόμα και αν οι βουλευτέ ήθελαν να το κάνουν αυτό, ο, οι κανόνε περί ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα παρεμπόδιζαν τέτοια παρέμβαση κυβερνητική. Είναι ένα τμήμα του προβλήματο η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ένα τμήμα τη λύση. Αυτό αποδεικνύει η υπόθεση. Ευχαριστώ. Σας ερωτώ κύριε Τέναντ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Yeah. Κύριε Στοχόφσκι. Λοιπόν, προσπαθήστε να εξηγήσετε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για την κατάρρευση, για τη χροκοπία της Τόμας Κούκ που μας το εξηγήσετε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς να προειδοποιήσουμε τους πολίτες σας να μην ταξιδεύουν να πάνε στην Αίγυπτο και αλλού με την Τόμας Κούκ. Η δική σας κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία τους προειδοποίησε από το να, μην πάνε σε αυτούς τους προορισμούς. Είναι ευθύνη της κυβέρνησής σας να τους βοηθήσει, να τους προειδοποιήσει, δεν νομίζετε. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για την απάντηση. απάντηση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ είπα ότι ακόμα και αν η Βρετανική κυβέρνηση, το Βρετανικό Κοινοβούλιο ήθελε να σώσει την Τόμας Κουκ, δεν θα μπορούσε. Γιατί διότι υπάρχει νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ενώση για την κρατική ενίσχυση από τα παγόρευα. Αυτό θέλω να πω. Τι προσπαθείτε να κάνετε, να αντιστρέψετε το επιχείρημα και να πρέπει να καταλάβετε ποια είναι η νομοθεσία σα. Ότι λόγω τη νομοθεσία Ευρωπαϊκή δεν, δεν θα μπορούσε να σώσει η Βρετανική κυβέρνηση το Μασκούκ. Ευχαριστούμε. Και τώρα Warborn για το ΕΛΚ. Κύριε Warborn, Ευχαριστώ. Χρειαζόμαστε κάποια δράση τώρα να ενισχύσουμε το επιχειρηματικό κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στον τομέα του τουρισμού και των μεταφορών. 12 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που εργάζονται στον τουριστικό τομέα και ένα στους πέντε στους νέους εργάζεται στον τουρισμό. Βέβαια, η χρεοκοπία των μεγάλων επιχειρήσεων δημιουργεί τσουνάμι, κύματα που πλήττουν μικρές εταιρείε, ξενοδοχεία, εταιρείε ταξί, μικρά ξενοδοχεία μικρές εταιρείες οι οποίες είναι οι πιο ευάλωτες ακόμα και αν τα μεγάλα προβλήματα ξεκινάνε τι μεγάλε εταιρείε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εστιαστεί επί τη βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα Ευρώπη στον τομέα. Το επιχειρηματικό κλίμα στην Ευρώπη πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με σήμερα, πάνω απ' όλα για τις μικρές επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουμε σε σημαντικές υποδομές ε, που, που ενώνει την Ευρώπη υποδομή. Πρέπει να μειωθεί το διοικητικό άχθος και η γραφειοκρατία για τις μικρές εταιρείες και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ενιαία αγορά είναι πραγματικά ολοκληρωμένη. Από εμά εξαρτάται, από εμά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό και κυρίω εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσουμε ότι θα εργαστούμε σκληρά, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Η χρεοκοπία τη Τόμα Κούκ είναι απλώ ένα σύμπτωμα ενό προβλήματο που έχει πολύ βαθύτερε ρίζε όσον αφορά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ελπίζω ότι θα πρέπει να ενώσετε τις δυνάμεις σας μαζί μου, να έρθετε μαζί μου και τα θέματα των επιχειρήσεων να έχουν προτεραιότητα στις, ε, στα προγράμματα που συζητάμε. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ούχελη. Παρακαλώ. Σοσιαλιστές και Δημοκρατές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Μιλάμε εδώ για μια σημαντική υπόθεση χρεοκοπίας, μια σημαντική εταιρεία. Βεβαίως ήταν καταστροφικές οι συνέπειες και σίγουρα Εδώ έχουμε 27 εκατομμύρια ανθρώπους που εργάζονται στον τουριστικό κλάδο στην Ευρώπη. Είναι μια από τις χειρότερες καταστροφές, λοιπόν, τις χειρότερες οικονομικές καταστροφές των τελευταίων ετών. Ήθελα λοιπόν να απευθύνω την ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είστε ε, ο σημαντικότερος εταίρος ε, για μας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε για τον κλάδο αυτό που μας έφερε μόνο πέρσι 25 εκατομμύρια τουρίστες και ακόμα περισσότερα διεθνώς. Ο κλάδος έχει πάρει διαστάσεις παγκόσμιες και εμβέλεια διεθνή. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια ευρωπαϊκή προσέγγιση τι θα κάνει η πολιτική πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έχει σκεφτεί καθόλου τον κλάδο του τουρισμού και δεν το είπε καθόλου αυτό στις ομιλίες ω τώρα. Ακριβώ λοιπόν αυτή η υπόθεση δείχνει πόσο σημαντικό είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε μια ισχυρότερη τουριστική πολιτική. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Νάχταγκαλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι εδώ γιατί ένας ε, Γερμανός συνάδελφος ξέμεινε με το τρένο. Όπως έχουν ξεμείνει ε, τόσες χιλιάδες τουρίστες ε, με την Τόμας Κουκ. Και τώρα έχει backup εμένα ο συνάδελφος. Ε, στην επόμενη πτώχευση τι θα κάνουμε. Θα πρέπει ο επιβάτης και ο ταξιδιώτης να είναι καλύτερα ενημερωμένος και ταχύτερα ενημερωμένος. Να υπάρχει σαφήνεια και ασφάλεια για το τι είναι ασφαλισμένο και τι δεν είναι και πολύ γρήγορα να μπορεί να επαναπατριστεί από τις διακοπές του. Ζητώ λοιπόν ένα σύστημα εθνικό ασφαλίσεων για να βεβαιωθούμε ότι κανένας τουλάχιστον τώρα τα Χριστούγεννα να μην ξεμείνει στον τόπο των διακοπών του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Ντεχόφσκι για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή από μόνη τη είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Οι Βρετανοί συνάδελφοι βάζουν τι φωνές ε, ότι είναι μόνο δικό τους πρόβλημα. Μα αυτό είναι γελίο, διότι εργαζόμενοι της Thomas Cook εξυπηρετούσαν τουρίστες παγκοσμίω. Είναι η μεγαλύτερο ταξιδιωτικό πρακτορείο, η μεγαλύτερη τουριστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1841. Αυτή πτώχευσε. Και αυτό θα πλήξει πολλέ άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του πολίτε του. Ο τουρισμό δεν αφορά μόνο, μόνο όσου ταξιδεύουν. Οι καταναλωτέ που αγοράζαν πακέτα ε, ταξιδιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από άλλε χώρε, όλοι θα την πληρώσουν. Αυτοί που δούλευαν επίση ε, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, όλοι αυτοί που μέχρι σήμερα θα μείνουν και στο και θα μείνουν απλήρωτε. Αυτά τα θέματα λοιπόν πρέπει να δούμε και να σκεφτούν οι Βρετανοί συνάδελφοι τι σφάλμα έκαναν όταν ψήφισαν υπέρ του Brexit. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε εργαλεία, είχαμε προγράμματα για να αντιμετωπίσουμε την αντιγεία αυτών που ε, ε, έμειναν χωρίς δουλειά. Θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε πολύ καλύτερα ακόμη και να επανεπατριστούν. Ευχαριστούμε πολύ ε, κυρία Γκραπίνα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν ήδη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Πρέπει να την συζητήσουμε. Είναι η χρεοκοπία μιας εταιρείας 178 ετών με εκατοντάδες χιλιάδες ε, υπαλλήλους και πελάτες. Θα πρέπει όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί τον τουριστικό κλάδο λίγο σοβαρότερα. Είναι ένα σοβαρότατο ποσοστό του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ε, κοινή. Πρέπει να έχουμε μια δημοσιονομική γραμμή. Πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη δράση. Διότι ακόμα και αν πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία, δεν καταλαβαίνω δεν θα πρέπει να μελετήσουμε αυτή την πτώχευση. Λέτε δεν είχε ασφάλεια η εταιρεία αυτή. Δεν μπορούμε όμω να αφήσουμε του εργαζομένου στην τύχη του, ούτε του πελάτε, ούτε του τουρίστε είναι όλοι σε σύγχυση. Δεν ξέρουν ε, τι θα του συμβεί, γιατί η εταιρεία έχει κακοδιαχείριση. Έχουμε ένα μισή δις ευρώ ε, ποσών που δεν έχουν επιστραφεί. Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν. Θα πρέπει να στηρίξουμε τους επιβάτες, τους τουρίστες, τους πελάτες, τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τέτοιες τραγωδίες να επαναλαμβάνονται με τόσο παραδοσιακές τόσο παλιές εταιρείε, τη δεύτερη τουριστική εταιρεία του κόσμου. Ευχαριστούμε. Και τώρα ε, από την Ρινιού ο κύριος Βόντεν. Κυρία Βόντεν, η κατάρρευση της Thomas Cook είναι μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες ε, της εποχής μας. 21.000 θέσεις χάθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι άλλες τόσες χιλιάδες θα υποφέρουν στην Ευρώπη. Δηλαδή όσοι έμειναν άνεργοι και οι οικογένειές τους. Οι υλικέ καταστροφές και ε, η καταστροφή της διαβίωσης των εργαζομένων και των ε, υπεργολάβονται στο Μασκούκ είναι τεράστια. Ε, δεν φτάνει όμω εδώ η ωραία, τα ωραία λόγια συμπάθεια. Ε, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν να πληρώσουν τον νίκη του. Πρέπει να του προσφέρουμε επιμόρφωση και κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν αλλού. Πρέπει να υποστηρίξουμε όσου θέλουν να δημιουργήσουν νέε επιχειρήσει και να δώσουν ε, νέε θέσει εργασία για να αντικαταστήσουν αυτέ που χάθηκαν. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να καταραίει από τη μια μέρα στην άλλη έτσι, αφήνοντα τον κόσμο να μένει μπλοκαρισμένο σε διάφορα μέρη του κόσμου και δημιουργώντα τέτοια δυσφορία. Συνάδελφοι, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά για να βεβαιωθούμε ότι καμία ευρωπαϊκή εταιρεία δεν έρχεται αντιμέτωπη με την ε, περίπτωση να μην έχει αρκετά κινήτρα επειδή δεν ε, ε, ψηφιοποιήθηκε αρκετά. Ο κόσμο αλλάζει στην Κορνουάλη. Ένα στου πέντε, την περιφέρεια, ένα στου πέντε εργάζεται στον τουρισμό με Airbnb ε, που είναι ε, με το Airbnb να είναι μια σαφής πρόκληση για τις κλασικές εταιρείες. Πρέπει να δούμε λοιπόν το πώς αλλάζει αυτός ο τουριστικός κλάδος παντού προσπατεύοντας τους ωραίους προορισμούς της Ευρώπης από την καταστροφή τους λόγω του μαζικού και ανεξέλεγκτου τουρισμού. Ευχαριστούμε ο κύριος Κάνεφ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε σαν εκπρόσωπος μιας χώρας για την οποία ο τουρισμός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά το ΑΕΠ και την απασχόληση, υποστηρίζω όλα τα μέτρα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οικογένειες, τις τοπικές ε, επιχειρήσεις που αναμειγνύονται στον τομέα του τουρισμού. Κάποιες πτυχές του προβλήματος υποτιμήθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ άλλων. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση μεριδίου της αγοράς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε τελικά γίνεται πολύ μεγάλη εταιρεία για να χρεοκοπήσει. Too big to fail. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει επικίνδυνη κάθετη συγκέντρωση των τουριστικών υπηρεσιών κάτι που επηρεάζει τους κανόνες περί ανταγωνιστικότητας και δεν θεωρούμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα μοντέλο οριζόντιας και κάθετης συγκέντρωσης υπηρεσιών που επηρεάζουν όχι μόνο τους ε, καταναλωτές αλλά επηρεάζονται αρνητικά και οι μικρές επιχειρήσεις και οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε. Η ε, Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Βέντ, παρακαλώ. Η κατάρρευση της Thomas Cook... η Τζόρτζια Μπράουνινγκ φόρεσε μια στολή και πήγε στο μπαρ το τοπικό με συναδέλφους για να βοηθήσει τους τουρίστες που είχαν ε, ξεμείνει. Δεν πληρώνονταν, αλλά δεν ήθελαν να αφήσουν έτσι τους εργαζομένους. Είχαν μια καλή δουλειά που κατέρευσε μια νυχτή. Αυτή η κατάρρευση λόγω μεγέθους είναι μοναδική, αλλά όχι λόγω μορφής και τύπου. Πολύ συχνά, όπως κατά παρελθόν, τελικά ε, τα ίδια θύματα είχαμε. Ο Φρανκ Χάουζερ, ο πρόεδρος μπορεί να την αράξει και να απολαμβάνει τα εκατομμύρια που πήρε από μπόνουση. Ενώ χιλιάδες έχασαν τη θέση απασχόλησης και οικογένειε οικογένειες πολεμάνε να πληρώσουν λογαριασμού. Η διοίκηση γνώριζε ότι η κατάσταση ήταν επικίνδυνη. Η Τζόρτζια και οι συνάδελφοι που εργαζόταν τον Τόμα Κούκ το ήξεραν. Όλη η Ευρώπη πρέπει να μάθει από την κατάρρευση στο Μασκούκ. Ο κοινωνικό διάλογο μεταξύ διοίκηση και εργαζομένων θα πρέπει να ενισχυθεί στην Ευρώπη, ούτω ώστε κανεί να μην κολλάει, όπω είδαμε αυτό που έπαθαν οι ταξιδιώτε σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Κύριε Καρβάλιο. Πρόεδρε, πρόεδρε, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά είναι αποφασιστική σημασία και χρειάζεται να προστατεύονται ε, σοβαρά τα δικαιώματά τους. Είναι τεράστια σημασία το τουριστικό κλάδο για την ευρωπαϊκή εσωτερική ε, αγορά και ενιαία αγορά μάλλον και σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη. Η πτώχευση της Thomas Cook θα πλήξει όχι μόνο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών αλλά και τις τουριστικές περιοχές όπως το Αλγκάρβε ή το Αλεντέζου. Εδώ λοιπόν είναι ε, ολόκληρε οικογένειε, επιχειρήσει, ε, τοπικέ οικονομίε που πλήττονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι κανόνε που ισχύουν εφαρμόζονται σωστά, ότι τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα εκταμιεύονται και χρησιμοποιούνται και ότι προβλέπονται πρόσθετα μέτρα. Μέτρα που θα επιτρέψουν να προστατευτούν οι πελάτε των αερομεταφορέων ώστε οι καταναλωτέ αμέσω να αποζημιωθούν για τη ζημιά που υπέστησαν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την εύρωστη λειτουργία της, ε, την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και το ε, επίπεδο προστασίας των καταναλωτών το οποίο έχουμε θέσει ως στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Κέτον Ντάλεγκ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ε, Τόμας Κουκ, το βρετανικό μοντέλο, κήρυξε την πέκευση του το Σεπτέμβριο, είναι χιλιάδε αυτοί που έμειναν μπλοκαρισμένοι και 22.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 9.000 στον ΕΒ έμειναν άνεργοι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η ε, Τόμα Κουκ πτώχευσε λόγω κακοδιαχείριση. Όμω η αρχή πολιτική αεροπορία πρέπει να επενεθεί για τι προσπάθειέ τη να φέρει τον κόσμο στη χώρα του, χάρη στην οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών. Η κυβέρνησή μα δεν έκανε όμω τίποτα για να προστατεύσει του καταναλωτέ, του εργαζομένου ή του φορολογουμένου. Ίσο, μάλιστα κάθισαν τα χέρια σταυρωμένα και άφησαν την εταιρεία να πτωχεύσει. Όχι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, όπως ακούσαμε να λένε κάποιοι, αλλά γιατί δεν το ήθελαν. Ε, ήταν ε, πολύ καλές ειδήσει ότι ε, η Hayes Travel μπήκε στην όλη ιστορία, επειδή είναι μια επιτυχημένη τουριστική ιστορία και βοήθησε να επιστρέψουν στη χώρα μας οι διάφοροι ταξιδιώτες. Τώρα, το, αυτό που ευαγγελίζεται το Brexit του Τζόνσον δεν θα φέρει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας και να μην αφήσουμε να καταστραφούν ούτε να ε, καταστρέφουμε εμείς οι ίδιοι, ε, αλλού τις ευθύνες όπως ακούσαμε να γίνεται απόψε. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Σκίτενταλ από το ΕΛΚ. Ε, Κυρία Σκίτενταλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Τόμας Κουκ είχε μεγάλε συνέπειες για την απασχόληση στην Ήπειρό μας. Αλλά τέτοια πλήγματα ε, έχει δεχτεί ο τουριστικός κλάδος και προηγουμένως και μπορεί να δεχτεί κι άλλα, ε, εάν σκεφτούμε και τι συζητήσει που γίνονται σε σχέση με τις κλιματικέ αλλαγές. Η UBS έχει εντοπίσει ότι αυτή η λεγόμενη ντροπή, η ενοχή τη ε, πτήση και των αερομεταφορών έχει οδηγήσει πολύ κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματάει να ταξιδεύει αεροπορικό. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μα και αυτή την αλλαγή. Από την άλλη, η αεροπορία έχει γίνει ολένα και περισσότερο φιλική προ το κλίμα και το περιβάλλον και βεβαίω ε, αυτό έχει να κάνει και με τι τεχνολογικέ εξελίξει. Εάν θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε τον τουρισμό, Πρέπει να σκεφτούμε αυτές τις ε, καταστάσεις, τα νέα φαινόμενα όπως την ενοχή ε, του να πετάει κανείς και πώς μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για να έχουμε βελτιώσεις, βήματα πρόοδου και με τεχνολογική υποστήριξη για να διασφαλίσουμε θέσεις εργασία και απασχόληση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκαρθία Μουνιός από τους Σοσιαλιστές και Δημοκρατές. Η κυρία Γκαρσία Μουνιάς, ο τουρισμός είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας ε, και έχει πολύ μεγάλη δυναμική στην Ισπανία. Η χρεοκοπία τη Thomas Cook προκάλεσε μια κρίση που έπληξε πολλούς τομείς, επαγγέλματα και υπηρεσίε, κυρίως στις νησιωτικέ περιοχές, όπου η προσβασιμότητα και η συνδεσιμότητα είναι ζωτική σημασία. Ο αντίκτυπος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν τεράστιο. Η απώλεια της συνδεσιμότητας και πολλών θέσεων εργασία. δηλώνουν ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν κοινέ προκλήσεις και στον τουρισμό και μας δείχνει την αναγκαιότητα να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό και να δημιουργηθούν μηχανισμοί πρόληψης και για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, να ε, προστατεύσουμε την ασφάλεια των επιβατών. Γι' αυτό ζητάμε από την Κομισιόν να λάβει υπόψη την ε, πρόταση του Κοινοβουλίου για να δημιουργήσει μία γραμμή προπολογισμού για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, να καταρτήσει νομοθεσία για να ορίσει ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση χρεοκοπία. και περιμένουμε και το κοινωνικό πακέτο του τομέα τη αεροπορία. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα για να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σούλτσε από το ΕΛΚ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όταν ε, χρεοκοπεί το δεύτερο μεγαλύτερο ταξιδιωτικό πρακτορείο του κόσμου, αυτό έχει συνέπειες και στους εργαζόμενους και στους χιλιάδες ε, πελάτες. Άκουσα πολύ κριτική σήμερα στην οδηγία περί ε, μαζικών ταξιδιών. Μα χάρη σε αυτήν υπάρχει κάποια αρρύθμιση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Έχουμε χώρες όπως ε, το Ενωμένο Βασίλειο, όπου τα πληρώνει στο τέλος όλα ο φορολογούμενος, άλλες όπως στη Γερμανία υπάρχει μια ασφάλιση τα οποία δεν, η οποία δεν επαρκεί όμως. Έχουμε 110 εκατομμύρια ασφαλισμένα, οι ζημιές είναι τριπλάσιες. Οπότε θα πρέπει να ξαναδούμε την οδηγία αλλά κυρίως την εφαρμογή της στα κράτη-μέλη. Να επενέσω την Κομισιόν για την γρήγορη έκρηση της ε, χρηματοδότησης στην Κόντορ, μια εταιρεία στη Γερμανία η οποία δεν έφταιγε για την ε, χρεοκοπία και έτσι προστατεύτηκαν ε, χιλιάδες θέσεις εργασίας και χιλιάδες τουρίστες οι οποίες μπόρεσαν να πάνε στις διακοπές τους και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν. Σας ε, ευχαριστώ. Αντάμοβιτς για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ως καθηγήτρια πανεπιστημίου στο δίκαιο του τουρισμού και των μεταφορών στην Πολωνία και στον κόσμο εδώ και χρόνια υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που προστατεύει τους ε, πελάτες ε, των ε, τουριστικών επιχειρήσεων χρεοκοπία της ε, Thomas Cook ε, μας δίνει ένα νέο δίδαγμα σε ό,τι αφορά τα νέα εργαλεία που πρέπει να υπάρχουν για την προστασία των πελατών του κλάδου του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλάμε για διασυνοριακές υπηρεσίες. Η οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια χέρι της ε, υποστήριξής μου, αλλά ως νομοθέτες ε, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην προστασία των καταναλωτών και των μεταφορέων, αλλά και των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού. Είναι επίσης σημαντικό να παρέχουμε προστασία και στους ταξιδιώτες. Η κυρία Σπυράκη για το ΕΛΚ. Ε, κυρία Επίτροπε, η Ελλάδα είναι η δεύτερη αγορά της Thomas Cook μετά την Ισπανία. Η εταιρεία στην Ελλάδα διέθετε 68 ξενοδοχεία, το 12% των ελληνικών ξενοδοχείων δηλαδή, κυρίως σε 8 νησιά και έφερνε 3 εκατομμύρια τουρίστες σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου ερευνών και προβλέψεων του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου της ελλάδας το δύο χιλιάδες είκοσι εξαιτίας της κατάρρευσης της thomas cook θα έχουμε απώλεια εσόδων δύο πέντε δισεκατομμύρια ευρώ η κατάρρευση αυτή είναι πλέον συστημικός κίνδυνος για τον ελληνικό τουρισμό κάποιοι μιλάνε για τη lehman brothers του ελληνικού τουρισμού. δεδομένου ότι υπάρχει η βούληση από την πλευρά της ευρωπαϊκής ένωσης και της κομισιόν να επιτρέψει κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος και είδαμε την αρχή που έκανε η γερμανία οφείλουμε μέσω αυτού του ψηφίσματος που σήμερα συζητάμε εδώ να πάμε παρακάτω να εξετάσουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο υποστήριξης για τις οικονομίες των χωρών που πλήττονται που θα μπορούσε να περιλαμβάνει κρατικές ενισχύσεις φοροελαφρύνσεις ίσως και τη δημιουργία ενός ταμείου εγκυοδοσίας για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. κυρίως όμως θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρόταση υποδιερεύνηση ο έλεγχος αυτών των μεγάλων εταιριών που δεσπόζουν στην αγορά του τουρισμού όπως και άλλες μεγάλες εταιρείες κυρία πρόεδρε κυρία επίτροπε εάν ο ευρωπαϊκός τουρισμός θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικός θα πρέπει να χαράξει μια νέα στρατηγική προωθώντας τη μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από τους tour operators την ουσιαστική διαφοροποίηση του προϊόντος την ενίσχυση των συνεργασιών και κυρίως να δώσει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα αντί στους αριθμούς. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε ο καταλογός των ομιλητών, ενώ τώρα περνάμε στο Catch the Και καταρχήν, ε, η κυρία Ward για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Uh, Ευχαριστώ. Η κατάρρευση της Τόμας ε, Κούκ είναι τραγική και μπορεί, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Άφησε 150.000 ε, ε, τουρίστες εγκατελελειμμένους, πάρα πολλούς με παιδιά και πολλές οικογένειες εργατών που είχαν εργαστεί σκληρά για τις διακοπές τους. Η κατάρρευση θα μπορούσε να κοστίσει μέχρι και 9.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στα κεντρικά γραφεία ασχολούνταν 450 άτομα και στο αεροδρόμιο στην περιοχή μου είχαμε χιλιάδες προσωπικού ε, και 17 καταστήματα στο Μάντσεστερ που υποστηρίζονταν από, την, ε, από το συνδικάτο TSSA. Η Τόμας Κούκ λέει ότι συντηρητική, ε, η γραμματέας της συντηρητικής κυβέρνησης ε, δεν ε, μίλησε καν στους διευθυντές πριν την χρεοκοπία. Ευτυχώς οι 600.000 παραθεριστές προστατεύονταν από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ταξίδια καθώς οι συντηρητικοί προσπαθούν να μας βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπονομεύουν την προστασία των καταναλωτών. Αυτό το δίκτυ ασφαλείας ε, δεν θα υπάρχει ε, υπό την κυβέρνηση του Μπορις Τζόνσον μετά το Brexit. Σας ευχαριστώ. Φερέιρα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε η Thomas ε, Cook, ε, ε, μια τεράστια εταιρεία, έκανε να έχουμε τεράστιες απώλειες θέσεις εργασία, είχε 200 ξενοδοχεία και πάνω από 100 αεροπλάνα και οι συνέπειες μας δείχνουν την πραγματικότητα σε ένα τομέα που έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων πολυεθνικών ομίλων και υπάρχουν όμως και ένας τεράστιος

Ιστός μικρών και μεσαίων ε, επιχειρήσεων. Έχουμε ένα τομέα με πολύ μεγάλη εκμετάλλευση και χαμηλούς ε, μισθούς και ε, έχουμε, αυτό να έρχεται σε αντίθεση με τα τεράστια κέρδη των καπιταλιστών όταν εφαρμόζουν κάποιες επιζήμιες πρακτικές και από ό,τι φαίνεται άλλοι πληρώνουν το λογαριασμό. Επίσης είδαμε ότι και οι καταναλωτές βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση. Πρέπει να δράσουμε επί αυτής πραγματικότητας. Αυτή η οποία είχε μεγάλο αντίκτυπο στην Πορτογαλία, ιδίω στη Μαδέρα και στο Αλγκάρβε και ε, τελικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που ανακοινώθηκαν εδώ για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της χειροκοπίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε. Και τώρα η κυρία Τέσσερ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, η συζήτηση αυτή δείχνει πως η χρεοκοπία τη Τόμα ε, Κούκ έχει πολλές αιτίες και απαιτείται μια πολύπλευρη αντιμετώπιση και για να προλάβουμε την χρεοκοπία και εάν παρελπίδα δεν την αποφύγουμε να δούμε τις συνέπειες. Τα αποτελέσματα και τα διδάγματα θα μπουν στην έκθεσή μας ε, για την εφαρμογή του πακέτου, για την εφαρμογή της οδηγίας για τα ταξίδια. Και βεβαίως ε, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Βεβαίως η συζήτηση αυτή μας ε, έδωσε πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίε, Πολλοί από εσάς ζητήσατε συγκεκριμένες πολιτικέ για τον τουρισμό. Υπάρχει μια νέα θητεία μπροστά μα για να εξεταστεί αυτό το αίτημα και για να αξιολογήσουμε την ανάγκη ανάπτυξη μια νέα στρατηγική για τον τουρισμό στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στο ευρύτερο πλαίσιο των οριζόντιων πολιτικών. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα να επαναλάβω πω, ε, σύμφωνα με τι προτάσει τη Κομισιόν για το επόμενο ΠΔΠ, πολλά προγράμματα προβλέπουν στήριξη του τουρισμού, π.χ. τα διαρθρωτικά ταμεία, το InvestEU, το Ταμείο για την Ενιαία Αγορά, Δημιουργική Ευρώπη, ο Ορίζοντας και αυτό μας δείχνει το ότι έχει ενταχθεί ε, το θέμα του τουρισμού στις διάφορες πολιτικές και ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι λογικό καθώς ο τουρισμός είναι αλληλένδετος με άλλους κλάδους της οικονομίας. Σας ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους βουλευτές για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, η συζήτηση για το θέμα αυτό τελείωσε. Την πέμπτη θα ψηφίσουμε. Και Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Δήλωση της Κομισιόν για τον κίνδυνο του βίαιου ακροδεξιού εξτρεμισμού εν συνεχεία των πρόσφατων γεγονότων στο χάλι της Γερμανίας. Πριν περάσουμε στην συζήτηση, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην διαδικασία και HDI και στην ε, μπλε κάρτα θα πρέπει να ζητάτε το λόγο με την ε, συσκευή που έχετε μπροστά σας για τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ. Πρώτος έχει τον λόγο ο κύριος Κίνγκ, εξ ονόματος Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Μια σημαντική όσο και επίκαιρη συζήτηση απόψε. Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στο χάλε της Γερμανίας ε, υπογράμμισαν την πραγματική και αυξανόμενη απειλή του ακροδεξιού εξτρεμισμού και στη συγκεκριμένη περίπτωση αντισημιτισμού. Μια απειλή η οποία δυστυχώς ε, τονίστηκε ήδη από την ε, σφαγή αθώων στο Christchurch ε, νωρίτερα φέτος. Μετά από αυτά τα δύο γεγονότα γνωρίζω πως όλοι σκεφτόμασταν τους οικείους των θυμάτων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την απειλή και να συνεργαστούμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κράτη-μέλη για να εντείνουμε τις προσπαθίες μας για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση. Ας είμαστε σαφείς. Ο βίαιος εξτρεμισμός είναι βίαιος εξτρεμισμός. Οποιαδήποτε ιδεολογία μίσους ε, και αν έχει. Δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας. Ούτε τζιχατσμός, ούτε ακροδεξιά, ούτε ακροαριστερά ο ρατσισμός, ο αντισημιτισμός, η ξενοφοβία, ο υπερεθνικισμός είναι θεμελιωδώς αντιδημοκρατικά και αντιευρωπαϊκά. Η Τζο Κόξ, μια βουλευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν δολοφονήθηκε από έναν Βρετανό πατριώτη, την δολοφόνησε ένας ακροδεξιός τραμπούκος. Οι ευρωπαϊκές χώρες μας ανήκουν σε όλους μας. Όχι σε αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον πατριωτισμό τους για, ως δικαιολογία για δολοφονίες. Η Κομισιόν καλωσορίζει την ε, πρωτοβουλία της Προεδρίας και μάλιστα αυτό φάνηκε και στην συζήτηση του Συμβουλίου Δικαιοσύνη και Εσωτερικών στις 8 Οκτωβρίου που ενέκρινε κάποιες προτάσεις της Προεδρίας. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να στηρίξει όλα τα κράτη-μέλη και την Προεδρία και προφανώς να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάθε δυνατό τρόπο. Βεβαίω το έργο μας για την αντιμετώπιση της, ε, του βίαιου εξτρεμισμού και της ε, τρομοκρατίας καλύπτει όλες τις μορφές ε, εξτρεμισμού. Μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε εστιάσει στην τζιχαντιστική τρομοκρατία που πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα δεδομένης της φύσης της απειλής αλλά η Κομισιόν εστιάζει όλο και περισσότερο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον βίαιο ακροδεξιό εξτρεμισμό, ειδικά μέσω του δικτύου ενημέρωσης ε, για την ριζοσπαστικοποίηση που συνεργάζεται με αστυνομία, δεσμοφύλακες, ε, δασκάλους και άλλους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης. Και θεωρούμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Πρώτα απ' όλα, συμφωνούμε με όλους όσους λένε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε το περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Πριν από τρία χρόνια υπογράψαμε με τις ε, πλατφόρμας ε, έναν ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς για να αντιμετωπιστεί η ρητορική μίσους. 28% ε, του περιεχομένου αφαιρέθηκε. Και τώρα μπορώ να πω ότι έχουμε φτάσει στο 72% του περιεχομένου αυτού. Βεβαίω ο κώδικας ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους δεν έχει τελειώσει και δεν υπάρχει κάποιο σημάδι πως η δημιουργία και η κυκλοφορία του έχει μειωθεί. Η Κομισιόν και οι πλατφόρμες θα συνεχίσουν να εντείνουν την συνεργασία μας στο φόρουμ ε, του διαδικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συνεδρίασε πριν από δύο εβδομάδες και το θέμα αυτό, ακριβώς η αντιμετώπιση του βίου ακροδεξιού εξτρεμισμού, ήταν πρώτο-πρώτο στην ημερησία διάταξη. Η συνεργασία αυτή είχε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία τονίστηκαν από την γρήγορη αντίδραση των εταιριών αυτών στην επίθεση του Χάλε. Αφαιρέθηκαν οι 200 διαφορετικές παραλλαγές ε, του βίντεο και το λεγόμενο μανιφέστο, μεταξύ των οποίων και μια ηχογράφηση. εντό δύο ώρων έγιναν αυτά, οπότε καλωσορίζω την συνεργασία με τις εν λόγω Επιπλέον, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η σχετική μονάδα της Europol θα έχει τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπίζει το περιεχόμενο του βίαιου ακροδεξίου εκτρεμισμού και είμαι σίγουρος ότι θα το στηρίξετε. Η Europol αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με 350 πλατφόρμες κοινωνικών μεσών. Αλλά υπάρχουν ακόμα πλατφόρμες σήμερα που αρνούνται να συνεργαστούν με τις προσπάθειες μας για να κατέβει τρομοκρατικό περιεχόμενο μεταξύ των οποίων και ακροδεξιό. Για μένα αυτό είναι ένας λόγος ε, για τον οποίο θα πρέπει από κοινού συνομοθέτες να κινηθούμε γρήγορα στις διαπραγματεύσεις για μια ρύθμιση που θα αντιμετωπίσει το τρομοκρατικό περιεχόμενο. Πρέπει να γίνει αυτό, να πατάξουμε αυτό το δηλητήριο και να σώσουμε ζωές. Ας υπάρξουν σαφή αποτελεσματικά μέτρα για την διαγραφή αυτού του περιεχομένου, μεταξύ των οποίων και η άμεση μετάδοση τέτοιων επιθέσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία λόγου. Δεύτερον, η Κομισιόν είναι έτοιμη να στηρίξει περαιτέρω τα κράτη-μέλη και τις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση. Η απειλή ε, που αποτελεί ο ακροδεξιός εκτρεμισμός ε, υπάρχει στον προσανατολισμό του 2020 για μια συντονισμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό περιλαμβάνει το να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις και τις περιφέρειες να αναπτύξουν ε, σχέδια δράσης για να προλάβουν το φαινόμενο αυτό, μεταξύ των οποίων και με προγράμματα εξόδου. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να στηρίζει επίσης ε, δήμους και πόλεις στις προσπάθειες τους να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό υπάρξε το συνέδριο πόλης κατά της ριζοσπαστικοποίησης ε, μαζί με την Επιτροπή των Περιφερειών και επιπλέον ε, έχουμε μια πιλωτική ομάδα πόλεων που ενδιαφέρονται για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης. Τρίτον, και αυτό το, νόμισαν τα, το τόνισαν τα κράτη-μέλη στο Συμβουλίο, πρέπει να στηρίξουμε τους γείτονές μας στις προσπάθειές τους αυτές. ειδικά στα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχει το σχετικό αντιτρομοκρατικό σχέδιο, το οποίο υπογράψαμε πριν από δύο χρόνια και καλύπτει όλες τις μορφές ε, ριζοσπαστικοποίησης και βιαίου εξτρεμισμού. Για να το εφαρμόσουμε, η Κομισιόν ε, συνάπτει συγκεκριμένες συμφωνίες με όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες για να καταβοληθούν όλες οι μορφές του εξτρεμισμού. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε να προχωρούμε σε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας και τους εταίρους μας στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Τστάτλερ εκ μέρους του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας καταφέραμε να περάσουμε μία δήλωση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και έτσι δεσμεύτηκαν όλα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε μία τακτική διασφάλισης των εβραϊκών εγκαταστάσεων. Φαίνεται αυτό ότι είναι κατεπήγον. Υπήρχε τον Δεκέμβριο μία έκθεση της ε, Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πρόκειται για μια έρευνα στην οποία απάντησαν 16.000 ε, Εβραίοι, οι οποίοι εκπροσωπούν μεγάλο ποστό των Ευρωπαίων Εβραίων. Το συμπέρασμα είναι ότι νιώθουν όλο και πιο ανασφαλείς στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι έχει συμβεί μέχρι στιγμή. Προφανώ λίγα πράγματα, γιατί δεν καταφέραμε στο Γιόμ Κιπούρ μάλιστα να έχουμε μια συναγωγή, η οποία ήταν αφύλακτη και να μπορεί να περνά απ' έξω ένας άνθρωπος να σκοτώνει ε, δύο άλλους και μόνο ως εκθαύματος αποφεύχθηκε μεγαλύτερη σφαγή. Στη μέση της Γερμανίας ε, δηλαδή έχουμε πράγματα τα οποία χαράζονται στη συλλογική μνήμη όχι μόνο της εβραϊκής κοινότητας. Θα πρέπει λοιπόν να υπενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη ότι δεν αρκούν οι δηλώσεις. Τώρα θα πρέπει επιτέλους να έχουμε συγκεκριμένες πράξεις ε, Έχουμε μια συνεργασία εδώ και δεκαετίες στην Αυστρία που μπορεί να αποτελέσει νομίζω υπόδειγμα. Δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί ένα δράμα σαν το Χάλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέστερ για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κυρία Πρόεδρε, ένα αναζητή ε, τρομοκράτη ε, επιτέθηκε σε μια συναγωγή στο Χάλι και σκότωσε δύο ανθρώπου που περνούσαν τυχαία από εκεί. Οι Εβραίοι ε, ζουν σε όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια. Και στην περιοχή μου, στο Ντόρτμουντ, εξακολουθούν να υπάρχουν Εβραίοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν αντισημητικά κλισέ. Η εφημερίδα εκεί μας λέει για παρενοχλήσεις ε, που αντιμετωπίζουν διάφοροι μαθητές ε, ή κάποιος ο οποίος φορούσε μια κύπα και ζει καθημερινά τον αντισημιτισμό, ένας φοιτητή στο πανεπιστήμιο και του λένε εκεί πέρα «Έλα μωρέ, τι διαβάζεις εσύ θα περάσεις αφού είσαι Εβραίος». Και σκέφτεται το Σαββατοκύριακο εάν ε, είναι σωστό να υπογράψει με το όνομά του ένα άρθρο το οποίο αφορά το πόσους συμπαθούντες ε, βρήκε ο δολοφόνος ε, του Χάλε. Ειδικά μάλιστα εντός της αστυνομίας. Το γεγονός ότι την ημέρα του Γιώμ Κιπούρ δεν φυλασσόταν η συναγωγή είναι ένα συστημικό πρόβλημα ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν μεμονωμένος ε, δράστης ε, και οι... αυτοί οι οποίοι του όπλησαν το χέρι βρίσκονται και εδώ μέσα, παραδείγματος χάρη στα έδρανα του ΑΕΦΔ. Λοιπόν, δεν αφορά μόνο τους Εβραίους, μπορεί να μας πλήξει όλους ε, και πρόκειται για μια επίθεση κατά της δημοκρατίας στην οποία πρέπει να ανταχθούμε σήμερα ενωμένοι. Σας ευχαριστώ. Το λόγο κυρία Μπέρ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι εικόνες ε, του Χάλε και των άλλων ε, χτυπημάτων βεβαίως μας αφήνουν άναυδους. Αλλά δεν αρκεί να θρυνούμε τα θύματα. Πρέπει να φροντίσουμε ο... να μην κερδίζει έδαφος ο αντισημιτισμός στην Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο υποτιμούμε, καμιά φορά ε, είναι καλυμμένος ως ειρηνική διαμαρτυρία παραδείγματος χάρη ε, άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται διαμαρτύρονται για την πολιτική του Ισραήλ. Ε, εμφανίζεται ξανά η λέξη Εβραίος ή Γιαχούντι βρισιά. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, όλοι θεωρούν ότι υπάρχει αντισημιτισμό στην ε, χώρα του. Ναι, πράγματι δεν υπήρχε φρουρά στην συναγωγή την ημέρα του Γιώργου Κιπούρα, αλλά γιατί ε, φυλάσσονται και κινδυνεύουν περισσότερο οι συναγωγές από τι εκκλησίε και τα τζαμιά, γιατί χρειάζονται αστυνομία. Ποιο έλλειμμα υπάρχει στην κοινωνία μα έτσι ώστε ο αντισημιτισμός να εμφανίζεται. Πώς μεγαλώνουν οι νέοι, τι μαθαίνουν στα σχολεία ξεχνάμε πραγματικά την ιστορία μας μετά τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο παγκόσμιο. Τι κάνουν τα ΜΜΕ, τι κάνουμε εμείς με τα αντισημιτικά στερεότυπα, πώς αντιδρούμε σε τέτοια περιστατικά. Είναι, μας είναι πραγματικά αδιάφορο το ότι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς οι Εβραίοι και φεύγουν από την Ευρώπη. Ε, δεν επιτρέπεται, αγαπητοί συνάλφοι. Στα σχολεία θα πρέπει να διδάσκεται και το ολοκαύτωμα και η σημερινή εβραϊκή ζωή. Χρειάζεται πρόληψη. Πρέπει οι νέοι να μάθουν να αντιμετωπίζουν την ψηφιακή βία, να υπάρξουν επαφές με εβραϊκά ιδρύματα. Όλα αυτά πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο. Μόνο η αναγνώριση ότι ο αντισημιτισμός μας αφορά όλους και μας απειλεί όλους θα μας δώσει την δυνατότητα να προστατεύσουμε τις αξίες της Ευρώπης. Άρα θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε κατά του αντισημιτισμού. Είτε προέρχεται από αριστερά, είτε από δεξιά, είτε από ψεύδο λόγους. Μας απειλεί όλους, ανεξαρτήτως ε, της ιδεολογίας από την οποία προκύπτει. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε ε, και ως πολίτες και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τώρα στην κυρία Καβατσίνη εκ μέρους των Πρασίνων. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Η εικόνα αυτή παραμένει στα μυαλά μας. Ένας ακροδεξιός ε, σκότωσε δύο ανθρώπους, ε, δύο τραυματίες επέζησαν. Συνέβη το αδιανόητο. Κάποιος σκοτώνει ε, λόγω μίσους. Ε, επειδή μισεί τους Εβραίους, τους μετανάστες στο κέντρο της Ευρώπης. Πρέπει να το πούμε με το όνομά του. Η επίθεση αυτή ήταν ρατσιστική. Κατευθυνόταν κατά της ανοιχτής κοινωνίας και των ευρωπαϊκών αξιών. Και προφανές ε, είναι ότι δεν είναι μόνος του αυτός ο άνθρωπος. Ε, έχουμε τα όσα συμβαίνουν στο Κέμνιτς που μιλάνε για αντικατάσταση πληθυσμών. Η Λεπέν που μιλάει κατά της ε, μετανάστευσης. Κόσμος που τρώει ξύλο επειδή φοράει μία κυπά. Όλα αυτά πάνε μαζί. Εδώ και χρόνια λοιπόν είναι ενωμένοι όλοι αυτοί. Και εδώ στο κοινοβούλιο αυτό προσπαθούν ε, να δημιουργήσουν ε, κλίμα κατά των μειονοτήτων. Και εδώ πέρα λοιπόν, στο κοινοβούλιο οι δεξιοί ε, ρίχνουν ε, λάδι στη φωτιά. Είναι η πολιτική πτέρυγα του, της ε, τρομοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε αποφασιστικά κατά οποιασδήποτε μορφής ρατσισμού και αντισημιτισμού. Και με ποινική δίωξη. Και ευτυχώς εδώ πέρα η Κομισιόν λέει ότι θα δώσει περισσότερο βάρος στο θέμα αυτό. Αυτό το οποίο συνέβη στο Χάλε. Είναι μια ε, ένδειξη του ότι οι δεξιοί δικτυώνονται πανευρωπαϊκά. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και οι μυστικέ υπηρεσίε και η αστυνομία αλλά και στην πολιτική. Θα πρέπει να δούμε ότι η δεξιά τρομοκρατία είναι δικτυωμένη παγκοσμίω και θα πρέπει όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις να ενισχυθούν κατά της δεξιάς ρητορική ε, στην ταβέρνα, στο δρόμο και στο κοινοβούλιο. Και θα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που κάθε μέρα υπερασπίζουν την ανοιχτή κοινωνία και τις ευρωπαϊκές αξίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόιτεν ε, έχει 100 λόγο. Σας ευχαριστώ. Η επίθεση του Χάλε είναι ένα φρικτό έγκλημα ενός αειδιαστικού ψυχοπαθέους. Βεβαίω είναι λυπηρή η απώλεια της ανθρώπινης ζωής, η οποία θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν κατάφερνε να μπει στην συναγωγή. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τυφλωμένος από αντισημητικό μίσος δεν, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση πως ο δεξιός εξτρεμισμός είναι επικίνδυνος και πρέπει να καταπολεμηθεί με όλα τα μέσα του κράτους, παντού και πάντα. Αλλά εμείς λέμε ότι το κράτος δεν θα πρέπει να ανέχεται κανέναν εξτρεμισμό. Ούτε δεξιό, ούτε αριστερό, ούτε ισλαμιστικό. Κανέναν εξτρεμισμό. Εδώ πέρα λοιπόν τα κράτη μας αποτυχάνουν. Δεν αρκούν οι εμπειρίες. Το γερμανικό κράτος θα έπρεπε να έχει οπλισμένους φρουρούς έξω από όλες τις συναγωγές τη μέρα του Γιώμ Κιπούρ. Το είχαν ζητήσει οι εβραϊκές κοινότητες, μάταια. Πρόκειται για αποτυχία του γερμανικού κράτους. Ευτυχώ ήταν γερή η πόρτα και εμποδίστηκε μια σφαγή, όπως το Christchurch. Δεν έκαναν τίποτα οι υπουργοί. Λοιπόν, αν τώρα εσείς οι οποίοι αποτύχατε κατηγορείτε το κόμμα μου, πρόκειται πραγματικά για κάτι το οποίο είναι σχρό και προσπαθείτε να αποσύσετε τις ευθύνες από πάνω σας. Και κάτι ακόμα. Ο αντισημιτισμός κατά των Εβραίων και του Ισραήλ σήμερα έρχεται κατά κύριο λόγο από τα αριστερά. Είναι στο DNA της αριστεράς. Εσείς, οι πράσινοι και οι αριστεροί, είστε αυτοί οι οποίοι πάντα ενοχλείστε και προσπαθήστε να εμποδίσετε την φιλοϊσραηλινή τάξη. Ε, στάση της ε, Γερμανίας. Και ε, συνεχώς επιμένετε να δίνονται λεφτά στην Χαμάς και έχετε επαφές με τη Χεσμολάχ. Και μας μιλάτε εμάς για αντισημιτισμό. να σας πω κάτι. Αν κυβερνήσουμε εμείς ποτέ, οι Εβραίοι συμπολίτες μας θα προστατεύονται. Προστασία την οποία εσείς δεν δώσατε. Παρόλα τα ψέματα, εμείς είμαστε φίλοι του Ισραήλ, είμαστε φίλοι των Εβραίων αντιληφθείτε το και σταματήστε να μας απευθύνετε τέτοιες κατηγορίες. Είναι κάτι το φρικτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη για τον πρώτο γύρο παρεμβάσεων ε, από τις πολιτικές ομάδες. Δεν μπορούμε να έχουμε μπλε κάρτες, ε, μόνο στη συνέχεια. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπουσάδε Βιλάλβα από το ECR. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, η αντιπροσωπεία τη ομάδα στην οποία ανήκω ανέκαθεν ήταν από τι πρώτε που καταδίκαζαν τον αντισημιτισμό. Σε αντίθεση όμω με άλλε ομάδε εδώ στο Κοινοβούλιο, εμεί είμαστε κατά οποιασδήποτε μορφή παραβίαση ε, και διάκριση ε, ε, για εθνοτικού, φιλετικού ή θρησκευτικού λόγου. Ακόμα και αυτού οι οποίοι οδηγούν σε αρνητική στάση εναντίον ανθρώπων που είναι υπήκοοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί πιστεύουμε στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και όχι στι συλλογικέ μάχε τι οποίε με τόσο μεγάλη χαρά δίνουν οι σοσιαλιστέ δημοκράτες. Όπως ε, γίνεται συνήθως, η αριστερά προσπαθεί να αλλάξει τη συζήτηση για ένα τραγικό γεγονός σε μια συναγωγή στη Γερμανία σε κάτι άλλο για να μιλήσει για φρονούντες. Εσείς ε, χρησιμοποιείτε μια επίθεση και εμείς απορρίπτουμε και καταδικάζουμε την κατάσταση γιατί προσπαθείτε να χειραγωγήσετε την κοινή γνώμη και να προσπαθήσετε να απονομιμοποιήσετε τις πολιτικές ε, επιλογέ που έχουμε. Γι' αυτό και ο τίτλο τη σημερινή συζήτηση είναι κίνδυνο τη βία τη ακροδεξιά και όχι ε, «Κίνδυνος της βίας ή του εξτρεμισμού» τελεία και παύλα. Γιατί εσεί δεν προσπαθείτε να ε, ε, γλιτώσετε από τον ε, εξτρεμισμό. Εάν πραγματικά θέλετε να καταπολεμήσετε τη βία και τον εξτρεμισμό θα πρέπει να πάτε σε μια περιοχή όπου κυριαρχεί ο Ισλαμικό νόμο και όπου οι γυναίκες δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι του ήσυχε. Ε, αν θέλετε λοιπόν να καταλαβαίνετε τη βία και τον εκτρομισμό, θα πρέπει ε, να καταδικάσετε αυτά τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης μου, της Βαρκελόνης, η οποία έχει μετατραπεί σε ναρκοπαίδιο λόγω της ε, ε, αποσχιστικής τάσης που υπάρχει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε Μίχελς ε, για την ΚΟΕ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο πρόβλημα στην ε, Γερμανία είναι πως ε, το Auschwitz έγινε το μέτρο του μίσους ε, κατά των Εβραίων. Οπότε οτιδήποτε ήταν λιγότερο από το Auschwitz επί δεκαετίες δεν είχε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, το, αυτό το ποτέ ξανά έχει γίνει πλέον μια κούφια φράση. Αυτά γράφτηκαν πρόσφατα στην εφημερίδα Die Μετά από το έγκλημα του Χάλε, ακούσαν πάλι την θεωρία του μεμονωμένου τρελού και πάλι το ECR μας μίλησε για ένα τραγικό περιστατικό. Ερωτώ, πώς μπορούμε μετά τις επιθέσεις στο Πρέβετ, τις επιθέσεις σε Παρίσι και Βρυξέλλες μετά τις σχετικές δίκες στην Γερμανία να μιλάτε για μεμονωμένους δράστες. Σήμερα πάλι υπήρξε μια εμπριστική επίθεση σε τζαμί στο Ντόρτμουντ. Όταν οι πολιτικοί ε, μιλάνε για ξαφνικό καμπανάκι, προφανώς κοιμόντουσαν επί δεκαετίες. Ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός ε, δυστυχώς ε, ποτέ δεν έφυγαν από την κοινωνία μας. Στην πραγματικότητα έχουμε μία αποτυχία της πολιτικής επί δεκαετίες και εδώ πέρα υβρίζονται και οι αντιφασίστες. Ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είχαμε σήμερα. Από την εκπαίδευση μέχρι την πολιτική ε, βλέπουμε πως ε, επικρατεί μία τύφλωση. Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός και ο αντισημιτισμός έχει πολλές ε, αιτίες. Το βλέπουμε και από την έλλειψη σεβασμού και τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Και εδώ μέσα, εδώ και χρόνια. Η βίαιη γλώσσα οδηγεί σε βία στους δρόμους. Το, μίος, το μίσος διαλύει την δημοκρατία μας. Πρέπει λοιπόν να τα αντιμετωπίσουμε αυτά συνολικά και διαρκώς και αγαπητοί κομισιόν όχι μόνο στο διαδίκτυο. Δεν βοηθάνε με μονομένα μέτρα. Μόνο περισσότερα λεφτά στην εκπαίδευση, στη δημοκρατία, την ένταξη και ε, έργα απένταξης από την τρομοκρατία. Αυτό λοιπόν χρωστάμε στα θύματα του Χάλε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λαγός έχει τον λόγο. Please use your mic. The translator cannot hear you. Thank you. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω λέγοντα αρχικά ότι φυσικά είναι καταδικαστέο το ότι συνέβη πριν από λίγε μέρε. Όμω, και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, δεν είναι δυνατόν να ξεχάσουμε ότι αν υπάρχει μια θρησκευτική ομάδα που αυτά τα χρόνια βρίσκεται υπό διωγμό, είναι ο χριστιανισμό και είναι και οι χριστιανοί. Και μάλιστα μου κάνει τρομερή εντύπωση πώ στο Κοινοβούλιο συζητάμε αυτή τη στιγμή και λέμε αυτά τα πράγματα, όταν πριν από λίγη ώρα μόνο έγινε μια συζήτηση για να υπάρχει μια συζήτησε και ένα ψήφισμα για τις διώξεις που υφίστανται οι χριστιανοί στη μέση ανατολή και στη συρία και η πλειοψηφία των βουλευτών αρνήθηκε να το συζητήσει. δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε la κάρτε ευαίσθητοι σε θρησκευτικά ζητήματα γιατί σύμφωνα με έρευνες που υπάρχουν και από το fox news οι χριστιανοί είναι η πλέον διωκόμενη ομάδα την τελευταία διετία τουλάχιστον. επίσης αν δούμε από διάφορα site και, ε, και διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβητήσεις στην πατρίδα μου τουλάχιστον στην ελλάδα το 2018 υπήρξαν 574 επιθέσεις σε χριστιανικούς ναούς για τους οποίους δεν ακούστηκε τίποτα επίσης υπήρχαν επιθέσεις σε πάρα πολλούς ναούς χίλιους εξήντα αν δεν κάνω λάθος σε χριστιανικούς ναούς στη γαλλία όπως και σε 450 περίπου στη γερμανία. Γι' αυτά πραγματικά δεν έχει ακουστεί τίποτα. πώς λοιπόν υπάρχει ο όρος και συζητάμε όλοι και λέμε για αντισημιτισμό αλλά δεν συζητάμε για αντιχριστιανισμό σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν. γιατί εσείς οι δημοκράτες και όπως τα συζητάμε θα έπρεπε λοιπόν να τα βάζουμε αυτά και να βλέπουμε τι γίνεται. ισχύουν από τη μία πλευρά καταδικαστέα σίγουρα αλλά αν ισχύουν στο πολλαπλάσιο από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να σιωπούμε. και όσο έχει να κάνει και επιτρέψτε μου δέκα δεύτερα ακόμα όσο έχει να κάνει με την ακροδεξιά βία τουλάχιστον στην πατρίδα μου σύμφωνα με έκθεση της europol στις 23 του 2018 η ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της ακροαριστερή βία με τρομοκράτε που είναι πάνοπλοι με βαρύ οπλισμό. μην διηλύσουμε λοιπόν τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλο. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Από το ΕΛΚΕ κυρία Νίμπλερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή για τον εξτρεμισμό και τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη. Πριν από 15 μέρες είχαμε αυτήν την φρικτή ένοπλη επίθεση σε μια συναγωγή στο Χάλε, στην οποία όπως γνωρίζετε δολοφονήθηκαν δύο άνθρωποι. Η φρικτή αυτή επίθεση μας δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε την εβραϊκή ζωή στη Γερμανία. όχι μόνο στην Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο αντισημιτισμός ε, ξαναεμφανίζεται σε πολλές ε, χώρες. Ε, βλέπουμε εβραϊκούς τάφους να βεβηλώνονται με αγγελωτούς σταυρούς νεοναζί, ε, κάνουν πορείες ε, και χαιρετούν ε, ναζιστικά. Αυτά ζούμε κάθε μέρα. Αρχές του έτους είχαμε εδώ την Σαλότ Κνόμπλαουχ επευκαιρία της Διεθνούς ημέρας για το ολοκαύτωμα και μας είπε ότι ο αντισημιτισμός αυξάνεται και όχι μόνο στη Γερμανία αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι Εβραίοι συμπολίτε μας σκέφτονται πλέον να φύγουν από την Ήπειρό μας. Βεβαίω, ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε να γίνει κάτι τέτοιο κανονικότητα. Αν δεν αισθάνονται ασφαλείς οι Εβραίοι συμπολίτε μας έχουμε αποτύχει. Θα πρέπει, θεωρώ, να υπάρξει μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία κατά του αντισημιτισμού και του δεξιού εξτρεμισμού. Βεβαίω, πρώτα απ' όλα το διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι τελείως ανεξέλεγκτο. Δεύτερον, θα πρέπει να διευθύνουμε τους νέους και τρίτον, ε, και το τονίζω αυτό, θα πρέπει να ονομάσουμε τα κόμματα εκείνα τα οποία διασπείρουν μίσος και προετοιμάζουν το έδαφος για τον αντισημιτισμό. Ο κύριος Μόιτερ έφυγε. Έχει δίκιο, πράγματι. Εξτρεμισμός πρέπει να καταπολεμηθεί και από δεξιά και από αριστερά. Αλλά όταν οι εκπρόσωποι του κόμματός του λένε ότι το μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο ε, ως μνημείο ντροπή, ε, τότε όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ Ιντσίρ. Κυρία Πρόεδρε, κάτι σάπιο υπάρχει στην Ευρώπη. Ο αντισημιτισμός ε, προχωράει σε πολλές χώρες στην Ευρώπη και βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο βία και τρομοκρατία από λευκούς εξτρεμιστές. Και αυτό φυσικά γίνεται γιατί έχει θεωρηθεί κανονικό και ο δεξιός εξτρεμισμός. Ακόμα και εδώ στην Ολομέλεια έχουμε ανθρώπους που έχουν τέτοιες απόψεις. Όπως είπατε, η λεκτική βία μετατρέπεται πολύ εύκολα σε σωματική βία. Η επίθεση στο Χάλε ήταν επίθεση κατά της δημοκρατίας συνολικά. Η βία και η τρομοκρατία από το δεξιό εξτρεμισμό δεν είναι κάτι καινοφανές ε, στην Ευρώπη. Το είδαμε και στη δεκαετία του 80 στην Βαρκελόνη και στη Νέα Ζηλανδία το 2019 και είδαμε και την Ευρώπη ε, να γίνεται ρήπια λόγω των ε, ακροδεξιών δυνάμεων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές θεωρούνται από την αστυνομία ως την απειλή που μεγαλώνει πιο γρήγορα. Ακόμα και η Ευρωπόλ στην έκθεσή της λέει ότι ο αριθμός των συλλήψεων από την βία ε, του δεξιού εξτρεμισμού αυξάνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Όλοι λοιπόν ουσιαστικά βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο με διαφορετικές εκφάνσεις. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιτίθεται στον οποιονδήποτε έχει διαφορετική πολιτική άποψη, γυναίκες, ε, Εβραίους, μετανάστες η Ευρώπη πρέπει να υψώσει το ανάστημό τη ενάντια σε όλα αυτά τα πράγματα. Ε, φυσικά εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο στα κράτη-μέλη και αυτό δημιουργεί τεράστιο χάσμα μεταξύ των αδικημάτων και των εγκλημάτων τα οποία καταγγέλλονται. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τους παρόχους ε, υπηρεσιών στο διαδίκτυο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις επιθέσεις μίσους ε, στο διαδίκτυο. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος και να χτίσουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Κέρνερ από το Ρινιού. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εδώ και χρόνια δολοφονούνται άνθρωποι από ρατσιστές και ακροδεξιούς. Και η απάντηση είναι ίδια. Το Τσέσου θέλει να απαγορεύσει τα παιχνίδια των υπολογιστών, άλλοι θέλουν να κλείσουν τα σύνορα και άλλοι να περιορίσουν τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτά δεν θα εμπόδιζαν το έγκλημα όμως το χάλε. Αυτό το οποίο θα το εμπόδιζε ήταν η παρουσία της αστυνομία. Αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν επιτέλους το προσωπικό και τους ε, πόρους ε, και την αστυνομική συνεργασία. Αλλά κάθε αντισημιτική επίθεση στην Ευρώπη είναι αποτυχία του κράτους και ντρέπομαι ιδιαίτερος ως Γερμανός ε, για το ότι οι Εβραίοι αισθάνονται πάλι ανασφαλείς στην Ευρώπη. Βεβαίως, η αύξηση του αντισημιτισμού οφείλεται, λέει, στην αύξηση της μετανάστευσης. Αυτό είναι λάθος τα στοιχεία της κρατικής ασφάλειας στη Γερμανία δείχνουν κάτι άλλο. Συνολικά τα αντισημιτικά εγκλήματα ναι αυξήθηκαν. Ναι και από άλλο αλλοδαπούς, αλλά ακόμη περισσότερο αυξήθηκαν αυτά από ακροδεξιούς. 2018, 1600 τέτοια εγκλήματα από ακροδεξιούς, ε, σαφώς λιγότερα από μετανάστες. Όποιος λοιπόν δεν λέει ξεκάθαρα ότι ο αντισημιτισμός είναι κύριος δεξιός, είναι λάθος και πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κούνκε από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το μίσος ε, κατά των Εβραίων είναι κάτι που το συναντάμε παντού, ακόμη και εδώ. Ακόμη και αν η λύκη είναι ντυμένη πρόβατα. Η επίθεση στο Χάλε αποτελεί έκφραση αντισημιτισμού και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να ντρεπόμαστε σε σχέση με το προς τα που θέλουμε να οδεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, πολλοί από εμά δεν εκπλαγήκαμε ετοιμότητα να προστατεύσει κανείς ανθρώπους που έχουν δικαίωμα να πιστεύουν ότι επιθυμούν και να ζουν ελεύθερα. Δεν ε, έτυχε διασφάλιση η ελευθερία αυτή και αυτό συνέβη στο Χάλε. Θα πρέπει να σταματήσουμε τους ακροδεξιούς εκτρεμιστές. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε προληπτικά μέτρα τα οποία θα τεθούν σε ισχύ θα έπρεπε μάλλον να ισχύουν ε, πριν να υλοποιηθούν οι επιθέσεις. Έτσι λοιπόν, εμείς οι πράσινοι καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απευθύνεται στα κράτη-μέλη για να λάβουν ε, κάποια προληπτικά μέτρα. Σε ευχαριστώ. Χάκαρα είναι από το ID. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλες ε, ε, αυτές οι βίες δράσεις ε, αποτελούν απειλή κατά της ασφάλειας. Αλλά εδώ καταδικάζουμε μόνο τις ακροδεξίες πράξεις. Γιατί συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι ε, και οι Ισλαμιστές αλλά και η ακροαριστερή βία είναι η κύρια απειλή κατά της Ευρώπης. Και πάλι οι Εβραίοι εδώ παρουσιάζονται ως ε, θύματα και μάλιστα έχουν διωχθεί και από κάποιες ε, χώρες. Όμως ε, οι βίοι Ισλαμιστές είναι η μεγαλύτερη απειλή και αυτό λόγω της ανεξέλεκτης μετανάστευσης. Ο εβραϊκός λαός πρέπει να χαίρει της υποστήριξής μας. Γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια θέματα στην ε, Ολομέλεια. Ακολουθούμε μια επικίνδυνη οδό. Αν αφιερώνουμε το χρόνο μας στο να καταδικάζουμε μόνο ένα μέρος του εξτρομισμού. Ε. Σας ευχαριστώ, από το Ευχαριστώ πολύ. Τα γεγονότα στο χαλέ μας δείχνουν ε, το μέγεθος αυτής ε, της ε, αντισημιστικής ντροπιαστικής πράξης που βλέπουμε όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στη Γαλλία, ούτε στο Βερολίνο ούτε στο Παρίσι. Τολμάει κανεί να πει ότι είναι Εβραίος. Βέβαια, νομίζω ότι οι Γερμανοί συνάδελφοι θα πρέπει να εξετάσουν την κατάσταση στη χώρα τους, αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και τα εγκλήματα που διεπράχθησαν ε, από τους Ναζί. Εδώ βλέπουμε μεγάλη ριζοσπαστικοποίηση και στα δεξιά και στα αριστερά. Στη Γερμανία η ακαδημαϊκή ελευθερία έκφρασης παρεμποδίζεται. Και φυσικά αυτό έπληξε και τον συνάδελφο Μπέρντ Λούκ, του βουλευτή. Στην ε, Γαλλία έχουμε κατάχρηση εξουσίας ε, απέναντι στα κίτρινα γυλαίκα ε, ε, και σε διάφορες πόλεις βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους ε, να διαδηλώσουν και υπήρξε ή καταστολή. Και μπορούμε όμως στη συνέχεια να ασχοληθούμε με τα θέματα της Πολωνίας με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ ο κύριος Σουρμπαν Κρέσπο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η άνοδο τη ακροδεξιάς ε, μας παραπέμπει στα χειρότερα φαντάσματα της Ευρώπης. Όμως υπάρχει επίσης κάτι επικίνδυνο εξίσου το πώς ε, ε, αγοράζουν τις προτάσεις της ακροδεξιάς. Αυτό το κάνουν τα μεγάλα νεοφιλελεύθερα κόμματα στην Καταλωνία, στη Γαλλία ή στη Μεσόγειο. Ε, από ό,τι φαίνεται η έκτακτη ανάγκη αιτιολογεί περικοπές δικαιωμάτων και ελευθεριών και τελικά κανονικοποιεί την ακροδεξιά. Η ευρωπαϊκή πολιτική ζει σήμερα μια λεπενοποίηση σε επιτάχυνση που θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία στην Ήπειρο αυτή η δημοκρατία την ε, κατακτήσει οι αντιφασίστες, να το θυμόμαστε. Και επίση ε, δεν φτάνει ε, σήμερα να φύγει το, το με του Φράνκο από την κοιλάδα, αλλά αυτό που επήγει είναι να καταπολεμήσουμε τις πολιτικές της άκρας δεξιάς και να μην υιοθετούμε τα ε, αρχικά κάτω από τα οποία κρύβονται. Και γι' αυτό πρέπει πάλι να φωνάξουμε ενώ πασαράν. Ακολουθεί η κυρία Φόξ για ένα λεπτό. Η επίθεση στο Χάλε ήταν ε, φρικτή. Είναι τόσο σοκαριστικό το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι που γιόρταζαν το Γιάμ Κιπούρ, τόσα εβραϊκά κέντρα χρειάζονται τώρα υποστήριξη. Αλλά έχω να πω κάποια πράγματα για αυτό που κάνουμε ω αντίδραση. Δεν πρέπει να είμαστε πολύ απλοϊκοί. Αυτοί που λένε ότι ο αντισημιτισμό περιορίζεται στην ακροδεξιά, πρέπει να πω ότι κάποιο ε, που βρίσκεται στα αριστερά τη πολιτική, δυστυχώ υπάρχουν και αριστεροί οι οποίοι είναι ε, αντισημίτε. Και δεν το λέω αυτό για να πω ότι α, έχουμε και από εδώ και έχουμε από εκεί, αλλά απλώ να είμαστε ειλικρινεί για το τι συμβαίνει. Και πρέπει να πω ότι είναι μεγάλη πρόκληση όταν βλέπουμε τέτοια βία να ε, ε, κατηγορούμε τους πάντες, αλλά πιστεύω ότι η γερμανή πολιτική ε, και κάθε κράτος μέλος δεν θα πρέπει να ζητά να γίνουν απαγορεύσεις, να γίνεται επίθεση στην ελευθερία του λόγου, διότι ε, μπορεί να επιτιθέμαστε στην ρητορία του Μέσου, αλλά δεν θα πρέπει να στερούμε την ελευθερία στον κόσμο να μιλήσει. Οι κατηγορίες για ρητορία για όποιον διαφωνεί μαζί σας δεν είναι πραγματικότητα, διότι στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι είναι ε, ο θάνατος του εξτρεμισμού. Εμείς είμαστε αυτοί που αγαπάμε την ελευθερία και ε, είμαστε κατά του αντισημιτισμού και της οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων. Ακολουθεί ο κύριος για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για αυτή τη συζήτηση η οποία είναι πολύ επίκαιρη και μας επιτρέπει όχι μόνο να δούμε τους δράστες αυτών των εγκλημάτων αλλά και τα θύματα. Και όταν στοχεύουμε στα θύματα διαπιστώνουμε και πάλι ότι υπάρχει αντισημιτισμός και ευρεοφοβία οι οποίες βρίσκονται στη ρίζα αυτής της ε, ε, εγκληματικής ε, δράσης. Η ακροδεξιά, η αρκαία ακροαριστερά, ο τζιχαντισμός, ο Ισλαμισμός, όλα αυτά ε, κάνουν τον όλοι αυτοί θεωρούν τον αντισημιτισμό ε, τον κοινό εχθρό και οι οπιτιμητικές συζητήσεις και το γεγονός ότι θεωρούμε ότι το λοκα... αυτόμα δεν συνέβησε δίνουν διαφορετικό ε, δυνατότητα και ανοίγουν το δρόμο για τη βία. Η σιωπή ήταν πάντα ο πιο αποτελεσματικό σύμμαχο και ο πιο διαστραμμένο σύμμαχο του αντισημιτισμού. Αυτό το περιβόητο δεν ξέραμε τίποτα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και ξέρουμε και βλέπουμε και ακούμε ότι ο αντισημιτισμός ε, προχωράει και πρέπει να τον καταπολεμήσουμε διότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γνωρίζουμε ότι όταν ε, ο αντισημιτισμός ε, προελάφνει αντιμετωπίζει την τραγωδία. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μιλάμε για μια σιωπηρή έξοδο των Εβραίων. Επιτρέψτε μου λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι εγώ να τονίσω αυτή τη στιγμή ότι στην Ισπανία χάρη σε μια πρωτοβουλία του ε, Λαϊκού Κόμματος του Παρτίδο Ποπουλάρ τα τελευταία χρόνια πάνω από 31.000 ε, Σεφαρδοί Εβραίοι έλαβαν Ισπανική υπηκότητα, που είναι απόγονοι αυτών οι οποίοι εκδιώχθηκαν το 1492. Σε μια πράξη αναγνώρισης λοιπόν, αναγνωρίζονται ως Ισπανοί και ως Ευρωπαίοι. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Μπιεντρών. Ευχαριστώ πολύ. Κατά τη συζήτηση αυτή ακούσαμε κάποιους σημαντικούς όρους στη χώρα μου λειτουργούσαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ακούσαμε και το Auschwitz. Όμως ε, δεν ε, βασιζόταν ε, στην ιδεολογία του κρεματόριου. Αυτή η ιδεολογία είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Εμείς όταν ε, ε, και με μια συναγωγή ή ένα τζαμί ή όταν ε, καταφερόμαστε κατά των ενυπεράσπιστων μεταναστών ή όταν μπαίνει φωτιά σε ένα χώρο υποδοχής μεταναστών, τότε βλέπουμε ότι όλα αυτά παρακινούνται από κάποιους ε, πολιτικούς ηγέτες. Μας λένε ότι οι μετανάστες ε, μολύνουν την κοινωνία μας ε, και εδώ έχουμε εκπροσώπους κομμάτων που ζήτησαν ελεύθερες ζώνες από ΛΟΑΔΜ. Έχουμε και τη χείρα ε, του Παύλα ε, ο οποίος δολοφονήθηκε γιατί κάποιος ήταν κατά των πεπιθήσεών του. Ο κύριος Αντάμοβιτς ε, ζητούσε να σταματήσει ο διωγμός εναντίον των ανθρώπων που βοηθούσαν τους μετανάστες. Η χείρα του έγινε βουλευτής είναι μεταξύ μας. Δεν πρέπει όμως ε, να το ξεχάσουμε. Προέρχομαι από μια χώρα όπου υπάρχει η αλληλεγγύη και απευθύνομαι στους ε, ανθρώπους ε, που είναι αλληλέγγυοι. Το μίσος πρέπει να το αποκαλούμε με το όνομά του. Θα πρέπει τα πράγματα να τα αποκαλούμε όπως έχουν πριν να δημιουργήσουμε ένα νέο Auschwitz. Ευχαριστώ, Φάνεν, για το Ρινιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν δύο εβδομάδε, ε, ένα άνθρωπο άνοιξε πύρε στη Χαλέ μια αντισημιστική επίθεση κατά μια συναγωγή στη μέρα του Γιώμ Κιπούρ. Και αναμετάδωσε για 35 λεπτά τι πράξεις του ζωντανά στο διαδίκτυο. Χιλιάδες άνθρωποι είδαν τι εικόνε ε, αυτές. Ε, και αυτό μα θύμισε τη σφαγή στο Christchurch. Χρειάζεται ε, γρήγορη αντίδραση, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, και να αποσυρθεί το τρομοκρατικό επιγραμμικό περιεχόμενο. Ε, ο κώδικας του 2016 δεν αρκεί ούτε η φυστάμενη νομοθεσία. Θα πρέπει να αποσύρουμε όλο αυτό το περιεχόμενο στις διάφορες πλατφόρμες και στα επιγραμμικά φόρα. Να μην χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για την κανονικοποίηση του εξτρομισμού. Επίσης, θα πρέπει να διαπιστώσουμε την άγνοια τη ιστορία Με Ένα ε, νέο στου 10 δεν γνωρίζει το ολοκαύτωμα. Έτσι λοιπόν να καταπολεμήσουμε το κακό στη ρίζα, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Έτσι λοιπόν θα καταστήσουμε πιο ελεύθερου και πιο υπεύθυνου του χρήστε του ίντερνετ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Λαγκοντίνσκι για του πράσινου. Εδώ και μέρες μιλάμε για το περιστατικό του Χάλε ε, εναντίον ο ένας του άλλου, χωρίς να ακούν ο ένας τον άλλον. Οι δεξιοί παριστάνουν ε, ότι δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα, σαν ε, να μην έχουν πει το ολοκαύτωμα ατύχημα της ιστορίας, σαν να μην ζητούν να αλλάξει η πολιτική μνήμης της Γερμανίας. Εγώ ο ίδιος μέλος της ε, εβραϊκής ε, κοινότητας, Γερμανός, Ευρωπαίος, ντρέπομαι για όλα αυτά. Παρόλα αυτά ε, επιμένω ότι προέκυψε αυτό το περιστατικό από την δεξιά. Αλλά και αριστερά του κέντρου πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Και εμείς πάρα πολύ απλά κοιτάμε μόνο τους δεξιούς. Πάρα πολλές από αυτές τις συζητήσεις είναι κυκλικές. Ε, συζητάμε αν ήταν ε, μεμονωμένος ή όχι, αν θα απαγορέσουμε το FDA ή όχι. Όλα αυτά είναι μάταια αν δεν βρούμε τους πραγματικούς υπεύθυνου. Υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όχι όλοι ένοχοι, αλλά υπεύθυνοι. Ακολουθούμε συνεχώς ε, τα, τις ίδιες διαδικασίες αντί να πούμε την αλήθεια. Και ναι, μπορούμε να κάνουμε κάποια απλά πράγματα. Μπορούμε να διασφαλίσουμε τις ε, ΜΚΟ που μάχονται κατά του δεξιού και αριστερού αντισημιτισμού. Να δημιουργήσουμε τις ελάχιστες συνθήκες ασφαλείας για τις εβραϊκές εγκαταστάσεις. Να δούμε το ψήφισμα για τον ρατσισμό και επιτέλους να τιμωρηθεί το μίσος ποινικά σε όλες τις χώρες. Και ακριβώς η νέα πρόεδρος της ε, Κομισιόν μπορεί να κάνει κάτι το απλό, να στείλει ένα μήνυμα ότι η καταπολέμηση του αντισημιτισμού είναι κάτι το βασικό. Μπορεί να φέρει την Καταρίνα Φωνσνό Βάλεν εδώ πέρα, να την πάρει στο επιτελείο της. Αυτό θα είναι νομίζω μια πολύ καλή αρχή για την νέα Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κυρία Ριβιέ, ο κύριος Ριβιέρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η επίθεση που έγινε στη συναγωγή του Χάλε ε, μας δείχνει ότι επιστρέφει ο αντισημιτισμός στην Ήπειρά μας, κάτι το οποίο βλέπουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Ε, το Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι τα αίτια του αντισημιτισμού, τα οποία θα πρέπει να βρούμε και να ε, εκριζώσουμε. Ένας ε, νεοναζί διέπραξε υποτίθεται αυτή την τρομοκρατική πράξη. Εδώ και 30 χρόνια, με κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις, αυτές οι επιθέσεις είναι ε, ε επιθέσεις ε, Αράβων ή Μουσουλμάνων τρομοκρατών, όπως αποδείχθηκε από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στη Γαλλία, τα ονόματα Ανιλή, Λόλ, και άνθρωποι οι οποίοι είναι βίαιοι και ε, ριζοσπαστικοποιημένη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται σε αυτές τις ε, μουσουλμανικές χώρες και να ε, σταματήσουμε να μην ξεχνάμε ότι η ακροαριστερά στην Ευρώπη είναι ο προθάλαμος του αντισημιτισμού. Θα πρέπει λοιπόν κατεπηγόντως να κλείσουμε όλα τα τζαμιά στην Ευρώπη των σαλαφιστών και να υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις και να καταδικάσουμε ε, το Ισραήλ για την ε, ε, ολοένα και πιο βία η δράση της ακροδεξι... ακροαριστεράς. Ράισον για το ECR. Κύρια Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο από αυτή την επίθεση, ότι ο αντισημιτισμός εν 2019 εξακολουθεί να είναι ζωντανός οι αριθμοί ε, ζωγραφίζουν μια τρομακτική εικόνα. Ο αντισημιτισμός είναι ένα τέρας με πολλά κεφάλια και πρόσωπα, αριστερά, δεξιά και ισλαμιστικά. Λοιπόν, απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει την καταπολέμησή του κορυφαία προτεραιότητα με επαρκείς δυνάμεις για να υπάρξει επιτέλους ο απαραίτητος συντονισμός με τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπιστεί πολύ σκληρότερα το θέμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, δεν επιτρέπεται πλέον να αποστρέφουμε το βλέμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί η κυρία Ρέγκο για την ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ τα υπάρχει μεγάλο κατάλογο θυμάτων. Ο Παύλο Φίσας, νομίζω ο κύριο Λαγός τον γνωρίζει, Τζο Κόξ, Κάρλο Παλωμίνο, ε, η σφαγή της Νοτόγιας συνεχείς επιθέσει στους δρόμους. Ε, πριν τέσσερι μέρε, μια ομάδα νεοναζί ξυλοκόπησε ένα νέο στη Βαρκελόνη. Η βία της ακροδεξιάς δεν είναι αποτέλεσμα ε, μιας στιγμής που λένε κάποιοι. Αποτελεί προϊόν μια αλυσίδα ευθυνών που ξεκινά από κάποιου, που καθόνται στο απέναντι έδρανα, στα απέναντι έδρανα ή ε, από κάποιου που τους ψηφίζουν ε, υπάρχει μία σειρά ε, λόγων που αιτιολογεί τις επιθέσεις κατά των γυναικών και υπάρχουν και δεσμοφυλάκες που ασκούν αυτή τη βία. Ε, και πέρα από το να προβληματιστούμε σοβαρά βλέπουμε το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανεύθυνο τρόπο να υιοθετεί τις ιδέες των φασιστών και των λόγων τους. Και γι' αυτό ε, έχουμε και τον δυστυχή τίτλο «Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής» ε, του χαρτοφυλακίου αυτού, όπως είδαμε. Ας ακούσουμε τι έλεγε ένας ε, παλιός Ισπανός αντιφασίστας. Δεν συζητάμε για τον φασισμό, αλλά τον καταπολεμούμε. Κυρία συνάδελφε, η παρέμβασή σας ε, προκάλεσε μια μπλε κάρτα. Την δέχεστε από τον συνάδελφο. Μπλε κάρτα. Την μπλε κάρτα πατήσατε. Αν δεν είναι μπλε κάρτα, συνεχίζουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, δίνω τον λόγο στον κύριο Φόρμαν για ένα λεπτό. Με ναι, μπλε κάρτα είναι. Where? You, you put a blue card? Α, μπλε κάρτα ήταν. Εντάξει. She accepted already, so... Δέχτηκε ήδη. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούω τέτοιε δηλώσεις όπως η δική σας. Δηλαδή ένας ε, γκέι ε, ε, μαύρος το χάρη ε, θα θεωρήσει ότι κάποιος που κάθεται από την άλλη πλευρά είναι ρατσιστής, ξενόφοβος. Εσείς ε, λέτε ότι έτσι την Ευρώπη. Όμως ε, εδώ μιλάμε για ρατσισμό, μιλάμε για τη δημιουργία μίσος. Ε, έτσι λοιπόν θα πρότεινα να δείτε τον εαυτό σας και στον καθρέφτη και να σκέφτεστε τι λέτε πριν να χρησιμοποιείτε τις διατυπώσεις. Γιατί η διατύπωση που χρησιμοποιείτε χρησιμοποιείτε όταν θα έρθουν οι πραγματικοί ναζί και ρατσιστές δεν θα μπορούσατε να τους εντοπίσετε και να τους ταυτοποιήσετε. You have, you have 30 seconds for the answer, please. 30 δευτερόλεπτα να απαντήσετε. Αυτό δεν έχει να κάνει με τομικά ζητήματα, αλλά με πολιτικές θέσεις και αυτό που ε, προτείνουν ε, πολλοί συνάδελφοι και ομάδες τους σχετίζονται με τη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και στρέφονται κατά πολλών ανθρώπων. Δεν πρόκειται λοιπόν για προσωπικό ζήτημα, πρόκειται για πολιτικές γραμμές και συγκεκριμένες ιδέες που διαχέουν δικές σας πολιτικές ομάδες. Εδώ δεν μιλάμε για άτομα σίγουρα και ε, θα είχα διαφορετικές ε, θέσεις εγώ σαν άτομα, αλλά εδώ υπερασπίζω μία πολιτική θέση. Αυτό που κάνει η δική σας οργάνωση είναι συνεχώς να ε, θέτει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να εξηγήσω κάτι. 30 δευτερόλεπτα είναι οι ερωτήσεις και 30 δευτερόλεπτα οι απαντήσεις. Το λέω έτσι γιατί είναι και ο χρόνος μας περιορισμένος. Περνάμε τώρα στην δική σας παρέμβαση. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι, από ό,τι κατάλαβα, εάν ε, μεταφράστηκε σωστά, ε, μας είπαν εδώ πέρα ότι εμείς δίνουμε το χέρι μας στην ε, δεξιά τρομοκρατία. Πρόκειται για προσβολή και αναμένω να τους ανακαλέσετε στην τάξη, κυρία Πρόεδρε. με συγχωρείτε, συνάδελφε, εγώ δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο. αφήστε με να τελειώσω. Θα το δούμε στα πρακτικά και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Συνεχίζουμε για την ώρα. Περνάμε τώρα στον κύριο Φαντάλεν. 1,5 λεπτό. Α, συγγνώμη, δικό μου λάθος. Είχα διαγράψει τον κύριο Φόρμαν. Με συγχωρείτε, δεν ήθελα. Λοιπόν, ο κύριος Φόρμαν έχει τον λόγο για τους ε, μη εγγεγραμμένους. Για ένα λεπτό. Την ίδια στιγμή που ένας δολοφόνος χτυπούσε στις πόρτες της συναγωγής ε, στη Χάλε, το Γιόμ Κιπόρ, την πιο ε, σημαντική μέρα της δικής μου της ημέρας, εγώ στεκόμουν έξω από τη συναγωγή στο Λονδίνο, φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ε, παρακολουθώντας την, τον εορτασμό στη δική μου την κοινότητα. Δυστυχώ, οι Εβραίοι ανά τον κόσμο προστατευόμαστε ε, δύο γενιέ ήδη μετά από το ολοκαύτωμα ε, και ο πατέρας μου είναι ε, επιβιώσας του ολοκαυτώματος. Ο αντισημιτισμός λοιπόν παραμένει στην κοινωνία μου και αποστελεί και προειδοποιητικό μήνυμα. Τι συμβαίνει τώρα με αυτή την ε, αναταραχή. Ο εξτρεμισμός ε, και τα ακραία φαινόμενα αυξάνονται όταν υπάρχουν προβλήματα. Εγώ μπήκα στο κόμμα του Brexit όχι λόγω πολιτικής ή γραφειοκρατίας, αλλά γιατί φοβάμαι ότι η Ευρώπη έχει πάρει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο δρόμο. Υπάρχει ένα επιζήμιο ευρωπαϊκό νόμισμα και ε, έχουμε στην πιο ακραία Ευρώπη που είχαμε ακόμα και μετά από δύο παγκοσμίου πολέμους. Μπορεί να είναι και η τελευταία παρέμβασή μου εδώ στην Ολομέλεια αυτό σας προειδοποιώ. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ε, ανανεωθείτε ως ε, μια εταιρική σχέση ανεξάρτητων ανθρώπων και θα πρέπει να βοηθάμε και όχι να παρακολύουμε τα όνειρα των ανθρώπων που εκπροσωπούμε. Λοιπόν, περνάμε τώρα στον κύριο Φαντάλεν ε, για το ΕΛΚ 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, το καλοκαίρι που μας πέρασε η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δημοσίευσε μια έκθεση Εκεί πέρα φαίνεται ότι τα τελευταία πέντε χρόνια ο αντισημιτισμός αυξήθηκε στην Ευρώπη. Ένα μεγάλο ποστό των Ευρωπαίων στην Ευρώπη παρενοχλήθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω της ε, καταγωγής τους και είπαν ότι έχουν αρχίσει να σκέφτονται να φύγουν από την Ευρώπη και η τελευταία επίθεση στο Χάλε οπωσδήποτε το επιβεβαίωσε αυτό οι αριθμοί είναι πολύ ανησυχητικοί και έχουμε ε, βαρεθεί να λέμε συνεχώς για το δημοκρατικό κράτος δικαίου. Θα πρέπει η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τον αντισημιτισμό πρώτη της προτεραιότητα. Με συγκεκριμένα μέτρα, παραδείγματο χάρη να παρακυρίσει τα κράτη-μέλη να εγγυηθούν την ασφάλεια των εβραϊκών εγκαταστάσεων. Να παρακινήσει τα κράτη-μέλη να αναφέρουν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το ολοκαύτωμα, τον αντισημιτισμό και την ιστορία των Εβραίων στην Ευρώπη. Και τέλος, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει κύρια υπόθεσή της την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Και θα πρέπει η συντονίστρια κατά του αντισημιτισμού να είναι υπό την άμεση εποπτεία της ε, Προέδρου της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Ward για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, τα συλληπιτήριά μου σε όλους όσους ε, ε, πλήγησαν από τα γεγονότα στο Χάλα και κυρίως τις οικογένειες των δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Ό,τι και να πούμε εμείς δεν μπορούμε να μετριάσουμε τον πόνο τους, αλλά ξέρω ότι σας υποστηρίζει όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Η πρόσφατη τρομοκρατική ενέργεια στο Χάλε είναι μία ακόμα επωνίδιστη πράξη κατά της εβραϊκή κοινότητας. Ο αντισημιτισμό και η απειλή του δεξιού εξτρεμισμού δυστυχώ αυξάνεται στην Ευρώπη. Ε, φίλοι αναφέρουν, ε, η Γαλλία συγγνώμη, έχει 57% αύξηση και 70% είναι αύξηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που ξεκίνησε η ε, μέτρηση το 1984. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο μας δείχνει ότι έχουμε 36% αύξηση σε ακροδεξιές περιπτώσεις για το 2018. Εγώ εκπροσωπώ πάνω από 500.000 Εβραίου υπηκόου στη Βόρεια Αγγλία και ξέρω ότι δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε εδώ. Ε, ο μόνο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τον αντισημιτισμό είναι ο πολιτιστικό διάλογος, ε, η εκπαίδευση και η μηδενική ανοχή ε, ενάντια σε αντισημιτικέ πράξεις και σε λεκτική βία. Και είμαι φανή για το μουσουλμανοεβρεοϊκό φόρουμ που έχουμε στην περιοχή μου. Έχουμε ε, καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα, πολυφωνία και όλα αυτά θα πρέπει πάντα να διέπουν το όραμά μας για μια κοινή Ευρώπη. Θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από το επονίδι στο παρελθόν, το οποίο οδήγησε στην τυρονία στην Ήπειρό μας και ε, μια Ήπειρος που ξεχνά το παρελθόν της δεν έχει μέλλον σε καμία περίπτωση. Thank Ευχαριστώ. Έχουμε δύο μπλε κάρτες για σας. Α, η μία μόνα. Κύριε Φόρμαν, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Φόρμαν. Όχι, δεν δέχομαι μπλε κάρτες από ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε αυτή την πλατφόρμα ως πλατφόρμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει δικαίωμα η ομιλήτρια να δεχτεί ή να αρνηθεί. Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Λυπάμαι. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτηση. Περνάμε στην κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα για το ρινιό ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Χάνα και ο Κέβιν είναι τα θύματα τη επίθεση στο Χάλε. Μία 40χρονη γυναίκα που τη άρεσε η μουσική pop και αυτό ένα νέο ζωγράφος 20 ετών εξέλιχθηκαν οι ζωέ τους από έναν δολοφόνο γεμάτο μίσο. Αυτός πυροβόλησε, Όμω ε, υπάρχει καλλιέργεια των πράξεων αυτών. Θα πρέπει να καταγγελούμε την αιτία των ακροδεξιών και αντισημιτικό εξτρεμισμό, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε και το πώ το τι είναι ο λόγος των ανεύθυνων ε, που παίρνουν ψήφου, ε, κατασκευάζοντα ε, άλλου μισητούς διαφορετικού. Θα πρέπει να προλάβουμε, να ερευνήσουμε, αλλά θα πρέπει και να επιθυμήσουμε τι μα οδήγησε σε αυτό τον ακροδεξιό εξτρεμισμό. Το πώ είναι τα φερέφωνα αυτοί που μιλούν και ποτέ δεν ακούν μπροστά του, η ειρήνη και ο λόγο, ο διάλογο, ο πλουραλισμό και η συμπάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχουν άλλοι. Συμβιώνουμε άτομα με δικαιώματα, άνθρωποι όπω η Γιάννα, ο ο Μοχάνετ δύο Σαλόμ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Ματζίτ για δύο λεπτά. Friends, Φίλοι, αλάικομ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τα ε, στέλνοντα τα μου συλληπιτήρια και την αιώνια μου μου στην εβραϊκή κοινότητα, ιδίω ε, σε όσου δέχτηκαν ε, επίθεση ε, στην ε, περίπτωση αυτή την, ε, στο Χάλε. Ε, είμαι θυμωμένος, θυμωμένος γιατί είμαστε και πάλι εδώ και πάλι πρέπει να είμαστε θυμωμένοι. Πόσο περισσότερο οι θρησκευτικέ μειονότητε ε, θα πρέπει να ρουλιάζουν απέναντι στο διάφορο πρόσωπο της Ευρώπης, να ρουλιάζουν σταματήστε, σταματήστε ε, να προωθείτε την ακροδεξιά, ε, σταματήστε ε, να ακολουθείτε διάφορα μοντέλα ψηφοφορίας και τις δημοσκοπήσεις. Όταν υποτιμάτε τις θρησκευτικές και για μειονότητες γενετιολογείτε τα ματηρά σύνορα και να αιτιολογείτε τις στρατιωτικές παρεμβάσεις, επελείτε τις ζωές και τους πολίτες τοξικά τμήματα του ευρωπαϊκού τύπου μέχρι τους αδιάφορους πολιτικούς και τους επιγραμμικούς εμπόρους της απανθρωποποίησης. Ε, σε έναν πιο δίκαιο κόσμο θα σας κατηγορούσαν ε, ως συγκατηγορούμενος σε κάθε τέτοιο έγκλημα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει ε, να υπερασπίσουμε όλα τα αδέρφια μας, τους μουσουλμάνους και τους Εβραίους στους δρόμους, είτε είναι σε προσευχή και σε κάθε πόλη και χωριό της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Τσεκάρδη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο δράστης ε, στο Χαλέ ε, ε, πολύ σωστά θεωρήθηκε τρελός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μίσος κατά του κράτους του Ισραήλ γίνεται όλο ένα και πιο ισχυρό. Πριν από κάποιους μήνες εδώ στο Στρασβούργο απογορεύτηκε η είσοδος Ισραηλινών σημεών ε, στο γήπεδο. Στην Ιταλία πολλές φορές ε, η ακροδεξιά δεν επέτρεπε στο εβραϊκό τάγμα να συμμετέχει στους εορτασμούς για την εθνική επέτεδο ε, σε ένδειξη διαμαρτυρίες κατά του Ισραήλ. Υπάρχουν και επιθέσεις ισλαμιστικές στο όνομα του αντισημιτισμού. Και υπάρχουν διαφορετικές εκφάνσεις του ίδιου προβλήματος, αλλά πάντα είναι το ίδιο ε, αποτέλεσμα. Παντού έχουμε διαχωρισμούς και έχουμε κουραστεί. Θα πρέπει ίσως να μάθουμε κάτι από το Ισραήλ. Παρά το γεγονός ότι συμβιώνουν εδώ και χρόνια με την τρομοκρατία, ποτέ δεν είναι... Ε, έσκυψαν το κεφάλι τους, δεν απαρνήθηκαν ποτέ τις ρίζες και τις παραδόσεις τους και το σύστημα των αξιών τους όπως πολύ συχνά κάνει η Ευρώπη. Την τρομοκρατία πρέπει να την παλεύουμε καθημερινά με κάθε μία μέσο όπως μας διδάσκει το Ισραήλ. Ευχαριστώ. Τόμασιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η βία πολιτική ή θρησκευτική φύσεω ε, δεν είναι κάτι καινούριο στην Ευρώπη. Το ε, γεγονό που είναι ανησυχητικό είναι ότι οι στόχοι είναι άνθρωποι με διαφορετικέ πολιτικέ απόψει και ευάλωτε πολιτικέ ομάδε ή άνθρωποι διαφορετική θρησκεία. Φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση σε κάποια στρώματα τη ευρωπαϊκή κοινωνία και αυτό φαίνεται με τον ε, χειρότερο δυνατό τρόπο και θα πρέπει εμεί να το καταγγείλουμε και να το καταδικάσουμε. Η επίθεση στο Χάλε αποτελεί υπενθύμηση του γεγονότο ότι οι βίαιοι άνθρωποι και οι βίαιε ιδέε υπάρχουν σε όλα τα φάσματα του πολιτικού, ε, σε όλε τι ε, πτυχέ του πολιτικού φάσματος και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα καταδικάσουμε. Ε, είναι πάρα πολύ κοινό πλέον το να εισβάλλει κάποιο σε θρησκευτικού χώρους και δεν επιτιθέμαστε μόνο σε μειονότητε. Πολύ συχνά έχουμε και αριστερού εξτρεμισμού που επιτίθεται σε καθολικές ε, εκκλησίες και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά εδώ. Το έγκλημα είναι έγκλημα, ο εγκληματίας είναι εγκληματία ανεξάρτητα του χρώματος τη ε, ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Κιζίλ Γιουρέκη, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώ δεν μπορώ να μιλήσω την μετρική μου γλώσσα, την τουρκική, παρά το ότι είναι επίσημη γλώσσα τη Κύπρου. Οπότε αναγκάζομαι να μιλάω διάφορες άλλες γλώσσες. Λοιπόν, ας είμαστε σαφείς. Δεν υπάρχει δεξιός εξτρεμισμός χωρίς εθνικισμό. Αυτό το ήξεραν πολύ καλά οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ήθελαν να ξεπεράσουν τον εθνικισμό και να δημιουργήσουν μια μεταεθνική ενότητα. Δυστυχώς όμως σήμερα βλέπουμε παντού στην Ευρώπη εθνικιστικές τάσεις. Και εθνικιστικούς εγωισμούς. Ας είμαστε σαφείς. Η ακροδεξιά βία είναι κυρίως αντρική βία που στοχεύει γυναίκες, ομοφιλόφιλους, μουσουλμάνους κτλ. Για να καταπολεμηθεί λοιπόν χρειαζόμαστε ένα νέο ορισμό του εμείς. Εμείς πρέπει να σημαίνει οι πλουραλιστές Ευρωπαίοι κατά των εθνικιστών που προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ομοιογένεια και να παραμερίσουν την ποικιλομορφία. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε συνάδελφε, τελείωσε ο χρόνος σας. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Χρειαζόμαστε πολιτικές που θα προωθήσουν την κοινωνική ένταξη. Ένα λεπτό είναι λίγο, το ξέρω, λέει η πρόεδρος, αλλά έχει τελειώσει εδώ και πολλή ώρα. Ακολουθεί ο κύριος Ραντατσόφσκι για ένα λεπτό. Ο εξτρεμισμός είναι ό,τι χειρότερο έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Θα πρέπει να είμαι αντικειμενικός. Οι δυτικοί μας φίλοι ε, είναι οι ιδρυτές ε, του ακροδεξιού και ακροαριστερού εξτρεμισμού, του φασισμού, του αντισημιτισμού, του ρατσισμού. Είχαμε πυρηνικούς ε, πολέμους, στρατόπεδα συγκέντρωσης, απεικιοκρατία και τα σλαβικά έθνη και οι Σλοβάκοι ποτέ δεν ε, πρόθυσαν τέτοιες ιδεολογίες. Πάντοτε πολεμούσαμε τέτοιες ιδεολογίες. Αν η Ευρώπη δεν δεχτεί, δεν δέχεται ε, να υπάρχουν τα σλαβικά έθνη στο κέντρο της Ευρώπης ε, και δεν είναι ενωμένη η Ευρώπη από το Βλαδιβοστόκ ε, μέχρι την α, δυτική της πλευρά τότε θα οδηγηθούμε σε καταστροφή. Εγώ είμαι περήφανο που είμαι Σλοβάκος. Σα ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Σούλτσα για ένα μισή λεπτό. Κύρια Πρόεδρε, κύριε εκπρόσωπο της Κομισιόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Τότε μιλάμε σήμερα για το Χάλε που βρίσκεται στην Σαξονία, στη δική μου περιφέρεια, με λυπή. Είμαι βουλευτής εδώ πάνω από πέντε χρόνια. Πάντα πάλευα για την πατρίδα μου στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα όμως να μην γίνει αυτή η συζήτηση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι πριν από 15 μέρες συμμετείχαν στην σίγη ενός λεπτού στις Βρυξέλλες, κάτι το οποίο συγκίνησε τους ανθρώπους στην πατρίδα μου. Στη Γερμανία Έχουμε χιλιάδες εξτρεμιστές, δεξιούς αριστερούς. Πολλοί από αυτούς είναι γνωστοί και στις αρχές. Αυτός ο δράστης δεν ήταν. Δεν ήταν γνωστός στις αρχές. Υπάρχει κάτι επίσης στη Γερμανία που πρέπει να το πούμε. Σε πολλά κοινοβούλια, τοπικά και στο εθνικό, ακούμε ρητορική του εθνικοσοσιαλισμού. Οι άνθρωποι αυτοί βεβαίως νομικά δεν υπεύθυνοι, αλλά δημιουργούν το υπέδαφος ε, για τα όσα συνέβησαν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ενωμένοι και δεν θα πρέπει να δίνουμε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Ραφαέλα για ένα λεπτό. Αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πάνω απ' όλα, να έχουμε αυτή τη συζήτηση, θέλω να στρέψω τη σκέψη μου στα θύματα του Χάλε και στους ε, συγγενείς τους. Ε, ο ακροδεξιός εκτρεμισμός ε, απειλεί παγκοσμίω την κοινωνία μας από το Christchurch μέχρι το Χάλε. Βλέπουμε ανθρώπους που πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι λόγω της φυλής τους, του φίλου τους και των πεπιθήσεών τους. Και όλοι γνωρίζουμε που οδηγεί το σκεπτικό αυτό η ακροδεξιά, η πλατφόρμα στο διαδίκτυο καταστούν πιο εύκολο να διαδοθούν αυτές ε, οι ιδέες ε, του μίσους ε, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το όπλο τους για να διαδώσουν τις ιδέες τους. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε τη συνεργασία των πλατφορμών και των εταιριών. Θα πρέπει να μπορούμε να καταλάβουμε πώς διαδίδονται οι πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες προς όφελός τους. Έτσι λοιπόν, καλώ την Κομισιόν ε, να πιέσει τις ε, εταιρείε του διαδικτύου και τις πλατφόρμες να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές και να είναι διαφανείς. Ευχαριστώ Φραντς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αυτή η αντισημιτική επίθεση στο Χάλε είναι απλά το τελευταίο κρούσμα των ρατσιστικών εξελίξεων. Ρωμά καίγονται, δολοφονούνται στην ε, Γερμανία και στην Ιταλία. Όλες οι μειονότητες κινδυνεύουν. Τους έχουμε και εδώ μέσα αυτούς ε, με τα εμπεριστικά τους λόγια με τα λόγια σας και τον χαζό ρατσισμό σας προετοιμάζετε το έδαφος για την πολιτική βία κατά των μειονοτήτων. Οι φαντασίες σας ε, αποτελούν ε, μια οφθαλμαπάτη η οποία αποσπά την προσοχή από τα κοινωνικά προβλήματα για τα οποία δεν έχετε καμία λύση. Μπορείτε μόνο να διχάζετε και να κάνετε προπαγάνδα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο τρόπος με τον οποίο θα προστατεύσουμε την ε, κοινωνία μας είναι μέτρο της κοινωνίας μας. Ο αντισημιτισμός και ο αντιτσιγκανισμός δεν έχουν θέση εδώ μέσα. Ο Κέβιν Ες και η Γιάννα Ελ δεν πρέπει να, να έχουν πεθάνει άδικα. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών στη μάχη της κατά του δεξιού μίσους. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί ο συνάδελφος Φεστ για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ. Η δεξιά τρομοκρατία στη Γερμανία είναι κίνδυνος, δεν ξέρουμε όμως ε, πόσο μεγάλος είναι. Βεβαίως υπάρχει η αρμόδια η υπηρεσία η οποία ε, κατέληξε στους ε, εννέα φόνους του ΕΝΕΣΟΥ. Βεβαίως είχαμε καταδίκη συνολικά σε 150 χρόνια φυλάκισης. Βεβαίως, ο ίδιος ε, άνθρωπος εμφανίζεται και στην δολοφονία του Βάλτερ Λούπκιο και είχε επαφές με τον ε, δράστη και βεβαίως ε, η δίκη κατά του κόμματος N5 διακόπηκε γιατί θα φαινόταν ακριβώς στην δίκη ποιος είναι πραγματικό μέλος αυτού του κόμματος και ποιος είναι αζάν προβοκατέρ των μυστικών υπηρεσιών. Θα πρέπει λοιπόν να μην υποτιμούμε τον δεξιό εξτρεμισμό, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια εργαλειοποίηση από τις μυστικές υπηρεσίες του γερμανικού κράτους που αποτελούν κομμάτι του. Σας ευχαριστώ, Σαϊμπή, για ένα λεπτό. Καταρχάς, ε, θα ήθελα ε, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στα θύματα ε, που ε, δολοφονήθηκαν από έναν ακροδεξιό και τα συλληπιτήριά μου προς τις οικογένειάς τους. Μιλάμε για μια ακροδεξιά τα τελευταία χρόνια η οποία σπρώχνεται από το μίσος. Υπάρχει ο Ζουλιάνο Ντούλ ο οποίος συμμετείχε σε ένα φόνο που σκότωσε την κόρη του απλώς και μόνο γιατί φορούσε ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τι έγινε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ε, λέγεται Ρίξ Ζεμούρ ε, και έχει καταδικαστεί για πρόκληση ρατσιστικού μίσους, τα μετέδωσε όλα αυτά σε μία εκπομπή. Εγώ βρίσκομαι αριστερά του ημικυκλίου και βλέπω πολύ καλά αυτούς που βρίσκονται στην άκρα δεξιά του ημικυκλίου, διότι βρίσκονται ακριβώς μπροστά μου. Είναι αρκετοί, φυσικά. Αλλά δεν θα πρέπει εδώ να εκλεκεύουμε την παρουσία τους. Θα πρέπει να ακούγονται απόψεις αλλά δεν θα πρέπει ε, να αντισταθούμε στο μύθος, με, μίσος με τη διάθεση να συμβιώσουμε όλοι μαζί. Ε, επιθέσεις σαν αυτές του Χάλε σε αυτή την περίπτωση δεν θα ξανασυμβούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντυπών για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, 9 Οκτωβρίου πριν από λίγες μέρες είχαμε μια αιματηρή επίθεση στο Χάλε. Τα ακούσαμε ήδη πολλές φορές, δολοφονήθηκαν οι άνθρωποι, δύο άλλοι τραυματίστηκαν κοινικά και στοχευμένα επέλεξε το Γιόμ Κιπούρο ο δράστης για να επιτεθεί. Στη Γερμανία τα σχετικά δικήματα αυξήθηκαν κατά 40% το 2018 σε σχέση με το 2017. Ξεκινάνε με λεκτικές επιθέσεις και καταλήγουν όπως βλέπετε μέχρι και σε φόνους. και χρησιμοποιούν το ίντερνετ για να διασπείρουν τα λόγια τους. Υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που καθορίζουν την ταυτότητά τους με το να ταπεινώνουν και να αποκλείουν άλλους. Αυτά βλέπετε ότι εκτροχιάστηκαν στο Χάλε. 9 στους 10 Ευρωπαίους Εβραίους έχουν την αίσθηση ότι ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί. Αυτό είναι βεβαίως αφορμή για ανησυχία αλλά και για να δράσουμε. Τα προληπτικά μέτρα είναι σημαντικά, αλλά προφανώς δεν επαρκούν. Δεν πρέπει να επιδείξουμε ανοχή σε αυτούς οι οποίοι επιχειρηματολογούν με μίσος. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για αυτή την πάρα πολύ σημαντική συζήτηση και ελπίζω να κινηθούμε μαζί κατά του μίσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον συνάδελφο τον κύριο Μπράιερ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε λόγω μίσους κατά κάποιων ανθρώπων και μειονοτήτων συχνά δολοφονούνται άνθρωποι. Απέναντι στο μίσος θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να είναι ενωμένοι και να υψώσουν το ανάστημά τους. Αντί να λέμε ότι φταίνε όλοι οι χρήστες του ίντερνετ ή οι γκέιμερ. Η απάντηση της ε, πολιτικής θα πρέπει να είναι περισσότερη δημοκρατία και συμμετοχή στην πολιτομία, πιο ανοιχτή κοινωνία και περισσότερη ανθρωπιά. Αντί να ξεκινάμε τώρα με σχέδια παρακολούθησης ε, ή απαγόρευσης της ανωνυμίας ε, στο δίκτυο που δεν θα μπορούσαν να έχουν σταματήσει τον δράστη του Χάλε. Πρέπει επιτέλους να επενδύσουμε στην κοινωνία των πολιτών ε, για να καταπολεμηθεί το μίσος, να υπάρξει μια καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο, να ε, υπάρξει μια δίωξη της σχετικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο και εκτός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ξοδέψουμε λεφτά σε αποθήκευση δεδομένων. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς κατά της βίας αλλά ποτέ να μην παραβαίνουμε τις αρχές μας. Αλλιώς οι τρομοκράτες θα έχουν κερδίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί η κυρία Σαρντόνα για ένα λεπτό. Είμαστε σίγουρα όλοι πολύ κοντά στην εβραϊκή κοινότητα για τα όσα συνέβησαν στη Γερμανία. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο, το οποίο σίγουρα πρέπει να καταδικάσουμε και εμεί είμαστε κατά οποιασδήποτε μορφή βία και ρατσιστικού ή θρησκευτικού εγκλήματο. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο αναρωτιέμαι πώ μπορεί η Ευρώπη να σιωπά. Ε, και για άλλα επεισόδια που συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες. Τον Οκτώβριο στο Παρίσι ένας άνδρας σκότωσε τρεις αστυνομικούς με μαχαίρι. Ήταν ε, Ισλαμιστής, φονταμενταλιστής και τον αναζητούσαν για ε, πρόκληση τρομοκρατίας. Και επίθεση σε κέντρο εμπορικό είχαμε και στο Μιλάνο την πόλη μου ένας ε, παράνομος μετανάστης μαχαίρωσε έναν αστυνομικό, ένα στρατιωτικό συγγνώμη, φωνάζοντας Αλάχ Αχμπάρ. Γιατί δεν μιλάμε λοιπόν για τον αντισημιτισμό στη Γαλλία δεν μιλάμε για την ε, τρομοκρατία και τον Ισλαμιστικό φονταμενταλισμό σε περιοχές και γκέτο όπου ε, ανθεί ο φονταμενταλισμός του Ισλαμισμού και ε, γιατί δεν μιλάμε και για την παρέμβαση της Τουρκίας στην Συρία. Εγώ θα ήθελα η Ευρώπη να ασχοληθεί και με αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε μπλε κάρτα, τη δέχεστε? Από τον κύριο Πόκαμ. Παρακαλώ, 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Τα συλληπιτήρια για την εβραϊκή κοινότητα αρκούν για 30 δευτερόλεπτα και μετά όλα τα υπόλοιπα τα έχετε αφιερώσει στον εξτρεμισμό άλλης φύσεως. Ε, πώς εκφράσατε, ας πούμε, εσείς τα συλληπιτήριά σας εδώ. Μικρόφωνο, Please use your mic. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ λόγω πολιτικής νοοτροπίας πιστεύω ότι αυτό που έχει περισσότερο σημασία είναι να κρίνουμε τα γεγονότα και όχι τα λόγια. Γι' αυτό ακριβώς εγώ εδώ δεν κάνω διάκριση ε, όταν συζητούμε την τρομοκρατία. Ο τρομοκρατίας δεν έχει χρώμα και έχω την απέτηση όμως η Ευρώπη να σταματήσει τα λόγια και να αρχίσει να δρά. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Περνάμε τώρα στο Catch the Eye. Δεν θα δεχτώ εδώ πέρα ε, μπλε κάρτες για να μπορέσουν να μιλήσουν όσο δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Συνεχίζουμε με την ε, κυρία Αντάμοβιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τα πρόσφατα γεγονότα στη Χάλεπ μας έδειξαν ε, σε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Πραγματικά ε, μας δείχνει ότι στην κοινωνία μας επικρατεί η εχθρότητα και αυτή η ρητορική του μέσου με οδήγησε να ασχοληθώ με την πολιτική δεν πρόκειται μόνο για ρατσισμό, ομοφοβία, αντισημιτισμό ή τρομοκρατία. Εδώ απειλείται η δημοκρατία. Πρέπει να χαράξουμε σύνορα μεταξύ της ελευθερίας εκφρασής και της ρητορικής μίσους. Ως νομοθέτες θα πρέπει να θέσουμε φιλόδοξους στόχους για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και online και offline. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες ε, του λόγου αυτού για την κοινωνία. Θέλω επίσης ε, να τα υπογραμμίσω όλα αυτά βάσει και της προσωπικής μου εμπειρίας. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι, υπόθηκε αυτό. Δεν μπορούμε την ευθύνη αυτή να την παραπέμπουμε ένα στον άλλο. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι, το υπογραμμίζω και μπορούμε να φτιάχνουμε τείχους, μπορούμε να καταδικάζουμε και να κατηγορούμε την αστυνομία και να λέμε ότι η αστυνομία αυτή που δεν έκανε τη δουλειά της, μπορούμε να φτιάξουμε και τείχη γύρω από τις συναγωγές, αλλά δεν αντιμετωπίζουν αυτά. Κονσάλης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ο βίαιος ε, ακροδεξιός εξτρεμισμός ε, που είδαμε στον Οκτώβριο στο χάλε, μας ε, υπενθυμίζει ότι ο μουσουλμανικός λαός ή ε, η ευρωϊκός λαός ή μετανάστες ή οι ΛΟΑΔΜ μπορεί να είναι αυτοί που υποφέρουν από τη ρητορική μίσους. Όμως δεν έχει κανένα νόημα να εκφανούμε εδώ λόγους για τις ευρωπαϊκές αξίες αν κατόπιν ε, στα κράτη-μέλη μας τότε κάνουμε συμφωνίες με αυτά τα κόμματα της δεξιάς ε, που υπερασπίζουν τη ρητορική μίσου. Και σε πάρα πολλέ κοινότητε και Δήμου ε, στην Ισπανία αυτοί που βγάζουν εδώ τέτοιου μεγαλόστομους λόγου, έρχονται και κάνουν συμφωνίε ε, με αυτά τα κόμματα. Πρέπει να δώσουμε πόρους στην τοπική αυτοδίκηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και μέσω του Ταμείου Συνοχής για την πρόληψη. Χωρίς την πρόληψη δεν θα καταπολεμήσουμε τη ρητορική του μίσου, θα υπερασπίσουμε την Ευρώπη και τη συμβίωση. Γιατί ε, ε, προλαβαίνουμε ακόμη να δράσουμε. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Φερέρα για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ο βίος ακροδεξιό εξτρεμισμός που εκφράστηκε μέσω των επιθέσεων του Χάλε θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να καταπολεμηθεί όμω, συνειδητοποιώντα ότι έχουμε ε, μια διαδικασία ριζοσπαστικοποίηση της ακροδεξιάς και του φασισμού στην Ευρώπη. Ε, αυτά συνδέονται με πολιτικές που επιτίθεται σε κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα, στην εθνική κυριαρχία και στη δημοκρατία. Οι πολιτικές που εξυπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο που προκαλούν κοινωνική αδικία και τις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά σχετίζονται. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί έναν επικίνδυνο ιστορικό ρεβιζιονισμό ε, και ε, βλέπουμε μια αξιοθρύντη προσπάθεια να εξισωθεί ο κομμουνισμός, ε, με το φασισμό και ε, φαίνεται σαν να εξομοιώνονται και τα θύματα και απαξιώνεται ο γόνος των κομμουνιστών υπέρ της ελευθερίας. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε καμία τέτοια ιδεολογία. Ευχαριστώ συνεχίζουμε με τον κύριο Ολρίχη Για ένα λεπτό. Όλες ε, οι μορφές του εξτρεμισμού θα πρέπει να καταδικάζονται. Ε, όταν κάποιος ε, πυροβολεί οικογένειες με παιδιά, μάλλον είναι τρελός. Όμως γιατί μιλάμε μόνο εδώ για ακροδεξιό εξτρεμισμό, σαν μην υπάρχουν άλλες μορφές εξτρεμισμού, γιατί δεν μιλάμε για τους τζιχαντιστές ε, ή για τους ακραίους Ισλαμιστές που διαπράττουν εγκλήματα στην Ευρώπη, διαπράττουν τρομοκρατικές επιθέσεις ε, και έχουμε και διάφορες ε, ζώνες γκέτο που δεν μπαίνει ούτε καν η αστυνομία. Γιατί δεν ε, μιλάμε για τα θέματα αυτά και γιατί δεν μιλάμε και για κινήματα αντιφασιστικά που, που επιτέθηκαν ακόμη και σε κάποιους συναδέλφους στη Σλοβακία και μάλιστα επιτέθηκαν στην περασμένη εβδομάδα σε μια γυναίκα Σλοβακία γιατί δεν συμφωνούσε με την άποψή τους. Πόλτσεκ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ για το λόγο. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτηριά μου στους συγγενείς των θυμάτων. Είναι τεράστιο πρόβλημα ο εξτρεμισμός στην Ευρώπη και δεν έχει σημασία αν μιλάμε για ακροδεξιό, ακροαριστερό εξτρεμισμό. Εδώ μιλάμε για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ας δούμε τι γίνεται. Κάποιες ε, ομάδες Εβραίων φοβούνται να πούν ότι είναι Εβραίοι. το χάρη, εδώ στη Γαλλία, πολλοί άνθρωποι νέοι σήμερα δεν ξέρουν τι ήταν το ολοκαύτωμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε το ολοκαύτωμα και κάνουν και διαλέξεις σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ολοκληρώνουμε με τον κύριο Πάτεν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι στην αίθουσα, Θεωρώ ότι η φωνή στο Χάλε είναι φρίκη και πραγματικά εκφράζω τα βαθιά μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Να υπενθυμίσω όμως ότι την προηγούμενο μήνα συζητήσαμε την ημέρα μνήμης ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια κοινή ιστορική ε, αφήγηση. Ο κύριος Φέστ που καθόταν εκεί μας υπενθύμησε ότι ξεχάσαμε να θυμηθούμε και το ολοκαύτωμα και πρότεινε μια τροπολογία η οποία συμπεριλήφθηκε στο ψήφισμα. Και παρά το γεγονός ότι υπήρχε ε, υποστήριξη και από αυτή την πλευρά και πολλούς ε, άλλους ευρωβουλευτές, πολλές ομάδες της αριστεράς το απέρριψαν και δεν πέρασε η τροπολογία. Τι μήνυμα στέλνει κάτι τέτοιο όταν το ίδιο το Κοινοβούλιο της Ευρώπης ε, γυρίζει την πλάτη του στην ανάμνηση του ολοκαυτώματος. Δεν πρέπει απλώς να μιλούμε. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι δράσεις μας και οι πεπιθήσεις μας ε, μετρούν και εδώ στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για να κλείσουμε ο λόγος στον Επίτροπο Κίνγκ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που συμβάλλατε σε αυτή τη συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η συζήτηση για τα θέματα τα οποία ετέθησαν σήμερα. Υπάρχουν ε, και άλλες περιπτώσεις οι συζητήσαμε τον αντισημιτισμό και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να τον αντιμετωπίσει. Το έχουμε συζητήσει επί μακρόν με τον συναδέλφους μας, τον Φραν ε, Τίμερ και τη Βέρα Γιούροβα και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό και να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον ακραίο εθνικισμό. Διότι αυτά είναι εκβάθρον αντίθετα στις κοινέ μα αξίες. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε το βίο εξτρεμισμό. Και το είπα και στην αρχή της συζήτησης και θα το πω και στο τέλος της συζήτησης. Ο βίος εξτρεμισμός ανεξάρτητα από την πηγή του. Μπορεί να είναι ακροδεξιός ε, βίαιος μπορεί να είναι ακροαριστερός, ε, τζιχαντιστικός εξτρεμισμός. Δεν κάνω διάκριση εγώ μεταξύ τους. Πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε το βίαιο εξτρεμισμό. Συμφωνώ με εκείνους που αναφέρθηκαν στην ανάγκη να επικεντρωθούμε στην πρόληψη να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το μίσος και τη βία. Και θα πρέπει κάτι τέτοιο να γίνει μέσω της εκπαίδευσης, θα πρέπει να γίνει και μέσω της αποτελεσματικής μας δέσμευσης με την κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή με τις τοπικές κυβερνήσεις, με τους δασκάλους, αλλά και με τους αστυνομικούς ε, και ε, τους φύλακες ε, στις φυλακές και ε, όλους αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Και θα πρέπει να συνεργαστούμε ως τμήμα αυτής της προσπάθειας και με τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτό είναι το όχημα και ο φορέας ο οποίος εξαπλώνει και επιταχύνει όλη αυτή την μισητή βία και το παράνομο περιεχόμενο. Και δεν γίνεται γιατί έχω κάποιο πρόβλημα με τις πλατφόρμες ε, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι και αυτές αντικείμενο κατάχρησης ε, και εξαπλώνεται έτσι το μίσος και το παράνομο περιεχόμενο. Αλλά πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους. η βία δραστηριότητα η εξτρεμιστική στο Χάλε την οποία συζητήσαμε σήμερα έγινε με σχολιασμό στα αγγλικά ήταν σχεδιασμένη για να διαβιβάσει ένα μήνυμα και να το εξαπλώσει σε όλες τις χώρες μας και ίσως και πιο πέρα ένα βίαιο μήνεσμα μίσους, διότι μετά από τα όσα συνέβησαν στο Christchurch ε, αντλήσαμε κάποια διδάγματα και εφαρμόστηκαν και το είπε και κάποιος εδώ στη συζήτηση. Μόνο μισή ώρα μετά από αυτή τη ζωντανή μετάδοση ε, είχε πέσει, ε, αφαιρέθηκε το περιεχόμενο. Δηλαδή, το είδαν κάποιοι ζωντανά, αλλά ήταν σχετικά μικρός αριθμός. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξαπλώνεται. Εξαπλώθηκε σε διάφορα κανάλια, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε διάφορα φόρουμ ε, και μπορεί ακόμα να το δει κάποιος αυτό το περιεχόμενο, όπως μπορεί κάποιος να δει περιεχόμενο από το, την επίθεση στο Christchurch, που σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους να συνεργαστούμε με τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να αντιμετωπίσουμε και να διαγράψουμε τέτοιο περιεχόμενο γιατί δηλητηριάζει ε, τα μυαλά των ανθρώπων. Και πραγματικά, όπως και κάποιοι από εσά, πιστεύω ότι οι αξίες μας είναι η δύναμή μας και θα πρέπει να προχωρούμε με τα πιστεύω μα όσο προωθούμε αυτή τη μάχη κατά της βίας και του μίσους και του ακραίου εξτρεμισμού. Και οι αξίες αυτές θα μας βοηθήσουν να την κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συνεχίζουμε με το επόμενο. Δήλωση της Κομισιόν για την ποινικοποίηση της σεξουαλικής αγωγής στην Πολωνία. Έχετε μεγάλη ζήτηση σήμερα κύριε Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ναι, ναι, κοιτάω τον τίτλο. Να περάσαμε. Ναι, ναι, περάσαμε. Δεν έχει ανέβει ακόμα ο καινούριο τίτλος αξιότιμα κύριοι βουλευτές του Κοινοβουλίου. Κάλεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια δήλωση για την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία. Από όσο γνωρίζω, δεν ισχύει αυτή τη στιγμή τέτοια νομοθεσία και η Κομισιόν δεν σχολιάζει σχέδια νόμου. Όμως μπορούμε μόνο να σημειώσουμε ότι λυπούμαστε ότι χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να συζητήσουμε αυτό το θέμα απόψε. Σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική πολιτική, όπως γνωρίζετε, το άρθρο 165 της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θεσπίζει ότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για το περιεχόμενο και την οργάνωση των εκπαιδευτικών του συστημάτων. Λεχθέντος αυτού, η Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αυτά είναι μέρος της διδασκαλίας. Δηλαδή, ε, μία πύλη ε, της Ευρώπης ε, για τους Χαράκτε τη πολιτικής, ε, του δασκάλου και του εμπειρογνώμονε ε, έχει ξεκινήσει μια δημοσκόπηση για το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τι απόψει ε, των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο συγκεκριμένο κλάδο. Η έρευνα είναι ανοιχτή μέχρι τις 20 Νοεμβρίου και είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες και τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν ε, στην ε, πύλη αυτή της σχολικής εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά τώρα το ποινικό δίκαιο και πάλι όπως γνωρίζετε, το άρθρο 83 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θεσπίζει ότι η Ένωση έχει αρμοδιότητα όταν υπάρχει σοβαρό έγκλημα διασυνοριακής φύσης. Τώρα, εδώ ε, έχουμε το αδίκημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και γυναικών. Όπως γνωρίζετε, η οδηγία 2011-93 περικοπεί την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη-μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευση και κατάρτιση για να αποθαρρύνουν και να μειώσουν την ζήτηση ε, που προωθεί τη μορφή κάθε ε, σεξουαλικής εκμετάλλευση παιδιών. Παραδείγματα μπορούμε να έχουμε, ε, είναι τα εξή εκστρατείε για τι συνέπειε, παραβίασης του νόμου, καθώς και βραχυπρόθεσμη και μικροπρόθεσμη βλάβη ε, σε όσους εμπλέκονται στα θύματα η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητές της δυνάμει των συνθήκων για να διασφαλίσει ότι η οδηγία αυτή θα εφαρμοστεί πλήρως και σωστά. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το να διασφαλίσουμε ότι η εθνική νομοθεσία δεν εμπλέκεται με, την, με το στόχο της οδηγίας, δηλαδή την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάει η συζήτηση με την κυρία Λουκατσιεβισκα για το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι και εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι που πρέπει να συζητήσουμε εδώ στο ημικύκλιο την σεξουαλική διαποδαγώγηση στην Πολωνία ώστε τα παιδιά στην Πολωνία να μπορούν να έχουν όπλα για να αντιμετωπίσουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ε, ή σεξουαλικές επιθέσεις. Ο Πάπας είπε ότι το σεξ είναι δώρο Θεού και πρέπει να υπάρχει σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία και ο Πάπα ε, το είπε έχοντας το νου του στις νέες γενιές. Ε, δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι τη σήμερα ημέρα στην Πολωνία η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα πολωνικά σχολεία θεωρείται κάτι ύποπτο. Ε, πρέπει να πω ότι σύμφωνα με κάποιους, εάν ε, δεν υπάρξει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για τα παιδιά μας, θα τα προστατεύσουμε από την παιδοφιλία. Και πραγματικά η κυβέρνησή μας ε, κοφεύει ε, σε όλα τα ουσιαστικά επιχειρήματα. Και τι γίνεται, όλο ένα και περισσότερα άτομα ε, πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδεδόμενες ασθένειες και υπάρχουν και εγκυμοσύνες σε κορίτσια κάτω των 15 ετών. Και υπάρχουν όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι που αυτοκτονούν γιατί είναι θύματα ε, και μίσους. 13.500 ε, παιδιά στην Πολωνία το 2018 ήταν θύμα σεξουαλικής βίας. Και μόνο μέσω της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι θα ξεκινούν τη σεξουαλική τους ζωή αργότερα και θα έχουν ε, και κατάλληλα όπλα ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις και να μην πέσουν θύμα βιασμού ή απόπειρα να ξεκινήσουν νωρίτερα τη σεξουαλική του ζωή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συγκατάθεση, να γνωρίζουν τα παιδιά τη σεξουαλικότητά τους ε, και να μπορούν να ξέρουν και τι γίνεται με την αντισύλληψη. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την παιδοφιλία. Δεν πρέπει σήμερα να επιτρέψουμε στα παιδιά στην Πολωνία να υποχρώνονται να λαμβάνουν πληροφορίες για τη σεξουαλική ζωή μόνο μέσω πορνογραφικού υλικού που μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ. Μπιεντρών για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε στο 2019, αλλά η συζήτηση φαίνεται να είναι του μεσαίωνα. Η παρούσα ε, κυβέρνηση της δεξιάς ε, στην Πολωνία υπέβαλε την τροπολογία του σχεδίου νόμου όσον αφορά την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης την περασμένη Τετάρτη. Ε, δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου το οποίο υπαγορεύεται από τα λόμπι των παιδόφιλων. Διότι προβλέπει κόλαση για τα θύματα και τον ουρανό για τους παιδόφιλους ποινικοποιείται οποιαδήποτε συζήτηση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Εάν ο Επίτροπος ε, έκανε την ομιλία του μετά από την ε, έγκριση αυτής της νομοθεσίας ε, στην Πολωνία, θα μπορούσε να λάβει και ποινή πέντε ετών φυλάκισης. Στην Πολωνία μπορεί κάποιος να φυλακιστεί για πέντε χρόνια για κλοπή ή για συζυγική βία. Έχουμε δηλαδή την ίδια ποινή και την ίδια ποινή τώρα θα επιβάλλουμε και στον παιδαγωγό ή στο γιατρό ο οποίος θα αναρτήσει στο διαδίκτυο ένα βίντεο για την αντισύλληψη. ή εάν στη διάρκεια ενός μαθήματος στο σχολείο ο δάσκαλος ε, παρουσιάσει στους νέους μαθητές ένα βίντεο για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και μπορεί στη συνέχεια ο καθηγητής να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Εάν λοιπόν δεν επιδείξουμε αλληλεγγύη, δεν ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, θα έρθουν και μας να μας ε, καταδικάσουν. Πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε αυτή τη βλακώδη μεσαιωνική ιδέα. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την κυρία Σήματσικα για το Ρηνίο για δύο Ευχαριστώ. Οι προτινόμενες αλλαγές στο ποινικό δίκαιο στην Πολωνία που de facto ποινικοποιούν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών δεν είναι παράδειγμα ε, κάποιες ε, ιδεολογικής πρότασης, ε, απλώς τίθεται και κατά των βασικών αρχών της σύγχρονης εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο στον 21ο αιώνα να απειλούνται οι καθηγητές με ποινή φυλάκισης επειδή θα εξηγούν στους νέους πώς να χρησιμοποιούν τα προφυλακτικά. Συνήθως κυβερνήσεις παγκοσμίω επενδύουν στην εμόρφωση σε μια εκπαίδευση που δίνει τα απαραίτητα εφόδια στα παιδιά ε, για να ε, μπορέσουν να ανταπεξελθούν στους προκλειστές ζωής. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Στερούνται τα παιδιά ε, το δικαιώματός τους αυτού. Οι εμπνευστές της νομοθεσίας είπαν ότι θέλουν να προστατεύσουν ε, τους ε, νέους ε, και τα παιδιά. Όμως το πρόβλημα είναι ότι ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί, γιατί χωρίς την κατάλληλη γνώση για πιθανή κακοποίηση από την πλευρά των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί η σεξουαλική βία γιατί αποτελεί αυτό τελικά πρόσκληση για τους ε, παιδεραστές και οποιαδήποτε απόπειρα απαγόρευσης της σεξουαλικής ε, διαπαιδαγώγησης ε, θα είναι εις βάρος της ασφάλειας των παιδιών. Η άλλη αρνητική συνέπεια θα είναι να αποθαρρυνθούν οι δάσκαλοι από το να κάνουν τη δουλειά τους καθώς έχουμε αυστηρές ποινές. Αυτό θα στείλει ένα πολύ άσχημο μήνυμα σε όλο τον κλάδο και θα δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου και διώξεων εσως Ίσως ε, ε, κάποιοι όπως πρότειναν ότι δεν θα εφαρμοστούν ε, αυτές οι σκληρές ποινές και θα υπάρξει συντηρητική ερμηνεία του νόμου όμως δεδομένης της επιθετικής εκστρασίας που είδαμε και κατά τον ΛΟΑΔΜΑ στην Πολωνία τους προηγούμενους μήνες είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε σε αυτές τις διασφαλίσεις. Έτσι λοιπόν εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλύτερο αν αποσυρθεί η πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Δύο λεπτά ο κύριος Άντρεσεν, εκ μέρους ε, των Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Διαφορετικής Συμμαχίας. Ο κόσμος πρέπει να έχει δικαίωμα να μάθει για την αγάπη, για τη σεξουαλικότητα. Όταν έχουν ερωτήσεις για το φίλο τους, για τη σεξουαλικότητά τους, χρειάζονται απαντήσεις και η επιστήμη μας λέει ότι ήδη από την ηλικία των 12 ή των 13 νέοι αρχίζουν να διερωτώνται για τη σεξουαλικότητά τους, για το σώμα τους, για την αγάπη των έρωτα. Είναι σημαντικό λοιπόν να πάρουν απαντήσει νέοι να μάθουν την αγάπη, να λένε ναι, να λένε όχι, να έχουν αυτοπεποίθηση. Το καλύτερο λοιπόν είναι να έχουμε δημόσια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, γιατί αν την απαγορεύσουμε από τα σχολεία, οι νέοι θα ρωτούν άλλου ε, ή ε, θα ντρέπονται. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε του δημόσιου εκπαιδευτικού ε, και να προωθηθεί η δημόσια σεξουαλική αγωγή. Πρέπει να προωθήσουμε ανθρώπινα δικαιώματα για όλου, για τι γυναίκε, για του ΛΟΑΔΜ, για όλου όσου θέλουν να ζουν σε ελευθερία. Η πολιτική κυβέρνηση δημιουργεί φόβο και δεν υπάρχει κάτι χειρότερο να τρομάξει κανείς ε, το νέο άνθρωπο όταν δεν μπορεί να ε, νιώθει ελεύθερα με τον έρωτα με τη σεξουαλικότητά του και σίγουρα οι ομοφιλόφιλοι και, και τα νερά κορίτσια θα πληγούν περισσότερο οι ομοφιλόφιλοι είναι τα θύματα της σεξουαλικής βίας ε, και αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και από νεαρή ηλικία και στην Πολωνία θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα, αλλά και σε όλα τα άλλα κράτη που κάνουν αντίστοιχα. Δεν θέλουμε ιδιωτική μεταχείριση σε βάρος των νεαρών οφειλοφίλων, νεαρών κοριτσιών στην Πολωνία. Είναι σημαντικό. Εμείς οι πράσινοι στεκόμαστε αλληλέγγυοι με το ομοφιλόφιλο κίνημα, με όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους λέμε δεν είστε μόνοι σας, έχετε δικαιώματα, είμαστε στο πλευρό σας. Η πολωνική κυβέρνηση μπορεί να αποφασίζει να απαγορεύει σεξουαλική αγωγή, αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν βουλευτέ που στηρίζουν ε, τη νεολαία στην Πολωνία. Ευχαριστούμε. δύο λεπτά, εκ μέρου ε, τη ομάδα ID. Ναι, ευχαριστώ. Καλησπέρα σα. Σήμερα μιλάμε για την υποθέμενη ποινικοποίηση τη σεξουαλική αγωγή στην Πολωνία, αίτημα τη πολωνική αντιπολίτευση να μπει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ουσιαστικά ε, πρόκειται για μια δημοκρατική νομοποιημένη κυβέρνηση, την οποία γίνεται μια απόπειρα να την ε, απαξιώσουν κάποιοι σε σχέση με αυτά τα θέματα. Κάποιοι οποίοι μπορεί να διαφοροποιούνται ως προς την τοποθέτησή τους. Αυτό όμως είναι όνειδος. Μπορεί κανείς να έχει διαφορετικές απόψεις ε, για το κατά πόσο η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνει οι η δημόσια εκπαίδευση. Το θέμα είναι ε, τα παιδιά στο δημοτικό μπορούν να μιλούν για, και να μαθαίνουν πράγματα για παραφύση, σεξουαλική επαφή και τα Ε, πώς μπορούμε να το αποφασίσουμε αυτό. Ε, υπάρχει ένα σχέδιο ανάλογο σεξουαλικής αγωγής ε, στην ε, Γερμανία ε, που μπορεί κανείς κρατά τα μάτια να ψηλαφεί το σώμα τους. Ε, ε, όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων. Είναι κάτι αειδιαστικό. Ε, είναι μια προσπάθεια σεξουαλικοποίησης των παιδιών μας από την αρή ηλικία. Και τα παιδιά δεν μπορούν να χάσουν την αθωότητά τους τόσο νωρίς. Ε, γιατί και οι παιδεραστές ε, ουσιαστικά θα έχουν ανοιχτά τα παράθυρα και τις πόρτες ε, για να κακοποιούν και να βιάζουν ανηλίκους. Και βλέπουμε ότι και η αριστερή αυτή, η αδιαστική αυτή εκστρατεία διακόπτεται. Η Πολωνία έχουν μια κυβέρνηση. Πρέπει λοιπόν αυτούς τους έκφυλους ε, και διαστραμμένους αριστερούς να μην τους αφήσουμε να επηρεάσουν ε, τη θεμητή προσπάθεια της πολιτικής ε, κυβέρνησης. Ντροπή, ντροπή σας, δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Έσχος. I, uh, a blue card request. However... Uh, Διαπιστώνω ότι έχει ζητηθεί μια μπλε κάρτα, αλλά αυτά είναι, αυτές είναι ομάδες εκ μέρους πολιτικών ομάδων, άρα δεν δέχω, γίνονται δεκτές οι μπλε κάρτες. 1,5 λεπτό η κυρία Ζαλεύσκα. Εκ, μέρους του, της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, με θλίψη παρακολουθώ τη συζήτηση και τις φωνές που ακούγονται εδώ, γιατί μεταφέρονται ψεύδι. Παραδείγματο χάρη, ε, λέγονται ψέματα στην Κομισιόν και στους συναδέλφους γιατί η κυβέρνηση της Πολωνίας σε κανένα επίπεδο δεν, δεν προετοιμάζει νομοθεσία που θα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση όπως αναφέρθηκε στον Επίτροπο. Αυτό το οποίο επίσης είναι λυπηρό και εδώ υπάρχει μεγάλη σύγχυση είναι ότι υπάρχουν μέλη και έμπειρα όπως η κυρία Ουκατσιεύσκα που ψήφισαν στη συζήτηση ενώ είναι γνωστό ότι η ε, παιδεία και κυρίως η σεξουαλική παιδεία ε, είναι θέμα το οποίο ρυθμίζεται από τα κράτη-μέλη και όχι από την Ευρώπη. Και τέλος, έχουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ε, στην Πολωνία. Το 99 ήδη ε, συμπεριελήφθη στον νόμο για την παιδεία. Για όλα τα επίπεδα της παιδείας. Όμως, αυτή η διαπαιδαγώγηση ε, αντιλαμβάνεται τα παιδιά μαζί με άλλες ανάγκες όπως την συντροφική σχέση, την αγάπη, αυτοσεβασμό, σεβασμό του άλλου, αμοιβαίο σεβασμό και επίσης αντιμετώπιση κάποιων εξαιρετικών ή ακραίων ε, συνθήκων. Επίσης τα διδάσκει πώς να προστατεύονται από τις ιδέες που ε, προωθεί ο κ. Πυρός. Η κυρία Ροντρίγες Πάλοπ εκ μέρους της ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ. Το αποκαλούν stop παιδοφιλία, αλλά δεν είναι. Αυτό που η κυβερνήση της Πολωνίας θέλει να, ε, να κάνει είναι να ενοχοποιήσει την ε, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θέλει να συσχετίσει την σεξουαλική δαπαιδαγώγηση με την υποταγή. Ε, πρόκειται για μια πολιτική που ε, υποτιμά τις γυναίκες και προωθεί ε, την καταπολέμηση της, μάλλον και δείχνει την ομοφοβία. Θέλει η υπερκαθολική κυβέρνηση να περιορίσει τα δικαιώματα. Υπάρχει πολύ ε, μεγάλο ποσοστό ε, νέων ε, με το νιό του HIV. Η κυβέρνηση θέλει να περιορίσει τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα παιδιών, των παιδιών, κοριτσιών και αγοριών και να περιορίσει και τα δικαιώματα των γυναικών. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό. Η κυρία Φιτζέραλτ. Ευχαριστώ. Πριν από δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες συναντήθηκα με μια ομάδα κοριτσιών ε, στο πλαίσιο της ομάδας ε, για τα κορίτσια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συζητήσαμε για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται και το είδος της διαπαιδαγώγησης που είχαν διδαχθεί στο σχολείο. Καμιά δεν μπόρεσε να μου πει ότι είχε διδαχθεί ολοκληρωμένα ε, το θέμα του σεξ. Αυτό πρέπει να το προχωρήσουμε. Αν θέλουμε ισότητα των φίλων στην Ευρώπη, πραγματική ισότητα όπου οι γυναίκες, τα γόρια και τα κορίτσια καταλαβαίνουν τις αξίες και την ισότητα, πρέπει να προωθήσουμε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ό,τι να την εμποδίσουμε. Πρέπει να ε, διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά, όπως γνωρίζω από την, Ιταλία, από την Ιρλανδία, μάλλον η έλλειψη διαπαιδαγώγησης παρά η ίδια η διαπαιδαγώγηση που οδηγεί σε ε, άσχημες συνέπειες. Και τι συμβαίνει. Εμποδίζεται η διαπαιδαγώγηση, περιορίζεται η γνώση του τι σημαίνει ε, σεξουαλική κατάχρηση και τελικά ε, ε, υπονομεύονται τα θεμελιώδη, οι θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας μας. Πρέπει να διδάξουμε την σεξουαλική ζωή στα παιδιά και αυτό ότι είναι απολύτως ανοησία ότι αυτό μπορεί να διευκολύνει την ε, παιδοφιλία. Αντιθέτως θα βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν και να κατανοήσουν τι εστί σεξουαλική βία και η στέρηση αυτής της διαπαιδαγώγησης τα κάνει ευάλωτα όχι μόνο τότε αλλά σε ολόκληρη τη ζωή τους και δεν νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός της διαπαιδαγώγησης ε, με απλά μέσα. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να είναι προσεκτικά και υπεύθυνα όταν ε, αποφασίσουν να προχωρήσουν και πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσουμε από την πολωνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το ηλεκτρονικό σύστημα για τα αίτημα της μπλε κάρτας έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Τώρα, για δύο λεπτά η κυρία ε, Ρέγνα. Ευχαριστώ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το κατά πόσον θα το κάνουν αυτό οι δάσκαλοι στην Πολωνία ε, για να υπάρχει μια υγιή σχέση των νέων με το σώμα τους, με τη σεξουαλικότητά τους. Ε, είναι κάτι ε, που αν το κάνουν μπορεί και να πάνε πέντε χρόνια φυλακή οι δάσκαλοι. Αυτό είναι πραγματική ντροπή και πρέπει στεναρά να αντισταθούμε σε αυτή την πολιτική. Αυτό το οποίο χρειάζεται στην Ευρώπη είναι περισσότερη ανοιχτή διαπαιδαγώγηση και σεξουαλική σεξουαλική αγωγή πρέπει να είναι ένα μάθημα ε, για τους νέους ε, και αυτό είναι και ο στόχος μας. Ε, μία από τις βασικές απαιτήσει της επόμενης διάσκεψης κορυφής, του επόμενου μήνα στο Ναϊρόμπι, είναι ακριβώς η πρόσβαση σε δημόσια σεξουαλική αγωγή. Θέλουμε λοιπόν πρόοδο και όχι οπισθοδρόμηση. Είμαστε κατά λοιπόν αυτής της υποβάθμισης των δικαιωμάτων γενικών και των νέων. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση των ε, πολωνικών αρχών να απαγορέψουν και να ποινικοποιήσουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι κόντρα στον καιρό ε, το να ανατίθεται η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε, ε, στην πορνογραφία είναι αντίθετη με τις αξίες. Είναι ένα οξύμορο το οποίο δεδομένου ότι η Πολωνία έχει συνυπογράψει την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή κατά κάθε διάκριση κατά της γυναίκας, αλλά και άλλες διεθνείς συμβάσεις κατά των, ε, των φιλετικών διακρίσεων. Ναι, θα πρέπει να μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και να συζητήσουν ε, τα διάφορα ζητήματα που αφορούν το φύλλο η παιδεία, η διδαχή, η εφαρμογή της των παιδαγωγικών μεθόδων σε μια βασική ε, πτυχή της ανθρώπινης ε, κατάστασης όπως είναι η σεξουαλικότητα είναι ωφέλιμη. Ε, αντίθετα είναι ακατανόητο το να απαγορεύεται να συζητώνται αυτά τα θέματα. Στην Ναβάρα, μια περιοχή της Ισπανίας, η αντιδραστική δεξιά ήθελε να βγάλει από τα σχολεία ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο καταπολεμούσε τα στερεότυπα του φύλου και το οποίο βραβεύθηκε από πολλούς διεθνείς οργανισμούς όπως και από την UNESCO. Σας ζητώ να προβληματιστείτε. Μιλάμε για παιδεία, για ελευθερία, για διαπαιδαγώγηση. Βρισκόμαστε στην Ευρώπη. Το να τιμωρούνται τέτοιου είδους προγράμματα είναι ενάντια στην ιστορία και κατά των ίδιων των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα. Ε, από την κυρία Ζαλεύσκα για σας. Τε δέχεστε? Δέχεστε την μπλε κάρτα? Μάλιστα. Δεν τη δέχτηκε η κυρία Βιλμπάου Μπραντίκα. Γιάκη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάτε για ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, αλλά κανείς από εσά δεν διάβασε καν αυτό το νομοθέτημα. Εσείς διαδίδετε ψευδείς πληροφορίες. Εγώ διαβάζω αυτό το νομοθέτημα αυτή τη στιγμή. Άρθρο 1. Οποιοςδήποτε δημόσια προωθεί ή εγκρίνει συμπεριφορά παιδοφιλική θα ε, υπόκειται σε πρόστιμο την ποινή της περιορισμού της ελευθερίας του ή την ποινή της στέρησης της ελευθερίας του για μέχρι δύο χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ποινικοποίηση της παιδείας, αλλά παγόρευση της πρόθεσης της παιδοφιλίας, που είναι παρούσα σε περισσότερες, στους περισσότερους ποινικού κώδικες των κρατών μελών. Θα ήταν καλύτερο τα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαβάζουν το νομοθέτημα πριν να κατηγορούν οποιονδήποτε. Σας ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό τώρα. Α, συγγνώμη. έχει ζητηθεί μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Μάλιστα. Παρακαλώ, μπορείτε να θέσετε την ερώτησή σας. Έχετε 30 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ. αιτιολογούνται, υπάρχουν μάλλον αιτιολογήσει για τις τροπολογίες ε, του νομοθετήματος που αφορά τους νέους Πολωνούς ε, και την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Κύριε Γιάκη, πώς μπορούν τα παιδιά να αμυνθούν ενάντια στην ε, παιδοφιλία ή τις άσχημες συμπεριφορές, πώς ε, μπορούμε να αποφύγουμε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην πορνογραφία στο δίκτυο, εάν δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να αντισταθούν σε τέτοια πράγματα. 30 δευτερόλεπτα για την απάντηση. Μέσα από το δίκαιο μπορούν να αμυνθούν τα παιδιά αρκεί να δημιουργηθεί μια τέτοια νομοθεσία. Εάν δεν συμφωνείτε για την τιμωρία αυτού που προωθεί την ε, παιδοφιλία, ενώ θεωρείτε έγκλημα στα περισσότερα κράτη-μέλη, τότε έχετε πρόβλημα με την ερμηνεία αυτού του νομοθετήματος. Εγώ σας λέω την αλήθεια. Το δείχνουν αυτό και οι έρευνες για την παιδοφιλία. Να μην ε, ε, εκνευρίζεστε όταν ακούτε μία ενοχλητική αλήθεια. Δεν είναι το νομοθέτημα αυτό το, της κυβέρνησης είναι ένα νομοθέτημα των πολιτών και η πολωνική κυβέρνηση είπε ότι οποιοδήποτε νομοθέτημα δεν θα απορριφθεί πριν από την πρώτη ανάγνωση. Οπότε λέτε ηθελημένα λανθασμένα πράγματα. Πρόεδρος Διακόπτη, 30 δευτερόλεπτα έχετε για την απάντησή σας. Η κυρία Αντάμοβιτς, 30 δευτερόλεπτα επίσης. Δεν θέλω να σπαταλώ χρόνο για να διαβάζοντας και άλλες δικαιολογίες ε, για το νομοσχέδιο αυτό. Αλλά ο κύριος Γιάκη λέει πράγματα που είναι αναλυθή. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η παιδοφιλία, μάλλον ότι η, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν ε, είναι τίποτα άλλο παρά ιατρικές γνώσεις. Δεν πρόκειται για να ε, προσπάθει να πιστεί κάποιος να ξεκινήσει σεξουαλικές ε, σχέσεις γιατί η άγνοια των νέων οδηγεί σε σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα, καταθλίψεις και άλλα ψυχολογικά νοσήματα και προβλήματα. Άρα το ερώτημα που τίθεται για τους γονείς είναι προτιμούν να μάθουν τα παιδιά τους για την σεξουαλική ζωή από τους ε, συνομιλίκους τους, από το διαδίκτυο ε, ή μάλλον θα προτιμούσαν τα παιδιά τους να μάθουν για την σεξουαλικότητα από επαγγελματίες, από εκπαιδευτικούς και δασκάλους που είναι και εκπαιδευμένοι ζητήθηκε μπλε κάρτα για την κυρία ε, Ζελεύσκα. την δέχεστε? Απάντηση ναι. 30 δευτερόλεπτα για την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ρωτώ το εξής. Είδατε τα βασικά κείμενα αυτού που ονομάζουμε ε, εκπαίδευση ή διαπαιδαγώγηση για την ε, οικογενειακή ζωή και διαπιστώσατε ότι εκεί αντικατοπτρίζει το 21ο γονέας, Ο, ο γονέας, ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει το παιδί για τη ζωή και γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα ειδικό προφυλακτικό πρόβλημα, ε, πρόγραμμα προφύλαξης το οποίο παρέχεται δια νόμου και εκεί περιλαμβάνονται όλα τα σοβαρά ζητήματα. Ναι. Θα σας διαβάσω ε, μια αιτιολόγηση και θα σας πω τι ποινικοποιείται. Τα μαθήματα που προωθούν τη σεξουαλική δραστηριότητα ή που επενούν τη σεξουαλική δραστηριότητα οτιδήποτε περί αντισύλληψης, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ε, ε, νοσημάτων, ε, θέματα ορίμανσης κτλ. Εγώ είμαι μητέρα. Γνωρίζω και το πρόγραμμα αυτό και άλλα προγράμματα. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά η υπεύθυνη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και διαπαιδαγώγηση, αν, αν λείπει αυτή η διαπαιδαγώγηση, θα έχει φοβερά αποτελέσματα μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ηλεκτρονικό σύστημα. Αν θέλετε να υποβάλλετε ερώτημα μέσω ε, μπλε κάρτας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το ηλεκτρονικό σύστημα. Ε, ο κύριος Τσουχαντάρου για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι γιατρός και πάντοτε ήμουν υπέρ της εκπαίδευσης ε, υγείας. Είναι ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη των ασθενειών. Όταν μιλάμε για ε, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα των νέων που είναι μια μεγάλη ε, ε, μεγάλη επιδημία στην Ευρώπη, το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Όπως λέμε στη Ρουμανία, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει υγεία. Ε, αυτά, αυτό που είναι καλό για τα παιδιά μας δεν θα πρέπει να, ε, να, να το καθυστερούμε. Ας αφήσουμε την υποκρισία και ας λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες που καταδικάζουν το δικαίωμα στην υγεία και την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν μπορούν να περάσουν, δεν πρέπει να περάσουν. Ελπίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ε, χώρες θα αντιμετωπίσουν το θέμα διαφορετικά και άρα η ελευθερία στην πολυμορφία συνεπάγεται πάσης φύσεως παιδεία. Ευχαριστώ κυρία ε, Κάλτσμπρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο στην Πολωνία στήριξε ε, τις εργασίες για το νομοσχέδιο αυτό γιατί σε αυτό γίνεται λόγος για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία ότι δεν θα πρέπει ε, ουσιαστικά να γίνεται γιατί έτσι θα μειωθεί η παιδοεραστία υποτίθεται. Αυτό είναι όμως ένα σφάλμα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Το μόνο μπορεί να συμβεί να πάνε στη φυλακή εκπαιδευτική που θα κάνουν μαθήματα σεξουαλικής αγωγής. Αν δεν έχουν οι νέοι όμως αυτές τις γνώσεις ε, ε, από μόνοι τους ε, θα προστατευτούν πολύ χειρότερα από σεξουαλικές και πράξεις. πράξει. Είναι πολύ σημαντική η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για τα νεαρά παιδιά, για το πώ μπορούν να, είναι κύριοι και κύριε του σώματό του. Και σίγουρα χρειάζεται ισότητα, να μπορεί να ζουν όλη τη σεξουαλικότητά του. Δεν έχει ακόμη ψηφιστεί το νομοσχέδιο, αλλά νομίζω ότι είναι καιρό ε, αυτή την μισογενική πρόταση να την ε, προσπαθήσουμε να την ε, ακυρώσουμε. Γι' αυτό συζητούμε σήμερα να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρότυπα για την παιδεία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Κέμπα. Για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ουσιαστικά πρόκειται για νομοσχέδιο το οποίο υπογράφουν 265.000 άνθρωποι. Είναι ουσιαστικά μια πρωτοβουλία όχι κυβερνητική αλλά από την κοινότητα των πολιτών. Εσείς λοιπόν εδώ τι ήρθατε να κάνετε, να προωθήσετε την παιδεραστία γιατί εδώ ε, θέλουμε να ε, προωθήσουμε ένα νόμο κατά της παιδεραστίας. Αυτό είναι, ε, αυτός είναι ο λόγος αυτή, αυτού του νομοθετήματος. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η παιδεραστία Εσείς όμως τελικά αυτό βλέπω να θέλετε να υποστηρίξετε. Κατάρρεψη των ε, φραγμών για τα θύματα. Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Να, να μην μπορούν να προστατευτούν τα θύματα. Κύριε Πεντρού, δεν μπορείτε να αποπροσανατολίζετε το Κοινοβουλίο γιατί είναι ένα σοβαρό θεσμικό όργανο. Εδώ μιλάμε για απαγόρευση της παιδεραστίας, όχι για κάτι άλλο. Πολύ επιλεκτικά ε, τα λέτε για αυτό το νόμο. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε, να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας. Και η μονάδα, η βασική, είναι η οικογένεια. Εκεί, ε, στο πλαίσιο της οικογένειας, οι γονείς είναι αυτοί που σύμφωνα με το Πολωνικό Σύνταγμα θα πρέπει να, να, να τρέφουν τα παιδιά τους. Ευχαριστώ. Κύριος Μπίεντρουν έχει μια ερώτηση προς εσάς. Τη δέχεστε όχι. Και έχετε από την κυρία Ντάμοβιτς μπλε κάρτα. Νιέτ, δεν τη δέχομαι. Then we proceed. One minute, Mrs. Jones. Άρα προχωράμε, κυρία Jones, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πίτρο Κίνγκ, δεν είναι θέμα διδασκαλία, είναι θέμα ισότητα, αξιοπρέπεια και δικαιωμάτων των παιδιών που είναι θεμελιώδει αξίες τη Ευρωπαϊκή Ένωση και που περιλαμβάνονται στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ένα από τα βασικά δικαιώματα κάθε κοινωνία, είναι, υποχρεώσει κάθε κοινωνία είναι να διδάξει ε, τις θεμελιώδεις αρχές, την αρχή του σεβασμού, την ισότητα και τη αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι καθήκον μα ω γονεί και ω νομοθέτες, να μπορέσουν οι μελλοντικέ γενιές να μάθουν για τον εαυτό τους, το σώμα τους, το δικαίωμά τους και την αυτονομία τους. Η στέρηση του δικαιώματος της γνώσης και της σωματικής του αυτονομίας θα υπονομεύσει ουσιαστικά τα δικαιώματά τους. Η ποινικοποίηση της διδασκαλίας της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε παιδιά κάτω των 18 ετών αποτελεί σφάλμα γιατί ε, ε, οφείλεται σε επιθετικές πολιτικές απόψεις που δεν είναι δικές τους. τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΚΙ και των γυναικών κυρίως ε, παραβιάζονται όπως και οι δεσμεύσεις της Πολωνίας από τις ε, διεθνείς συμβάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταδικάσει το νομοσχέδιο και να βοηθήσει τις γυναίκες και τα άτομα ΛΟΑΔΚΙ από την στέρηση των δικαιωμάτων. Τους ευχαριστώ.

Πολωνία έχει γίνει πιο συντηρητική από το 2018. Οι νέοι στην Πολωνία εξαρτώνται από την, για την ενημέρωσή τους από το ίντερνετ. Μπορεί να συναντήσουν όχι μόνο το αυτά που προσπαθούν να βρουν για να αντισταθμίσουν την λυπή του σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αλλά και πολλά ύποπτα site μπορεί να συναντήσουν. Το νομοθέτημα αυτό προτείνει μέχρι και πέντε χρόνια φυλάκιση. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θεωρείται απειλή. Οι διφρονούντες λοιπόν δεν θέλουν να μείνουν σιωπηροί. Το στο ίντερνετ θέλει να δείξει στην, ε, ε, στην ε, νεολαία πως το, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν είναι έγκλημα. Μία, ένα περίφημο φω, φωτομοντέλο έγραψε ολόκληρο βιβλίο για να δείξει πως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν είναι παράνομη. Η, οι συντάκτε αυτού του νομοθετήματο γνωρίζουν ότι είναι η παιδοφιλία, η σεξουαλική θεπαιδαγώγηση είναι πλέον μέσα στα σύγχρονα, στη σύγχρονη διδακτέα ύλη ε, και θα πρέπει να βελτιωθεί, όχι να απαγορευτεί. Γιατί αυτή εμποδίζει τον κίνδυνο διάδοση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών, αλλά και ε, την παιδοφιλία επίσης. Δυστυχώ η Πολωνία οπισθοδρομεί και εμεί στο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να δείξουμε ε, και να στηρίξουμε όλους τους θαραλέους ανθρώπους που, στην Πολωνία οι οποίοι αντιστέκονται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρασνοντεύσκη θέλει να σας θέσει μια ερώτηση. Τη δέχεστε? Μαξοβά. Κυρία Μάξοβα, δέχεστε ε, μπλε κάρτα? Κυρία Μάξοβα, δέχεστε την μπλε κάρτα? Όχι. Προχωρούμε τότε. Ένα λεπτό η κυρία Βυσνιεύσκα. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά ένα νομοσχέδιο το οποίο προτείνεται στο Πολωνικό Κοινοβούλιο από μια ομάδα πολιτών δεν πρόκειται για νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει τέσσερις παραγράφους. Πρώτον, ε, ποινικοποιεί την παιδεραστία και επιβάλλει κυρώσεις. Δεν νομίζω να είναι κανείς κατά, εκτός από τον κύριο Μπιεντρών. Δεύτερον, δημοσίευση των σεξουαλικών επαφών με παιδιά. Παράγραφος 3. Δημοσίευση στα μέσα ενημέρωσης αυτών των πράξεων και τέλος προώθηση της των σεξουαλικών επαφών και σεξουαλικών ε, δραστηριοτήτων με άτομα με ανηλίκους ε, επισύρει ε, φυλάκιση. Άρα είναι ε, ψεύδος αυτή. Σας παρακαλώ, κάντε την ερώτησή σας και τηρήστε το χρόνο. Μα παραπλανάτε το σώμα. τα μέλη της ομάδας σας ψήφισαν υπέρ τα μέλη του κόμματό σας ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου. Κυβερνάτε εσείς στην Πολωνία, δεν κυβερνούν Αριανοί και εσείς έχετε την πλειοψηφία. Γιατί παραπλανάτε το σώμα. Κύριε Μπιετρώνη, θα το πω ξεκάθαρα ώστε να το αντιληφθείτε. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αποτελεί πρωτοβουλία πολιτών. Δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Έχετε άγνοια βασικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών γιατί ως εθνικός βουλευτής ε, δεν είστε εθνικό βουλευτή, είστε ευρω, ευρωβουλευτή. Είναι έσχο. Σα παρακαλώ, λέει ο πρόεδρο, μην προσβάλλετε τα μέλη. Η κυρία Ινσύρ για ένα λεπτό. Εγώ δεν είναι. Γνωρίζουμε που ζούμε. Ζούμε στο 2019 και μιλάμε για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Πολωνία. Μπορείτε να τα ξαναπείτε παρακαλώ. Ναι, έλεγα λοιπόν, αγαπητέ Περό, αγαπητέ Επίτροπε Κίνγκ, ζούμε στο 2019. Η Ευρώπη είναι Ευρώπη των περιφερειών. Έχουμε τον νόμο για την άμβλωση Και τώρα έχουμε ε, το νόμο που θέλει να απαγορεύσει σεξουαλική διαπαιδαγώση στην Πολωνία. Δεν θέλει λοιπόν πλέον να γίνεται ε, τέτοιο μάθημα στα σχολεία. Και είναι μια παράνομη δραστηριότητα που μπορεί να κολλαστεί και με φυλάκιση για τους εκπαιδευτικούς. Βλέπουμε λοιπόν πόσο ακραία συντηρητική είναι η στάση της ε, ε, πολωνικής κυβέρνησης και όποιος θεωρεί ότι αυτό έχει ως στόχο την καταπολέμηση παιδεραστίας ψεύδεται. Οι νέοι πρέπει να μάθουν το σώμα τους, να εξασφαλίσουν την ε, σωματική τους ακαιρεότητα και την ε, γενικότερη ακαιρεότητά τους. Γιατί αυτό μπορεί πράγματι να αποτρέψει ε, τη δεκτική μεταχείριση και την κακοποίηση, την κατάχρηση. Όλοι έχουν το δικαίωμα να ορίζουν το σώμα τους. Γι' αυτό χρειάζεται και σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, γιατί θα προωθεί στην ισότητα. Δεν θέλουμε λοιπόν να, ε, να κάνουμε βήματα προς τα πίσω, αντίθετα βήματα προς τα μπρος και θέλουμε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για όλους. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζαλεύσκα, η κυρία Ζαλεύσκα θέλει να σας θέσει μια ερώτηση. Δέχεστε. Όχι, ο κύριος Κρασνοντεύσκη θέλει να σας θέσει μια ερώτηση. Δέχεστε. Όχι. Και ο κύριος Γιάκη από ό,τι βλέπω. Δέχεστε. Και τρίτη φορά όχι θα πω. Τρίτωσε το όχι. Μάλιστα. Έτσι ολοκληρώνω το κατάλογο των ομιλητών και προχωρούμε στη δικασία Catch the Eye. Σόιντροβα. Děkuji za udělení slova. Kolegyně a kolegové, já nesouhlasím s tím, abychom dělali... Σας ευχαριστώ. Η ε, σεξουαλική δεπαιδαγώγηση στην Πολωνία θα πρέπει να ε, γίνει ευρωπαϊκό θέμα. Αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχεί και να συζητάμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η προστασία των παιδιών κατά των ε, των καταχρήσεων, η προστασία των παιδιών που εκτίθενται σε πιέσεις ε, σεξουαλικές μέσω του ίντερνετ ή της τηλεόρασης τα παιδιά δεν είναι κατάλληλα ενημερωμένα για τα σώμα τους. Δεν είναι αλήθεια αυτό γιατί στην βιολογία ή και σε παρόμοια μαθήματα ε, μαθαίνουν για το σώμα τους και πώς λειτουργεί. Άρα ε, εκπαιδεύονται στην βιολογία, στην οικογένειά τους και στην ηθική. Ε, εγώ φοβάμαι ότι γίνεται μια απόπειρα να ξεχωριστεί η σεξουαλική επαιδαγώγηση και να απομακρυνθεί από τις οικογένειες. Είμαι κατά τέτοιου είδους σεξουαλικής δαπαιδαγώγησης. Κατανοώ ότι ορισμένοι από εσάς ανησυχείτε για άλλες πηγές ενημέρωσης των παιδιών όπως η πορνογραφία και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό ε, είναι θέμα του κάθε κράτους μέλους να προστατέψει τα παιδιά του. Ο κύριος Κρασνοντεύσκη. Άκουσα τη συζήτηση μέχρι τώρα, αλλά ήταν πολύ παράξενη. Μιλάμε για ένα νομοθέτημα που προήλθε από τους πολίτες και έφτασε στο Πολωνικό Κοινοβούλιο. Οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν το γνωρίζουν, δεν έχει ακόμα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες εκτός από τα πολωνικά και πολλοί εξ πήραν το, λόγο, πήραν το λόγο και μίλησαν για το δικαίωμα. Δεν ήξεραν όμως καθόλου για τι πράγμα μιλούσαν. Είναι μια αυτόματη αντίδραση που υπάρχει όταν ε, μπορεί κανείς να αρχίσει να επικρίνει την πολωνική κυβέρνηση και βασίζεστε σε λανθασμένες πληροφορίες. Οπότε παρακαλώ για το μέλλον κάνω μια έκκληση. Αν θέλουμε να συζητήσουμε κάτι, ε, διαβάστε το πρώτα, δείτε τα έγγραφα και μετά μπορούμε να συζητήσουμε για τα πάντα αλλά με σοβαρότητα. Και παρακαλώ να μην ε, μιλάτε θυμαγωγικά. Ένα λεπτό, κύριο Σόκορ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής. Καθορίζει τις ζωές και τις αξίες μας. Όπως και το πολιτικό μέλλον της Υπήρου μας. Θα πρέπει να πω ότι η παιδεία έχει προχωρήσει, έχει εμπλακεί όλο και περισσότερο με την πολιτική και αυτό δεν είναι νέο φαινόμενο, ε, ιστορικά συμβαίνει από παλιά. Όμως δεν είναι κάτι καλό, γιατί οδηγεί σε ολοκληρωτικές περιόδους ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Η παιδεία πρέπει να στηρίζεται σε γεγονότα και στην επιστήμη. Κάνω έκκληση. Μην συζητάτε για την παιδεία ε, με βάση την ιδεολογία. Τα στοιχεία, τα γεγονότα πρέπει να γίνουν γνωστά και μετά να συζητάμε με βάση αυτά. Το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να μελετηθεί σωστά ώστε να μπορούμε να αποφασίσουμε. Πρέπει να... One minute, Mr. Ευχαριστώ. Είμαι πεπισμένος ο κύριος Πόλτσακ ότι η παιδεία είναι η λύση, ιδίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με το σκοταδισμό και την επικίνδυνη συμπεριφορά τη σεξουαλικά μεταδόμενες νόσους, βιασμό, ε, εγκυμοσύνες ανεπιθύμητες, ε, αμβλώσεις κτλ. Όλα αυτά είναι επιπτώσεις της έλλειψης πληροφόρησης κύριος Μπιντρούν ε, μπόρεσε να εκφραστεί ελεύθερα ουσιαστικά. αλλά η συνάδελφο ε, που το επιτέθηκε δεν το επέτρεψε ουσιαστικά να έχουν μια συζήτηση. Αλλά η συζήτηση νομίζω είναι καλή. Πρέπει να καταδικάζουμε τα κακό σκήμα στον θεσία και ελπίζω να μας ενημερώσει η κυβέρνηση ότι δεν θα πέρασε αυτό το νομοσχέδιο. Πρόεδρος, εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει στην πρώτη σύνοδο Ολομέλειας Νοεμβρίου. Επόμενο σημείο στη μέση διάταξη είναι δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις καταιγίδε στην Ευρώπη, ιδίω ε, τις έντονες βροχοπτώσεις στην Ισπανία και τον τυφώνα στις Αζόρες Πορτογαλίας. I Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο King. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η Επιτροπή γνωρίζει προφανώς πολύ καλά τις επιπτώσεις των καταιγίδων και των πλημμύρων σε διάφορες περιοχές της νότιας και ανατολικής Ισπανίας, όπως και του τυφώνα Λορέντσο στις Αζόρες. Πραγματικά εκφράζουμε την λύπη μας για όλους ε, όσοι έχασαν τη ζωή τους και τα υπάρχοντά τους. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή σε συνεργασία με τις Ισπανικές και Πορτογαλικές αρχές επιδιώκει να βρει τρόπους να ε, αντιμετωπιστούν οι ζημιές. Μιλάμε για περιοχές που έχουν πληγεί από ε, ε, σοβαρές φυσικές καταστροφές, οι οποίες δικαιούνται οικονομική ενίσχυση. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν ήδη έχουν συναντηθεί με τις αρχές της περιοχής της Βαλένσια και των Αζωρών για να εξηγήσουν τις ε, προϋποθέσεις και τις διαδικασίες βάσει των οποίων θα ενεργοποιηθεί το Ταμείο ε, αλληλεγγύης. σε μια πρόσφατη επιστολή στην Κομισιόν, οι Ισπανικές Αρχές ε, ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να ζητήσουν τη βοήθεια του Ταμείου Αλληλεγγύης όταν ε, ολοκληρωθεί η εκτίμηση των ζημιών. Αν ε, η αίτηση υποβληθεί εντός της προθεσμίας και οι μελέτες της Κομισιόν διαπιστώσουν ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις ανεργοποίησης του Ταμείου, τότε θα προτείνει ε, ε, η Κομισιόν ένα ποσό βοήθειας το οποίο θα εγκριθεί από εσάς και από το Συμβούλιο. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρόκειται για περιφερειακές καταστροφές όπως ταξινομούνται όπου η βοήθεια μπορεί να φτάσει μέχρι το 2,5% του συνόλου των άμεσων ζημιών. Επιπλέον το ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία μπορούν και αυτά να παρέμβουν με βοήθεια για τις ε, ε, εργασίες αποκατάστασης. Κάποιες από τις ζημιές, αν, αν κάποιες από τις έχουν πλήξει και τον αγροτικό τομέα, το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει ενδεχομένως για ζημιές από φυσικές καταστροφές και να βοηθήσει με προληπτικές δράσεις. Οπότε και αυτό μπορεί να στηρίξει τους ε, αγρότες για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Για την αποζημίωση των ζημιών στους πρωτογενείς παραγωγούς από ε, βροχοπτώσεις και πλημμύρες, τα κράτη-μέλη μπορούν, όπως γνωρίζετε είμαι σίγουρος, να μελετήσουν την χορήγηση κρατική, κρατικών ενισχύσεων. Υπάρχουν όλοι οι τρόποι που σας ανέφερα. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε όλους όσοι πλήγησαν από αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Συνεχίζουν οι δηλώσει εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Δύο λεπτά η κυρία Μπενχουμέα εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να πω ότι ήδη ενέκρινε το πρωί ε, τη συμπερίληψη ε, στο, ε, στην σχεδιάταξη αυτό το, του θέματος, κάτι πολύ θετικό. Η Ισπανική κυβέρνηση υπολογίζει, λέει, ακόμη τις ε, ζημίες για τη Μούρθια, τη Βαλένθια, την Αλμερία μετά αυτές ε, τις καταρακτώδεις βροχές ε, που έπληξαν την Ισπανία από τις 12 έως 15 Σεπτέμβρη. Πρόκειται για ζημίες ε, που τώρα έχουν υπολογιστεί και θέλω να καταγγείλω την αδράνεια της κυβέρνησης του Πέντρο Σάντσεθ που ασκούσε καθήκοντα τότε για να δρομολογηθεί και να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης ως δεμότερο δυνατόν διότι ιδίω η Μούρθια καλύπτει όλες τις προποθέσει για να είναι δικαιούχος αυτού του Ταμείου. Δυστυχώς όμως υπήρξαν έξι νεκροί. Υπήρξαν ζημίες που η κυβέρνηση, η περιφερειακή κυβέρνηση της Μούρθια τις υπολογίζει σε 560 ε, εκατομμύρια και ε, πολύ ψηλέ επίσης και στην Βαλέθη και στην Ανταλουσία πάνω από 100 εκατομμύρια και εκεί. Ε, και υπάρχουν πολίτε οι οποίοι περιμένουν από την Ευρώπη να αντιδράσει. Μια βασικέ ευρωπαϊκέ αξίε είναι η αλληλεγγύη. Και το Ταμείο Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη γι' αυτό το λόγο υπάρχει. Για να αντιδρά και να αποκρίνεται στην ανάγκη των πολιτών που βιώνουν ε, δραματικές συνθήκες που τους ξεπερνούν, σαν αυτές που είδαμε στην Ισπανία. Από εδώ λοιπόν από το Ευρωκοινοβούλιο ζητώ από το Συμβούλιο και από τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο στο, το Ταμείο Αλληλεγγύης να δομολογηθεί και το λέω γιατί μπορεί να επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό στις Βαλεαρίδες, στη Βαλένθια ή στην Καταλωνία τις μέρες αυτές που μιλάμε. Να επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα καταρακτώδεις βροχές, πλημμύρες. Δεν πρέπει λοιπόν να καθυστερούμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε εβδομάδες για να αντιμετωπίσουμε φυσικές καταστροφές σαν αυτές που είδαμε στην Ισπανία ή σαν αυτές που υπέσαν στις Αζόρες, Πορτογάλοι γειτονές μας. Θα πρέπει να είναι αλληλέγγυα Ευρώπη, να μπορεί να αντιδρά γρήγορα και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των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 Eh, Έλεγα ότι χαίρομαι και εγώ που, που προσθέθηκε το θέμα αυτό στην ημερήσια ε, διάταξη, αλλά ήταν ατυχή η παρέμβασή τη προλαλή σα, γιατί οι βροχοπτώσει και τεράστιες καταστροφές ε, δεν θα πρέπει για κομματικού ε, λόγου να χρησιμοποιούν αυτή τη συζήτηση, επειδή έχουμε εκλογέ τον Νοέμβριο. Όλε οι κυβερνήσει κάνουν τη δουλειά του σε αυτονομίες, σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε Ομοσπονδιακό, που ήδη έγινε η αρχική εκτίμηση των ζημιών και θα πρέπει να περιμένουμε να υπολογιστούν όλε οι ζημιές για να γίνει μια σωστή εκτίμηση. Και θέλω να πω ότι η κλιματική αλλαγή ουσιαστικά είναι αυτή που ευθύνεται για το φαινόμενο αυτό ε, των πολύ ε, έντονων ροχοπτώσεων, Εγώ τα φρία λέγεται στα Ισπανικά και πλήττει τις Βαλεαρίδες, τη Μούρθια, την Αλμερία και τη δική μου την περιφέρεια ε, στη Βαλένθια, αλλά και ε, στην υπηρετική χώρα Ναβάρα, Ριόχα, Μαδρίτη. Όλα αυτά είναι συνέπεια μιας κλιματικής αλλαγής που όλοι έχουμε την ευθύνη να καταπολεμήσουμε. Αυτό που ζητάμε τώρα λοιπόν είναι ε, να δράσουμε όλοι μαζί, ώστε όλοι οι πόροι, όλα τα μέσα και βέβαια και οι ευρωπαϊκοί πόροι και μέσα να τεθούν στην υπηρεσία των πολιτών. Πολίτες θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι εκεί η Ευρώπη όταν τη χρειάζονται. Πρέπει όμως ε, εκτός της αποζημίωσής τους να επενδύσουμε και εδώ και η ανάγκη των ταμείων των ευρωπαϊκών να επενδύσουμε για να μην ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται με αρκετά μεγάλη συχνότητα. Στη Μεσόγειο έχουμε ξηρασίες έχουμε απερίμωση ε, και ταυτόχρονα τέτοιες καταρακτός βροχές ε, που ουσιαστικά δεν βοηθεί ε, το νερό, η ποσότητα όπως πέφτει να συγκεντρωθεί για να αντιμετωπίσει ακριβώς τη ξηρασία και τις επιπτώσεις της. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε ώστε να μην ξανά τέτοια φαινόμενα και όταν έχουμε συναγερμό να ε, ε, αναλαμβάνεται έγκαιρα δράση ώστε στις περιοχές αυτές να μην ξανασυμβούν αυτές οι καταστροφές. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά, κύριε Σολίθ Πέρεθ από το Renew. Νοτιοανατολική Ισπανία ε, ζήσε ε, τα τελευταία 140 χρόνια τρομερή φαινόμενα, 150 χιλιόμετρα ε, ρηπές του αέρα, βροχές, καταστροφικές οι επιπτώσεις, 6 νεκροί, πάνω από 4.000 άνθρωποι κενώθηκαν, έμειναν χωρίς σπίτια, χωρίς ρεύμα και επίσης υποδομές σε πάνω από 25 δήμους υπέστησαν ζημιές. Ε, όμως εδώ είναι η πύλη για την Ευρώπη αυτή η περιοχή. Πάνω από 3.000 εκτάρια γης ε, υπέστησαν καταστροφές. 500 εκατομμύρια πόλη στη Γεωργία. Πάρα πολύ μεγάλη ε, η ε, ζημιά και για το οικοσύστημα που είναι δύσκολο τώρα να επαναλάβουμε, μάλλον να γυρίσουμε στην πρώτερα κατάσταση. Σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές λοιπόν οι επιπτώσεις και οι καταστροφές. Εμεί αυτό που ζητάμε πέρα σε αυτήν την κατάσταση είναι να δομολογηθεί, να κινητοποιηθεί το Ταμείο για να αντιμετωπιστούν ε, τα μεγάλα, οι μεγάλες καταστροφές ε, των ε, πλημμυρών, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν αλείς γεωργοί, να μπορέσουν να οικοδομήσουν τη ζωή τους και το μέλλον τους. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι μία ακόμα φυσική καταστροφή σαν αυτές που θα πλήξουν τους τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Και όλα αυτά καταδεικνύουν πόσο αναγκαίο είναι όλα τα κράτη-μέλη μαζί να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Μπορεί τώρα να έπληξε το φαινόμενο την Πορτογαλία και την Ισπανία. Αύριο θα πλήξει άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Δυστυχώ δεν θα εξαφανιστεί αυτό το πρόβλημα. Στην Ισπανία σήμερα είχαμε συναγερμό για μια νέα καταιγίδα που πλησιάζει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκοί μηχανισμοί όπω το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελληνική Ένωση που θα ανταποκρίνεται σε αυτά τα προβλήματα. Αλλά χρειάζεται κάτι ακόμα, να γίνει επιστημονική έρευνα για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, για τον περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν αυτά τα φαινόμενα στην οικονομία, στο περιβάλλον και βέβαια πιο πολύ στην ανθρώπινη ζωή. Ευχαριστώ. Thank you. Two minutes, Mr. Δύο λεπτά ο κύριο Ντρεώστο, εξ ονόματο του ID. Ευχαριστώ, Πρόεδρε εκφράζουμε πάνω απ' όλα τη δική μας ε, ε, ε, συμπάθεια στις οικογένειες των θυμάτων και στους πληθυσμούς που επλήγησαν από αυτή τη τραγωδία, δηλαδή της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αλλά και άλλων περιοχών που επλήγησαν στην, στην Ήπειρό μας. Μόλις πριν από ένα χρόνο η καταιγίδα Βάια έκανε, προκάλεσε ζημιά στην Ιταλία για άνω των 6 δις ε, ε, ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Λεγγύης προσέφερε 250 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε τις κλιματικές αλλαγές που προκαλούν διαρκώς πιο έντονα καιρικά φαινόμενα και δεν μπορούμε επίσης να πούμε πως αυτό το, αυτή η κλιματική αλλαγή καθορίζεται από την ανθρώπινη ε, ανάπτυξη και από, άρα από τη ρήπαση οι δεσμεύσει που έχει αναλάβει το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πράσινο σύμφωνο, το Green Deal, θα πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα για να έχουμε τα, γρήγορα και τα αποτελέσματα. Όμω τα πρώτα αναμενόμενα αποτελέσματα που μπορεί να επηρεάσουν για τι κλιματικέ αλλαγέ θα, θα πάρουν δεκαετίε. Εν τω μεταξύ, τα ακραία φαινόμενα θα συνεχιστούν και ίσω να γίνουν και πιο έντονα από τα σημερινά και ε, θα επιδεινώσει την κατάσταση ο υψηλό υδρογεωλογικό ε, κίνδυνο ε, η τσιμεντοποίηση. Μετά από την καταιγίδα σκεφτόμαστε τις ζημιές αλλά πρέπει να έχουμε και τους απαραίτητους πόρους. Τα κράτη μαζί με την υποστήριξη της Ένωσης θα πρέπει να αναπτύξουν ε, ε, project με ε, μακρόπνοα ώστε να μπορέσουν ε, να καταπολεμήσουν τις καταχρήσεις που μεταφράζονται πολλές φορές όπως και σε αυτή την περίπτωση σε τραγωδίες. Ε, προστασία υδρογεολογική, ώστε να προστατευτούν εκείνοι που τις επόμενες ε, εστιώσεις στις επόμενες δεκαετίες να μην έχουμε τόσο πολλά έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, η κυρία Νουέβα Ρουίθ, εξ ονόματος της GUE Μιλάμε για συνέπειες. Είναι κοινικό να ακούμε το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ηγέτης πριν από λίγο καιρό γελιοποιούσε τη χώρα μας, ε, αρνούμενος στις κλιματικές αλλαγές. Το κόμμα το οποίο συστηματικά συνεργάστηκε με κατασκευαστικές εταιρείες που έχτιζαν σε ζώνες που, που, που, που κινδύνευαν από πλημμύρες, ε, όπου ε, μπόρεσαν να κερδίσουν μόνο λίγοι ενάντια στην ασφάλεια των πολιτών και αυτό με μεγάλη αδιαφάνεια όσον αφορά την υδρογεωλογική κατάσταση της χώρας. Θα πρέπει αυτό να αλλάξει. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2007 ήδη αναγνωρίζει τις κλιματικές αλλαγές. Ε, πέρα από αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα αλλά πρέπει, δεν πρέπει να πληρώνουν πάντα οι ίδιοι και γι' αυτό είναι σημαντικό το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργήθηκε για να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις ε, σοβαρών φυσικών καταστροφών να προσφέρει αλληλεγγύη σε περιφέρειες στην Ισπανία όπως η Ναβάρα, οι Βαλεαρίδες ή η Βαλένσια. Ε, χρειαζόμαστε μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη μετάβαση, σε ένα νέο πρότυπο και να σταματήσει η κερδοσκοπία με βασικούς πόρους όπως το νερό. Για ένα μισή λεπτό, κύριο Φερνάντε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 2 Οκτωβρίου στην, υπε, στην υπερπεριφερειακή περιοχή ε, ε, ε, των Αζωρών ε, μια μεγάλη καταιγίδα προκάλεσε 3,5 δίσεις ζημιές. Έχουμε πολύ σημαντικό νησιωτικό σύνολο εκεί. Το λιμάνι των Αζωρών καταστράφηκε και οι ζημιές είναι ε, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Να λάβετε υπόψη ότι έχω το, ε, αφού πέρασαν κάποιες μέρες, αφού ενέκρινε ε, το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο, το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο ε, συγκεκριμένα κονδύλια για να καλυφθούν αυτές οι ζημιές. Είναι απαραίτητο όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι γρήγορη. Η αλληλεγγύη είναι ουσιαστική στην πράξη και για την κινητοποίηση του Ταμείου Λιλικής ή για την ε, εκ νέου προγραμματισμό των Ταμείων ε, για το 2020 ε, είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενεργήσει σύμφωνα με τους νόμους και γρήγορα. Πορτογαλία ε, περιμένει χρήματα από το ορίζοντα 2020 τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο που υποφέρει από πολύ σημαντικές ζημιές και δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένη περιοχή που χρειάζεται παραπάνω στήριξη σε μια τέτοια έκτακτη κατάσταση. Σας ευχαριστώ. 1,5 λεπτό η κυρία Καρβαλιάης. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από δύο εβδομάδες ε, μίλησα ε, σε αυτή την ε, αίθουσα για τον τυφώνα Λορένσο που πέρασε από την Σαζόρες. Ήδη τότε είχα, είχαμε δει τις ζημιές και ε, γίνονταν υπολογισμοί και υπολογίζαμε ότι θα ήταν πολύ, πολλά τα χρήματα. Πρόκειται για εφτά εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια περιοχή όμως ιδιαίτερα απομακρυσμένη και οι ζημιές αυτές έχουν πλήξει όλη την κοινωνία. Ε, κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, υπηρεσίες, ε, λιμενικές υποδομές, ε, σκάφη, αλλά και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ε, γίνονται ε, προσπάθειες σε περιφερειακό επίπεδο και σε κρατικό επίπεδο και έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για να ε, υποδεχτούμε τον κόσμο που έχει αναγκαστεί να φύγει από τα σπίτια του. Εδώ όμως ζητώ και πάλι τη στήριξη για να εγγυηθούμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τις Αζόρες. Μια στήριξη που θα πρέπει να είναι πραγματική, γρήγορη και αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Αντρουέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για τις βροχές και τους τυφώνες ε, είναι ένα θέμα που μάλλον ε, ε, έχει σχέση με ανακοινώσεις παρά με προβλητική. Πραγματικά οι λαοί που αντιμετωπίζουν τους κινδύνους δεν πρέπει να περιμένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς για να σωθούν. Το θέμα είναι γιατί το ΕΛΚ θέλησε να συμπεριλάβει το θέμα των φυσικών καταστροφών στην ημερήσια διάταξη. Γιατί ενώ σε δύο μέρες θα ψηφίσει για να πάνε να μην πάνε τα ε, ε, χρήματα στα ε, για, τη, για την ελληνική στα θύματα των φυσικών καταστροφών μετά από οι οδηγίες επιτροπής. Αυτό είναι α, ανήθικο. Οπότε πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση γιατί σε 48 ώρες όταν ψηφίσουμε για τη σωτηρία των θυμάτων των φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη δεν θα βρισκόσαστε εδώ. Πρέπει η ομάδα Ιδαντιτέ και Δημοκρατία να βρίσκεται εδώ για να βοηθήσει τη διάσωση αυτών των ανθρώπων. One minute, Mr. Ferreira. Ένα λεπτό, κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, ο τυφώνας Λορέντζο προκάλεσε σημαντική καταστροφή στις Αζόρες. Καταστράφηκαν σπίτια, Άνθρωποι οι οποίοι έμειναν χωρί σπίτια, καταστράφηκαν υποδομέ, τηλεπικοινωνίε, ενέργεια και άλλε υποδομέ. Καταστράφηκε το εμπορικό λιμάνι που είναι ουσιαστικό για τι επενδύσει αλλά και για την ε, ε τροφοδοσία των νησιών ε, ε, των Αζωρών και του Κόρβου πάρα πολύ ε, μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αναγκάστηκε να φύγει από τα σπίτια του. Οι υποδομές έχουν φύγει. Θα χρειαστεί κινητοποίηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η στήριξη θα πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο σύντομα. Πέρα από αυτό όμω είναι τώρα καιρό για να ξεκινήσουμε ένα προβληματισμό για την ε, καταλληλότητα των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μα ώστε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου καταστάσει. Θεωρούμε πω είναι απαραίτητο και υπάρχει και δυνατότητα για προσαρμογή εφαρμογή πέρα από το Ταμείο Αλληλεγγύης στο, μπορεί αυτό να τελειοποιηθεί, βελτιώθηκε στο παρελθόν και μπορεί ακόμα να βελτιωθεί. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα διαρθρωτικά ταμεία. Λείπουν χρήματα για να καλύψουμε μια τρύπα, παίρνουμε από αλλού. Ενώ θα πρέπει να μιλήσουμε για εξαιρετικέ καταστάσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις και γι' αυτό στις περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε και έκτακτα κονδύλια. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό ο Νόβακοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ευθύ εξ αρχή να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και τη συμπάθειά μου στις οικογένειες που έχασαν ε, τους δικούς τους της πλημμύρας Ισπανίας. Μιλάμε για ένα μέσο που δεν είναι ταχείας αντίδρασης, το γνωρίζω. Όμως πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης του χρόνου απόκριση. Γνωρίζω ότι έχουν ε, γίνει επενδύσεις ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας του Ταμείου και ο χρόνος ε, που απαιτείται για να φτάσει η βοήθεια στις περιοχές που έχουν πληγεί. Όμως πιστεύω ότι η αλληλεγγύη είναι αλληλεγγύη την ώρα που πρέπει. Η βοήθεια είναι βοήθεια όταν παρέχεται την ώρα που πρέπει. Νομίζω λοιπόν ότι Ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά και πιστεύω ότι και αυτή αλλά και η επόμενη επιτροπή και ο νυν και ο επόμενος επίτροπος μπορούν πολλά να κάνουν. Πιστεύω ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να μελετηθεί έτσι ώστε να βοηθά τις περιπτώσεις αυτές με τρόπο ισορροπημένο. Γιατί η, ε, ατελείωτος, ο ατελείωτος αναπρογραμματισμός των επιχειρησιακών προγραμμάτων μπορεί να υπονομεύσει τους στρατηγικούς στόχους. Άρα το Ταμείο Συνοχής μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο αυτό μπορεί να προσφέρει στην περαιτέρω βελτίωση του Ταμείου για να βοηθηθούν οι πολίτες. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, η κυρία Σέρντας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει σημαντικά, μεγάλα σημάδια αλληλεγγύης, αλλά υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι οι άνθρωποι. Στη διάρκεια του περάσματος του τυφών Λορένζο από τις Αζόρες σε μια ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένη περιοχή, Ε, πολλοί άνθρωποι εξέφρασαν την συμπαράστασή του. Κατέστρεψαν, κατέστρεψε ο τυφώνας ε, τελείως το λιμάνι, ε, το οποίο είναι αυτό που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των νησιών. Εν γέννη, οι ζημιές ανέρχονται σε 330 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα μια φορά θα ήθελα να ζητήσω η Κομισιόν να δείξει την αλληλεγγύη της. Ε, θα δείξουμε ότι κυβερνόμαστε από ανθρώπους που προσέχουν τις ανάγκες ε, του κόσμου. Γρήγορη κινητοποίηση λοιπόν του Ταμείου Αλληλεγγύης και προγραμματισμός κονδυλίων για να στηριχθεί ο πληθυσμός των αζωρών και να αντιμετωπίσει τις τεράστιες ζημιές. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό κύριο Σαμάρο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όλοι μας μιλάμε για αλληλεγγύη σε αυτή την περίπτωση με την Ισπανία και με την ε, αυτόνομη περιφέρεια των Αζωρών, την ε, ε, απομακρυσμένη αυτή η περιοχή. Η αλληλεγγύη είναι ιδιαίτερα προσφυλή λέξη σε όλε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Πριν από λίγο είδαμε τον κύριο Πίτροπο που μα απαρίθμησε ένα σύνολο προοπτικών με βάση τις οποίες είναι δυνατόν να θετεθεί σε εφαρμογή, στην πράξη αυτή η αλληλεγγύη. Πιστεύω πραγματικά πω όπω ήδη ανέφεραν η Ιζαμπέλ και ο Ζεμανουέλ Φερνάντε και άλλοι ότι αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο ένας ε, κατάλογος υποθέσεων είναι το να ε, μεταφέρουμε αυτές τις υποθέσεις σε πράξη. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ε, προσαρμογές, αλλά οι πληθυσμοί, οι εταιρείε, οι άνθρωποι που αναφέραμε, άνθρωποι που δυστυχώς χάθηκαν, οικογένειες ε, που χτυπήθηκαν, αλλά και οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να αφήσουν τα υπαρχοντά τους, τη ζωή τους, την οικονομική τους ζωή που καταστράφηκε. Εάν υπάρχει λοιπόν μία στιγμή όπου αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης που τότε που δημιουργήθηκε ε, καλώς πέρα από τους υπόλοιπους μηχανισμούς που θα πρέπει να, να ενεργήσουν επί τόπου, θα πρέπει να το κάνουν αυτό έγκαιρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας είπε πως αυτό ε, ποτέ δεν πρόκειται να ε, ξεχαστεί και γι' αυτό θέλουμε να μας βοηθήσει και η Επιτροπή. Για ένα λεπτό. Η κυρία Λόπεθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να πω στην κυρία από το ΕΛΚΑ ε, να μην καταπιάνετε με πράγματα που, ε, με τα οποία δεν παίζει κανείς. Ε, δηλαδή με αυτούς που έχασαν ανθρώπους στις πλημμύρες ή με τον πόνο των εμπόρων που έπρεπε να καθαρίσουν τη λάσπη από τις εγκαταστάσεις και δεν ξέρουν πότε θα ανοίξουν. Ε, δεν είναι μόνο οι Βαλεαρίδες, η Καστίγια, η Λαμάντσα, η Βαλένθια και άλλες. Είναι η Ναβάρα με 600.000 κατοίκους που τον Ιούλιο είδαμε ε, στο μέσο, ιδίως στα Αρθάγια, και σε 22 χωριά ε, να χάνεται η ζωή ενός ανθρώπου, ε, να κλείνουν ε, πολλά σπίτια και πολλά καταστήματα που ακόμα δεν είναι κατοικήσιμα. Και μιλάμε και για μία κάθετη αλλαγή. Έχουμε την κλιματική αλλαγή και την πολιτική του νέου μέλλοντος από την Ένωση. Και κάτι άλλο. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Φυσικά ήταν εκεί η κυβέρνηση, εκεί ήταν και δημοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, έχει και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει απαντήσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό το Ταμείο Αλληλεγγύη να τροποποιηθεί, να επικαιροποιηθεί και να δημιουργηθούν νέοι μηχανισμοί από την Ένωση για να ανταποκρίνεται και να βοηθάει σε τέτοιε περιπτώσει πολίτε. Ένα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κυρία Πιθάρο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο τυφώνα Λορένς όταν έφτασε στις Αζόρες προκάλεσε τεράστιες ηλικές ζημιές, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι δυστυχώς υπήρξαν μάλλον ότι ευτυχώ δεν υπήρχαν ε, θύματα και αυτό είναι προ τιμήν των ε, δυνάμεων ε, των Αζωρών και του λαού των Αζωρών. Οι ζημιές ήταν τεράστιες. Το λιμάνι των Αζωρών καταστράφηκε εντελώς και είναι το λιμάνι το οποίο απαιτεί άμεση απάντηση γιατί αυτό τροφοδετεί τα νησιά το Φλόρες και του Κόρβο και από τις 3 Οκτωβρίου κάναμε έκκληση από πλευράς των σοσιαλιστών και 20 μέρες αργότερα δεν υπήρξε απάντηση λόγω εσωτερικών, εσωτερικής διαμάχης. Θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι για να μπορέσουμε να βρούμε απαντήσεις στα προβλήματα των ανθρώπων αυτών μέσα από το Ταμείο Αλληλεγγύης, αλλά κύριε Επίτροπε δεν φτάνει το 2,5% στήριξης για 430 εκατομμύρια ζημιές. Χρειάζονται πολύ περισσότερη ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για τους ε, ανθρώπους των Αζωρών. Και εμείς θα είμαστε εδώ για να θυμίζουμε ότι πρέπει να δοθεί μια απάντηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ όλους. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ομιλητών και φτάνουμε στη διαδικασία Catch the κυρία Σόιτρουμπα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είμαι ούτε Ισπανίδα ούτε Πορτογαλίδα. Ζήτησα το λόγο επειδή γνωρίζω τις επιπτώσεις της ε, κλιματικής αλλαγής, των ε, ακραίων ξηρασιών και πλημμυρών που αντιμετωπίζουμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις υπήρους. Είναι θέμα όλων των πολιτικών ομάδων. Δεν υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα που να να οικειοποιηθεί το θέμα. Το Ταμείο Ελληνικής θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό, ταχύτερο. Αυτό θα είναι δουλειά της νέας επιτροπής που θα πρέπει να λάβει μέτρα όπως ακούσαμε και από τον συνάδελφο προηγουμένως. Είναι όμως ε, καλύτερο πάντοτε να ε, ε, ε, ασχολούμαστε με την πρόληψη. Είναι πιο φθηνό και πιο αποτελεσματικό. Συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγέτη στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να αναγκάσει τους άλλους παγκόσμιους παίκτες να, πάρουν μέτρα, να φυτέψουν δέντρα και να φροντίσουν να ελαφρυνθούν τα φαινόμενα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσούταρο. Ε, ε, ε, κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνω ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γυλεγγύης είναι μια, μικρή, ένας μικρός επίδεσμος για μια βαριά πληγή. Θα πρέπει να γίνει αυτό που οφείλει να είναι πραγματική θεραπεία, επίγουσα θεραπεία για όσους το έχουν ανάγκη. Γιατί πραγματικά φτάνουν αυτές οι καταστροφές και δεν μπορούμε να ζούμε προστατευμένοι πάντα. Πρέπει όμως να, προλάβουμε. Σας είπα ότι η αποψίλωση των δασών στην Ευρώπη είναι πραγματικό δράμα. Στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο ο νόμος του Αντάρου εμποδίζει την αποψήλωση και την εκμετάλλευση ε, των ε, δασών. Όμως εδώ μιλάμε για ανθρώπους. Οι μηχανισμοί της πολιτικής προστασίας πρέπει να λειτουργούν σε συνδυασμό και τέτοιες μεγάλων ατυχημάτων ή φαινομένων. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους όταν και όπου έχουν ανάγκη και θα πρέπει η ελληνική ως ταμείο να λειτουργήσει πολύ καλά. Τρίτον, πρέπει να σκεφτούμε ότι καταλήγουμε σε καταστάσεις δύσκολες επειδή δεν έχει υπάρξει πρόληψη. Αν οι αγροτικές επιδοτήσεις ήταν ίδιες και για τους Ρουμάνους αγρότες ήταν καλύτερα. Ευχαριστώ closed. Ε, λίγη συζήτηση. The next item on the agenda is... Το επόμενο θέμα της ημερήσια διάταξη είναι οι ομιλία του ενό λεπτού ε, σύμφωνα με τον κανόνα 172. Mr. Ο κύριος μετά την, ε, στη Ρουμανία έγινε ε, πέρσι με επιτυχία η πρόταση μομφής και κατά πάσα πιθανότητα η κυβέρνηση συνασπισμού θα ε, αντικατασταθεί από μια συντηρική κυβέρνηση. Το έργο της νέας κυβέρνησης με τις επόμενες εκλογές θα είναι να εφαρμόσει μια πολιτική δημοσιονομική λιτότητα, να κάνει μια καλύτερη χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και να προετοιμάσει εκλογές, πράγμα σημαντικό σημαντικό εν ώψη του ε, προπολογισμού τη επόμενη χρονιά και βέβαια πρέπει να γίνουν διορθώσει. Όσον αφορά τους, σύμφωνα με του υπολογισμού ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, το 2017-2020 η κυβέρνηση τη Ρουμανία πήρε περισσότερα δάνεια από ό,τι κατά την περίοδο τη οικονομική κρίση. Το κόμμα που εκφράζει τα συμφέροντα τη ουγγρική μειονότητα θα είναι εταίρο τη επόμενη κυβέρνηση και θα συνεργαστεί ε, για να επικεντρωθεί στην υγιεινή ζωή, την παιδεία, την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην πλειοψηφία και την ουγγρική μειοψηφία. Πρέπει να ξεκινήσει διάλογος για ενδοεθνωτικές σχέσεις. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριος Λουέν. Ο Εθνικισμό είναι ο πόλεμο. ο προστατευτισμός είναι ο πορικό πόλεμο. Ε, και περί αυτού πρόκειται, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή επιβλήθηκαν σε πολλά προϊόντα δασμοί. Ο γεωργοδιατροφικό πανικό κλάδο έχει πληγεί τα μάλα, είναι όκτο σημαντικότερο στον κόσμο και έχουμε την περίπτωση με το κρασί, με τι ε, επιτραπέζιε ελιές και το λάδι, που είναι θύματα αυτών των δασμών. Δεν νομίζω ότι ο δρόμο ε, είναι περισσότερο πόλεμο και το λέω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ίσω η επιβολή δασμών δεν είναι η λύση. Η λύση είναι ο διάλογο. Πρέπει να βρεθεί λύση ε, μετά από διάλογο και συνεννόηση για να μην υπάρξει εμπορικό πόλεμο που θα μπορούσε με βάση το Ταφ να πλήξει μια ολόκληρη γενιά. Και σε ό,τι αφορά τι ενισχύσει τώρα, ζητώ ιδίω για τον τομέα του ίνου, ε, που είναι από του πλέον θηγέντε, ε, να υπάρξει αντιστάθμιση με ενισχύσει και να υπάρξει ένα σύστημα προώθηση των κρασιών. Ο εμπορικό πόλεμο, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι η λύση. Η λύση είναι ο διάλογο, η αντιστάθμιση, η αποζημίωση και η ενισχύση. Ευχαριστώ. Κυρία Μπιλμπά Παραντίκα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η καταλανική κρίση δεν έχει να κάνει με τη δημόσια τάξη. Υπάρχει πλήρη ε, απόρριψη τη βία ε, και δεν λύνονται τα προβλήματα με αποφάσει, ιδίω αν απειλείται το δικαίωμα τη διαδήλωση. Ε, ε, και της ασυλίας του Κοινοβουλίου. Εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό ζήτημα. Υπάρχει αδιέξοδο. Πρέπει να βρεθούν νέοι χώροι διαλόγου, εξέβρεση λύσεων. Στη δημοκρατία χωρίς νόμο τίποτα δεν είναι δυνατό. Που δεν μπορεί όμως ο νόμος ε, να είναι ένα εμπόδιο που θα ε, παρεμποδίσει τον διάλογο που πρέπει να υπάρξει. Και αυτό γίνεται τώρα. Ζητώ από την Ένωση να βοηθήσει να λυθεί η καταλληλική κρίση που είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα η Ευρώπη είναι ειδική στο να γεφυρώνει χάσματα και κρίσεις και πρέπει λοιπόν με διάλογο, με συνέστηση και με αμοιβαία αναγνώριση και με σθένος πολιτικό ε, να δράσουμε γιατί έτσι θα ε, μπορέσουμε να πετύχουμε μια μακροπρόθεσμη λύση στα προβλήματα και να μην κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καβατσίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, πολύ μιλάμε και πολλές ε, διαπραγματεύσεις γίνονται. Εγώ θέλω να μιλήσω ε, για την επισήμανση και των προϊόντων, ώστε να μην υπάρχει παιδική εργασία και να μην υπάρχει εκμετάλλευση. Ε, θα πρέπει να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Όλα τα προϊόντα ε, από την αρχή θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν προήλθαν από εκμετάλλευση από παιδική εργασία και από την αρχή θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν έχουν ρηπάνει το περιβάλλον ε, με τον τρόπο κατασκευής τους. Ε, δεν ε, μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Είμαστε στο 2019. Λίγα χρόνια μένουν αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και γι' αυτό τώρα χρειάζεται ένας νόμος που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα και θα καθιστά υποχρεωτικά αυτά τα πρότυπα. Θέλουμε να είμαστε ε, ένας ε, ηγέτης ε, στην αλυσίδα αξιών και να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτό το Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τοβαλιέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις 12 Οκτωβρίου ο ηγέτης του κόμματος, η ηγέτης του κόμματος για το μέλλον της Συρίας, Εύριν Καλάφ, σταυρώθηκε και το σώμα της ε, από τους ε, μοχθηρούς ε, δολοφόνους. Η ευρυνη είχε πτυχίο πολιτικού μηχανικού και είχε αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των γυναικείων δικαιωμάτων αλλά κυρίως στην ειρηνική συμβίωση μεταξύ Κούρδων, Σύριων, ε, και Σύριων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Ένα είδαλμα για το θάρρος, ε, το κουράγιο που ε, καταρρίφθηκε από το δολοφονικό φανατικό Ισλαμικό κράτος. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει και να παρακολουθεί αυτή την κατάσταση. Πρέπει να, να σταματήσει κάθε χρηματοδότηση προς την Άγκυρα, σταματήσουμε την γενοκτονία του κουρδικού λαού και την, ε, ε, τον εκμηδενισμό αυτού του στρατιωτικού σώματος που ήταν το μοναδικό το οποίο αγωνίστηκε κατά του Ισλαμικού κράτους και τον νίκησε. Είναι ένα στρατό στον οποίο αγωνίζονται πολλές γυναίκες και ήταν το μόνο χειρό κατά της ε, εισόδου του Ισλαμικού, της Ισλαμικής Τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. κυρία Σάιμπη. Όχι, δεν κάνουμε μπάνιο στις παραλίες Κώστα Μπράβο. Εδώ και πέντε μήνες δεν, έχουν, δεν έχετε δει, δεν έχουν δικαίωμα να συγκεντρωθούν. Για ποιον μιλάμε? Για, τις τρεις, για τους τρεις συναδέρφους από την Καταλωνία που δημοκρατικά εξελέγησαν όπως και όλοι εμείς στις 26 Μαΐου, αλλά που δεν μπόρεσαν να, βάλουν, να πατήσουν το πόδι τους στο ημικύκλιο αυτό. Γιατί τους κατηγορούνται, κατηγορούνται ότι οργάνωσαν ένα δημοψήφισμα. Δεν έκαναν κακό σε κανέναν, δημοψήφισμα οργάνωσαν. Η Καταλωνία αν είναι ανεξάρτητη ή όχι, ως Γαλλία δεν με αφορά. Το πρόβλημά μου είναι η χειραγώγηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς. Και αν θέτω το θέμα αυτό, σήμερα είναι ότι τίποτα δεν μας λέει ότι δεν θα είναι προηγούμενο και ότι αύριο κάποιος δεν θα υποφεληθεί να αποφασίσει ότι το α ή β μέλος της αντιπολίτευσης δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως σας το είπα και πάλι, δεν είναι θέμα να κρίνουμε την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Πρόκειται για την υπεράσπιση της πολιτικής ελευθερίας και της δημοκρατίας. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό θέμα και γι' αυτό δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Ρέσλερ. Κύριε Πρόεδρε, η ελευθερία της ε, μετακίνησης είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ένωσης. Για να μπορέσουν οι πολίτες Κροατίας να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλεονέκτημα, τα τελευταία δύο χρόνια η Κροατία φρόντισε να εφαρμόζεται πλήρως το κεκτημένο. Σήμερα πάνω από 6.500 ε, Κροάτες αστυνομικοί φυλάσσουν τα σύνορα και η ένταξη της Κροατίας στο Σέγγεν θα εξασφαλίσει την οικονομική συνεργασία αλλά και την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Αυτό λοιπόν συμφέρει όχι μόνο την Κροατία αλλά και όλα τα άλλα κράτη-μέλη και φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Είναι λοιπόν δίκαιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει για την τεχνική ετοιμότητα της Κροατίας ώστε να ενταχθεί στο Σέγγεν. Η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί αντικειμενικά. Πρέπει να απορριφθούν οι μη τεκμηριωμένες πολιτικές πιέσεις. Η Κροατία είναι έτοιμη για το Σέγγεν. Ο κύριος Ρούιθ Δεβέσα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Το μέλλον της Ευρώπης είναι το μεγάλο θέμα αυτής της θητείας για το Κοινοβούλιο χωρίς καμιά αμφιβολία. Πριν 10 χρόνια τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Και έκτοτε υπήρξαν διάφοροι μετασχηματισμοί και αλλαγές, ε, κάποια γεγονότα, το Brexit φυσικά, η κρίση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, οι επιπτώσεις ε, της οικονομικής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όλα αυτά μας ε, υποχρεώνει το να ξαναδούμε τις πολιτικές μας και τα θεσμικά όργανα και γι' αυτό Νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει για το μέλλον της Ευρώπης που θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ομοσπονδιακή πολιτική ένωση, δηλαδή πολιτική ένωση όπου δεν θα υπάρχουν εθνικά βέτο, ούτε αδιέξοδο στο Συμβούλιο και όπου το Κοινοβούλιο θα μπορεί να συναποφασίζει επίση όρει με το Συμβούλιο σε όλα τα ζητήματα. Άρα και στα θέματα τη φορολογία, των ιδίων πόρων και του πολιετού προεπολισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, στην πατρίδα μου τη Σλοβακία οι άνθρωποι μαθαίνουν φοβερά πράγματα για τις διαρροές, για τις επαφές μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος, της εισαγγελία των δικαστών Καθημερινά εμφανίζονται νέες ε, ταινίες και πληροφορίες σε σχέση με έρευνες για ε, τον, τη δολοφονία ενός νέου ε, δημοσιογράφου του Κούτσιακ και το πώς κανείς μπορεί να αγοράσει τη δικαιοσύνη. Επίσης, υπάρχουν μέλη της κυβέρνησης που καλύπτουν όλες αυτές τις δραστηριότητες και τα δικήματα. Αυτά τα μαθαίνουμε τους τελευταίους μήνες χάρη στο θάρρος των ε, ε, ε, δημοσιογράφων ερευνητών και της πίεσης της κοινωνίας μέσω διαδηλώσεων. Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος. Δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς στη Σλοβακία πρέπει να δώσουμε την μάχη για τη δικαιοσύνη και την δίκαιη κοινωνία. Όμως το θέμα της δικαιοσύνης σε ένα κράτος μέλος αφορά όλη την Ένωση γιατί αυτό φυσικά υπονομεύει την ε, εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Ε, αγαπητοί φίλοι, σαλάμ αλέκους. Αλλά δεν ξέρω πού βρίσκεστε ιδεολογικά. Δεν ξέρω πώς πήρατε την εξουσία ή για ποιο λόγο. Αν έχετε οποιαδήποτε επιρροή σημαίνει ότι η πολιτική στον 20ο αιώνα είναι υπέρ της κοινωνίας της ανθρωπότητας συλλογικά. Οπότε πρέπει να είμαι σαφής. Η κλιματική ε, δικαιοσύνη δεν υφίσταται χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Μιλάμε για τους φτωχούς, τους πιο ευάλωτους, οι οποίοι πληρώνουν τις καταστροφικές συνέπειες του κόσμου καθώς αυτός προχωρεί. Γι' αυτό χαίρομαι αυτούς που ταράζουν ε, τα νερά. Χαιρετίζω αυτούς που δεν πάνε σχολείο για να ε, φέρουν την προσοχή στο κλίμα. και επίση αποδεικνύεται ότι κανένας δεν είναι πολύ μικρός για να προκαλέσει αλλαγή. Κυρίως χαίρομαι αυτούς τους ανώνυμους ακτιβιστές που παλεύουν για τον τρόπο ζωής της απέναντι στην, ε, στα συμφέροντα. Πρέπει να έχουμε φωνές και δράσεις και να δράσουμε τώρα. Mr. Pardella. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτέλους τελειώνουν ε, τα πέντε χρόνια της Επιτροπής Juncker που ήταν καταστροφικές. Ε, καταστροφική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή Φοντερ φαίνεται να ακολουθεί στην ίδια γραμμή. Η σύγκρουση του Μακρόν τώρα με, τους, ε, με τα λόμπι των Αμερικανών άφησε να, να, μια αμφιβολία όσον αφορά την ανταξεκατησία του και η Επιτροπή Βαντερ προδιαγράφεται χειρότερη. Αφού συνεχίζει από τον σοσιαλισμό και, του και τους Περασμένη της θέλει να ε, ελέγξει όλα τα χαρτοφυλάκια από τη γερμανική σκοπιά. Δείχνει το πρόσωπο ενό μεγάλου μηχανισμού που είναι εξυπηρέτηση των γερμανικών αποκλειστικά συμφερόντων ενώ προσπαθεί να καλύψει, να αντιμετωπίσει την δίψα για δημοκρατία. Η κυρία Άντερσον. Την περασμένη εβδομάδα το, Ευρωπαϊ... Βρετανικό Δικαστήριο αποφάσισε κατά της ε, απόφασης που αφορούσε την Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και η νομοθεσία έγινε 21 χρόνια μετά την Συμφωνία. Είναι μια χώρα την οποία δεν μπορούμε να να ε, εμπιστευτούμε που ποτέ δεν τηρεί το λόγο της η κυρία Αλβιών. Πρέπει λοιπόν να μην συνενέσουμε στην ε, συμφωνία απόσυρσης γιατί το βρετανικό κατεστημένο θα ε, δουλέψει για να την υπονομεύσει σιγά σιγά. Όλοι χάσαμε από την περασμένη εβδομάδα ως με την αίμα η η ΕΜΑ έχει δικαίωμα την, ε, να υπερασπιστεί την Ιρλανδική ε, ε, υπηκότητα. Πρέπει να περάσει νομοθεσία η Βρετανία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ε, της Μεγάλης Παρασκευής. Ιδάλλως κάποιοι θα χάσουν την υπηκότητά τους. Αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε να συμβεί. Mrs. Κυρία Βόζεμπεργκ, Βριονίδη το 2015 η ελλάδα ανέλαβε το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού προβλήματος. η δήλωση ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας του 2016 δεκαέξι λειτουργήσε όμως εδώ και αρκετούς μήνες εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες έρχονται καθημερινά στα νησιά του βορειοανατολικού αιγαίου και η κατάσταση είναι εκρηκτική. τεράστιο συλλαλητήριο απόψε έγινε στη σάμο από απελπισμένους πολίτες. παράλληλα ο πρόεδρος ερντογάν εκβιάζει με νέε ανεξέλεγκτες ροές σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση η ελλάδα δυνατεί μόνη της να διαχειριστεί το πρόβλημα παρά τη μεταναστευτική πολιτική της νέας κυβέρνησης που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. δεν μπορούμε συνάδελφοι να προχωρήσουμε έτσι. πρέπει εδώ και τώρα να μοιραστούμε όλοι ανεξαιρέτως την ευθύνη του προβλήματος που είναι ευρωπαϊκό. οι χώρες που έχουν κλείσει τα σύνορά τους οφείλουν επειγόντως να δεχτούν τους πρόσφυγες που τους αναλογούν η λύση και η διαχείριση του θέματος επιβάλλεται να είναι άμεση αναλογική αλληλέγγυα αλλά κυρίως δίκαιη. σας ευχαριστώ. Mr. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2016 μετά το λεγόμενο πραξικόπημα, θα του έλεγα fake πραξικόπημα στην τουρκία τόνιζα από εδώ με αγωνία το εξή κάθε μέρα που περνάμε τον Ερτογάν στην εξουσία συσσωρεύεται το ανθρώπινο κόστος που θα καταβληθεί εντός και εκτός τουρκίας για απαλλαγή μα από αυτό το θηρίο. έκτοτε έγιναν πολλά φοβερά εντός τουρκίας και τώρα είμαστε ενώπιον ενός νέου εγκλήματο εναντίον των κούρδων. δεν είναι απλά θέμα προδοσία των συμμάχων μας ενάντια στη μάστιγα του ισλαμικού κράτου δεν είναι απλά θέματα ασφάλειας ή αξιοπιστίας. το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ενώπιόν μας τη Οθωμανική επεκτατική πολιτική που διαπράττει ο ερντογάν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. έχουμε λοιπόν ένα εγκληματία ο οποίος προαναγγέλει εθνικό ξεκαθάρισμα και παράνομη μετακίνηση πληθυσμών όπως ακριβώς επέβαλε το 1974 η τουρκία στην κύπρο και το έγκλημα συνεχίζεται. έφτασε η ώρα να οδηγήσουμε τον εγκληματία ενώπιον του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου στη χάγη. Mr. Davies. Κύριος Davies. Πρόεδρε, άκουσα την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιγράφεται στην, στη Βρετανία σαν αυτοκρατορία, ανεξέλεγκτη και, χωρίς, και αχαλήνοτη. Ε, ξέρω πως η, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά ε, ε, ελαττώματα, αλλά δεν είναι αυτοκρατορία σίγουρα. Ε, το ξέρω μετά από τόσα χρόνια θητείας εδώ. Είναι, μία, είναι ο πρωταθλητής της ευελευθερίας και της δημοκρατίας. Είναι απόδειξη ότι σε ένα κόσμο όπου οι υπερδυνάμεις μπορούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους στα μικρά έθνη, αλλά ε, εμείς αντιστεκόμαστε καλύτερα όλοι μαζί. Και βεβαίως ε, ενσωματώνει την πεποίθηση ότι δεν θα επαναληφθούν ποτέ οι συγκρούσεις του παρελθόντων. Η συμφωνία Brexit έχει επιτευχθεί στο Συμβούλιο και μεταξύ του Συμβουλίου και του Μπόρις Τζόνσον. Δικοί μου ψηφοφόροι δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία, δεν θέλουν καμιά συμφωνία. Θέλουν να μείνουν Ευρωπαίοι πολίτες και η Βρετανία να παίξει ηγετικό ρόλο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να φύγει. Ε, αν κερδίσουμε ή αν χάσουμε, ό,τι και αν γίνει, εμείς καλούμε τους συναδέλφους εδώ όλους να βασιστούν στην ε, ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σταθούν στο ύψος των προσδοκιών ώστε να λειτουργήσουν ως η δύναμη του καλού στον κόσμο. Η κυρία Σντάνοκα. Σήμερα το πρωί στη Ρήγα, ενώπιον της ε, Λιθωνικής Πρεσβείας, δείξαμε την αλληλεγγύη μας με το πολιτικό κρατούμενο Αλκίτουζας Παλέσκι, έναν από τους πιο γνωστούς ε, ε, πολέμιους του φασισμού, ε, πρώην μέλος του Κοινοβουλίου. Διώκεται για τις απόψεις του που αποκλίνουν από την επίσημη γραμμή όσον αφορά κάποια γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας της Λιθουανίας τον Ιανουάριο του 1991. Πολιτικοί κρατούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βαλτική θάλασσα είναι ε, ένας ε, πολύ γνωστός ε, αγωνιστής του Λιθανικού κράτους. Έχει συναντήσει τον Ραούλ Ραμέβα και τον Ζαλέσκι. Πολιτικοί κρατούμενοι λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνουν πώς πρέπει να γίνονται σεβαστές σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η απελευθέρωση αυτών των πολιτικών κρατουμένων θα ήταν μια καλή αρχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών. Κυρία Τσεκάρντι. In Στην Ιταλία, τα εθνικά μέσα μαζική ενημέρωση έδειξαν ότι η διάσκεψη κορυφή τη Μάλτα στις 23 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε ω ένα σημαντικό βήμα για τη λύση του θέματο των προσφύγων στην Ευρώπη. Τι απέγινε τίποτα. Ακόμα μια γελία σκηνοθεσία από είδαμε από όσα έγιναν από την τελευταία διασκέψη Κορφή των Υπουργών Εσωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ε, κατά τη γνώμη μου αυτό που μετρά δεν είναι το να κατανεμηθούν ξανά οι πρόσφυγε, αλλά να μην έρχονται. Η πολιτική του ε, μη χειροβέλτιστον δεν μπορεί να, δεν μπορεί να ισχύσει το να τους μοιράσουμε δίκαια σε όλες τις χώρες μπορεί να σημαίνει να μοιράσουμε δίκαια και άλλους θερμοκράτες. Στην Αφρική 1,5 δις ε, ζουν. Ε, πώς θα τους εμποδίσουμε να έρθουν στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το καθήκον να υπερασπιστεί τα σύνορά τη, το οφείλει στον πολιτισμό τη, στι χριστιανικέ τη ρίζε και στο σύστημα αξιών τη. Η διάσκεψη κορυφή της Μάλτας θα έχει, πρέπει να προσπαθήσει να βοηθήσει τις χώρες που έχουν πιο εκτεθειμένα σύνορα στα μεταναστά